Παρακαλώ καθίστε. Please. Παρακαλώ. Μπορείτε παρακαλώ να καθίσετε. Good afternoon everybody. Καλησπέρα σε όλους, καλώς ορίσατε. Φαντάζομαι ότι περισσότεροι από εσάς βρίσκεστε εδώ για την ακρόαση που αφορά την εμπορική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κεντρικής Αμερικής. Ευχαριστούμε που βρίσκεστε εδώ. Επιτρέψτε μου μόνο να αφιερώσουμε λίγα λεπτά σε κάτι που αποφασίσαμε σήμερα το πρωί να κάνουμε μια ψηφοφορία ηλεκτρονική χωρίς συζήτηση. Αποφασίσαμε σήμερα το πρωί ότι για να γνωρίζει ο εισηγητής τι πρέπει να κάνει, ε, σκόπιμο είναι να διεξαχθεί ψηφοφορία για το χωρί ψήφισμα, χωρί συζήτηση, χωρί τροπολογίες κατά πόσο αυτή η Επιτροπή θα ζητήσει από την Ολομέλεια του Κοινοβουλίου να παραπέμψει τη Συμφωνία Άκτα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτό αποφασίσαμε σήμερα το πρωί και αυτό πρόκειται να πράξουμε αυτήν εδώ τη στιγμή. Σας ζητώ και ξανά καμία συζήτηση, καμία παρέμβαση. Ναι, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ήθελα να γύρω ένα διαδικαστικό ε, θέμα. Κατά την άποψή μου, η διαδικασία ήταν λανθασμένη, Ζήτησα να μιλήσω πριν κλείσει η λίστα των ομιλητών. Μου αρνηθήκατε το δικαίωμα να μιλήσω. Ενώ στη συνέχεια ζητήσα, επιτρέψατε να μιλήσει ένα μέλος του ΕΛΚΑ, ξαναζήτησα να μιλήσω και πάλι δεν μου επιτρέπει να μιλήσω. Πιστεύω ότι όλα τα μέλη του παροντός κοινοβουλίου πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα να μιλήσουν και να πάρουν το λόγο όπως όλοι οι υπόλοιποι. δόθηκε ο λόγο στην ΚΟΕ όπως και σε όλες τις υπόλοιπες ομάδες που αποτελούν το παρόν κοινοβούλιο ειλικρινά. Κανένας δεν θα πιστέψει ότι είμαι προκατελημένο εναντί της ΚΟΕ. Ας προχωρήσουμε λοιπόν στην ψηφοφορία όπως συμφωνήθηκε άρχεται ε, η, ψηφοφορία συγγνώμη αφορά το κατά πόσο η παρούσα επιτροπή πιστεύει ότι εμείς ή κάποιος πρέπει να παραπέμψουμε να ζητήσουμε στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου επειδή αυτή η απόφαση θα πρέπει να ληφθεί από την Ολομέλεια το τι αποφασίζουμε εδώ είναι κατά πόσο θα ζητήσουμε από την Ολομέλεια να λάβει μια τέτοια απόφαση παραπομπής της άκτα στο δικαστήριο καμία συζήτηση, καμία τροπολογία ναι ή όχι επί της αρχής του κατά πόσο θα πρέπει να ζητήσουμε από την Ολομέλεια να ζητήσει από το δικαστήριο να αποφασίσει για τη συμβατότητα της συμφωνίας ΑΚΤΑ. Άρχεται η ψηφοφορία. Έχουμε μία επιπλέον ψήφο του ΕΛΚ. Μπορείτε να βγάλετε με από τις κάρτες σας παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με μεγάλη πλειοψηφία 5 υπέρ 21 κατά αποφασίσαμε λοιπόν στο εξή οποιοδήποτε θέλει μπορεί να επαναφέρει αυτό το ερώτημα Αυτό ήταν το μόνο πράγμα που με ανησυχούσε όσον αφορά τον εισηγητή. Αποφασίστηκε λοιπόν τώρα για το τι μπορείς να κάνεις αύριο. Μπορούμε να παραμείνουμε με το παρόν χρονοδιάγραμμα και να συνεχίσουμε με την διαδικασία ως έχει. Ευχαριστούμε λοιπόν πολύ. Τελειώσαμε λοιπόν με αυτό και ας περάσουμε στο σημείο 30. Έχουμε πολύ κόσμο εδώ πέρα στην αίθουσα. Are you ready now? Please. Are you ready now? Είμαστε έτοιμοι τώρα, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Vale.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 This is a hearing Έχουμε μία ακρόαση για τις ε, τυχές τις εμπορικές της συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κεντρικής Αμερικής. Όπως ξέρετε αυτή η συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κεντρικής Αμερικής συνήφθη και ολοκληρώθηκε το 2010. και μονογράφηκε το Μάρτιο φέτος. Έτσι λοιπόν, για να προετοιμάσουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ε, έκδοση της σύμφωνης γνώμης, η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, αρμόδια για το τμήμα που αφορά το εμπόριο της συμφωνίας αυτής, αποφάσισε να αναλάβει τα απαραίτητα μέτρα για να προετοιμαστεί και να εκπληρώσει το δικό της καθήκον. Έχουμε μια ομάδα παρακολούθησης για την Κεντρική Αμερική. Έχουμε ξεκινήσει συζητήσεις στην Επιτροπή μας. Σήμερα έχουμε ένα πολύ σημαντικό βήμα, στάδιο των διαδικασιών μας. Έχουμε οργανώσει ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα που ξεκινάει με την παρουσίαση από τον Επίτροπο Δεγκούχτ, τον οποίο και καλωσορίζω. Έχουμε εκπροσώπους κυβερνήσεων της Κεντρικής Αμερικής. Τους καλωσορίζω. Έχουμε επίσης μια σειρά προσκεκλημένων και βεβαίως και εν τέλει θα ακούσουμε τα μέλη της Επιτροπής μας και άλλους συναδέλφους του Κοινοβουλίου. Είναι πολύ σημαντική αυτή η χρονική στιγμή, όχι μόνο λόγω της σημασίας της ίδιας της ε, συμφωνίας, αλλά και λόγω των νέων αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα εμπορικά και ιδίω βέβαια του διεθνούς εμπορίου. Επίτροπε έχετε το λόγο θα κηρύξετε εσείς την έναρξη των εργασιών. Την Επιτροπή μας την γνωρίζετε καλά. Καθηγητά κύριε Μωρήρα, αξιότιμοι κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, κυρίε και κύριοι υπουργοί, πρεσβευτέ, κυρίε και κύριοι. Μπορεί από εδώ, από τις Βρυξέλλε, να φαίνονται πολύ μακρινές οι χώρε τη Κεντρικής Αμερική. αλλά για μένα εγώ έχω τη μεγάλη τιμή και ευτυχία να σας εξηγήσω γιατί δεν είναι τόσο μακρινέ ούτε και τόσο ασήμαντε. Έχει τεράστια σημασία αυτή η εμπορική συμφωνία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα μέλη τη, και πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή το χειρότερο δυνατόν. Για τρει λόγου. Καταρχά, γιατί υπάρχουν οικονομικά ωφέλη και για τι δύο πλευρέ. Έχουμε μια συμφωνία συνδέσεω με διάφορου ε, πυλώνε βεβαίω. Αλλά θα ήθελα να επισημάνω ότι ο κεντρικό πυλώνα είναι μια γενική και ευρεία συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, ένα ουσιώδες εργαλείο για την αντιμετώπιση μια σειρά προβλημάτων που έχει αντιμετωπίσει η Κεντρική Αμερική. Με τη διαπραγματεύση αυτή προκύπτουν νέε δυνατότητε επιχειρηματικέ για του εξαγωγεί και επενδυτέ από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τελωνιακή δασμή στην εισαγωγή βιομηχανικών προϊόντων και προϊόντων αλληλεία θα καταργηθούν. Θα έχουμε περίπου 90 δισεκατομμύρια ευρώ όγκο συναλλαγών. Επίσης, Προστατεύουμε ευαίσθητα και για τις δύο περιοχές προϊόντα με, ποσοστός, με την κατάργηση την αύξηση ποσοστώσεων ορισμένων γεωργικών προϊόντων. Ε, όπου δε αυτές καταργούνται δεν επιβάλλονται τελωνιακοί δασμοί. Εξαγωγές όπως το ουίσκι και ο ίνος από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν μηδανικό δασμό από τη θέση εφαρμογή της συμφωνίας. Η συμφωνία επίσης απλουστεύει τις τελωνιακές διαδικασίες οι χώρε τη Κεντρική Αμερική θα χρησιμοποιούν ενιαίο έντυπο για τα τελωνία του ύστερα από τρία χρόνια, πράγμα το οποίο θα ε, ε, μειώσει τον γραφειοκρατικό φόρτο όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για τι ε, χώρε τη περιοχή Κεντρική Αμερική και ιδιαίτερα μικρέ και μεσαίε επιχειρήσει. Οι εταίροι έχουν συμφωνήσει να καταργήσουν του φραγμού, τι επενδύσει και τι εισαγωγέ και έτσι γίνονται πιο ελκυστικές οι χώρες αυτές για επενδύσεις, ιδιαίτερα στον χώρο των ε, χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, των θαλάσσιων μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών. Οι συνθήκες που θα ισχύουν θα είναι για την Ευρωπαϊκή Ένωση ίδιες με, αυτούς που ισχύουν, με αυτές που ισχύουν για άλλους ε, ανταγωνιστές, δεδομένου δε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείες ε, ήδη έχουν συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με την περιφέρεια αυτή, βλέπετε πόσο σημαντική θα είναι η συμφωνία συμφωνίες για το εμπόριο, τις δημόσιες προμήθειες, την πνευματική ιδιοκτησία, ε, τοπικά προϊόντα όπως ο το και ε, η μπύρα της Βαβαρίας ή η γκράπα της Ιταλίας περιλαμβάνονται σε αυτή τη συμφωνία, όπως βλέπετε είναι ευρύτατη. Ταυτόχρονα όμως είναι και πολύ ισορροπημένη η συμφωνία, διότι έχουμε διαπραγματευτεί σε διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξη με την ανάπτυξη των εταίρων μας από την Κεντρική Αμερική ως κύριο στόχο. Συμβάλλουμε, πιστεύω, ως εκ τούτου στην ε, ανάπτυξη περιοχής, βελτιώνοντας τις συνθήκες ε, εργασίας των, των ε, επιχειρήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα έχουμε το σύστημα των γενικευμένων προτιμήσεων ως κύριο σύστημα από το οποίο λειτουργούν οι εισαγωγές και εξαγωγές. Αυτό αντικαθίσταται, κλειστά, δηλαδή ένα μονομε... με τη νέα συμφωνία ένα σύστημα μονομερές με ένα σύστημα πολύ πιο πολύπλευρο και πιο ωφέλιμο για τις ε, επιχειρήσεις. Βελτιώνεται η πρόσβαση στην αγορά των κρατών της Κεντρικής Αμερικής σε μια αγορά 540 εκατομμυρίων πολιτών και βελτιώνεται και η αξία των ε, οικονομικών συναλλαγών. Φερρυπίν ε, βελτιώνονται οι συνθήκες απασχόληση για πάρα πολλού εργαζομένους ε, από το Σαλβαδόρ, την Ονδούρα και πολλές άλλες χώρες. Αναμένεται η απελευθέρωση και στο χώρο της γεωργίας να προσφέρει καλά αποτελέσματα. Ήδη έχουμε μελέτες οι οποίες αποδεικνύουν ότι οι εξαγωγέ ε, οπόρων και ξηρών καρπών μπορεί να δώσουν πολύ καλά αποτελέσματα με συγκεκριμένα πολύ σημαντικές, ε, σημαντικά κέρδη στα γενικότερο εισόδημα των πρωτών αυτών που αναμένεται να αυξηθεί κατά 2,5 τουλάχιστον δισεκατομμύρια ευρώ συνολικά. Επίσης το ΕΠ θα αυξηθεί μεν, αλλά ιδιαίτερα μπορεί να φτάσει από 0,5% σε 3-3,5% αύξηση το συνολικό ΑΕΠ με σημαντικά και έμεσα ωφέλη, όπως η αύξηση των εξαγωγών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα σημάνει λιγότερη εξάρτηση των κρατών της Κεντρικής Αμερικής από τις εξαγωγές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, άρα μεγαλύτερη αντοχή στις δύσκολες εποχές και περισσότερη ανάπτυξη στις καλές εποχές. Άρα και οι δύο πλευρές κερδίζουν από την κύρωση της συμφωνίας. Αυτός ήταν ο πρώτος λόγος. Ο δεύτερος λόγος είναι μια ε, πρόοδος προς τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η συμφωνία δηλαδή δεσμεύει και τις δύο πλευρές να σεβαστούν, να εφαρμόσουν και να υλοποιήσουν μια σειρά από παγκόσμιου χαρακτήρα, οικουμενικού χαρακτήρα προδιαγραφές για το περιβάλλον, ε, κοινέ ε, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κεντρικής Αμερικής, μας δεσμεύει λοιπόν όλους το κείμενο να διαφυλάξουμε αυτές τις προδιαγραφές και ιδιαίτερα δεσμεύονται τα συμβαλόμενα μέρη να, έχουν, να διατηρήσουν υψηλό επίπεδο προστασία του εργατικού δυναμικού και του περιβάλλοντο και να μην, το να τι προδιαγραφέ αυτέ προκειμένου να ενισχύσουν το εμποριό του και ιδιαίτερα θα στηριχθούν και θα τηρηθούν οι ε, συμφωνίε, οι βασικέ ε, αρχέ των διεθνών συμφωνιών και συμβάσεων εμπορίου. Αυτά συνοδεύονται και από μια διαδικασία διαιτησίας. Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι δεν είναι αρκετά ε, αρκετά ισχυρός αυτός ο μηχανισμός, αλλά αυτό είναι σφάλμα, διότι καταρχάς μπορεί μονομερός να τεθεί σε λειτουργία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από μια χώρα της Κεντρικής Αμερικής η διαδικασία της ακόμη και με την ακόμη και παρά την αντίδραση του άλλου εμπλεκόμενου μέρους. Επίσης, διότι επιτρέπει ανεξάρτητη και αμερόληπτοι ειδικοί να κρίνουν μια υπόθεση και επίσης διότι οι αποφάσεις θα δημοσιοποιούνται και ως εκ τούτου θα ε, εξασφαλίσετε η απαραίτητη πίεση ε, για την ουσιαστική υλοποίηση των αποφάσεων της διατησίας. Η κοινωνία των πολιτών διατηρεί την πίεσή της, διατηρεί την πίεση και λογοδοσία προς εμάς, προς τις κυβερνήσεις. Ανοιχτές συνεδριάσεις των εκπροσώπων των κυβερνήσεων με προσώπους από, από το χώρο των μη κυβερνητικών οργανώσεων, όπου θα εκτίθενται όλα τα ζητήματα των συμφωνιών, όπου θα λαμβάνονται αποφάσεις δυνάμει και των συστάσεων της κοινωνία των πολιτών. Πάλι θα γίνονται δημόσια. Θα έχουμε επίσης ε, ρήτρα ανθρωπινών δικαιωμάτων, την ίδια αυτή πάγια και πολύ ισχυρή ρήτρα ανθρωπινών δικαιωμάτων που ε, ακολουθούμε παγίω στην πολιτική μας ε, με τρίτα κράτη, όπως ορίστε και στην συνθήκη της Λισαβόνας και ω εκ τούτου στηρίζουμε την προστασία της δημοκρατίας, του Κράτου δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των αρχών του διεθνού δικαίου. Η συμφωνία αυτή δεν αποτελεί λοιπόν εξαίρεση ως προς το στοιχείο αυτό. Και προσδιορίζει όρους για, ε, για το σεβασμό των ανθρωπινων αρχών, των κανόνων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όσο στοιχείο μπορεί να προβληθεί και σε δικαστήρια. Και στην πράξη αυτό σημαίνει ότι όταν μια κυβέρνηση παραβιάσει ενδεχομένω μια από αυτέ τι βασικέ αρχέ, η οδήποτε εκ των συμβαλωμένων μερών θα μπορεί και μόνο μερό ακόμη να αναλάβει μέτρα αναλογικά, τα οποία μπορεί να φτάσουν μέχρι και άρση τη ε, αναστολή μάλλον τη συμφωνία. Αυτή είναι η πολύ σημαντική δράση που μπορεί να προβλέψει μια συμφωνία όπω η παρούσα και σα διαβεβαιώ ότι εγώ τουλάχιστον από πλευρά μου θα αναλάβω κάθε μέτρο υπό την ευθύνη μου για να την υλοποιήσω ουσιαστικά. Όμω το πιο σημαντικό στοιχείο τη συμφωνία στον τομέα αυτών είναι νομίζω η Ευρώπη, η διαδικασία μέσα από την οποία ε, μια επιτροπή κοινοβουλευτικών, ε, μελών δηλαδή των κοινοβουλίων, των κρατών της Κεντρικής Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα ε, συστήσει, θα συσταθεί και θα μπορεί να ζητεί πληροφορίες, στοιχεία για κάθε κομμάτι συμφωνίας εμπορικής μεταξύ των δύο πλευρών. Έτσι λοιπόν, όχι μόνο βιώσιμη ανάπτυξη και ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά κάθε πτυχή μια τέτοια συμφωνία εμπορική θα μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εξέταση από την Εν Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Αυτή είναι η λόγη και αυτό είναι ο τρίτο και πιο σημαντικό λόγο να υποστηρίξουμε αυτή την συμφωνία. Στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού εγχειρήματο γνωρίζετε ότι ε, βρίσκεται ε, θεμελιωμένη η αρχή ότι πρέπει να ξεπεράσουμε την ε, στενόμυαλη προσέγγιση των εθνικών συμφερόντων και να προχωρήσουμε σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο, ενωμένοι για να αντιμετωπίσουμε τι προκλήσεις του σήμερα. Σεβόμαστε τους κεντροαμερικανού εταίρους μας. Πρέπει να υπογραμμίσουμε ιδιαίτερα ότι αυτή η περιφέρεια έχει επί πολλέ δεκαετίες αγωνιστεί σκληρά για να προχωρήσει προς περισσότερη ολοκλήρωση και όχι μόνο πολιτικά αλλά και οικονομικά. Με αυτό λοιπόν το κοινό περιφερειακό όραμα μπόρεσε να προχωρήσει στη διαπραγμάτευση και ε, σύναψη αυτής της πολύ σημαντικής και ε, ευρείας συμφωνίας. Μια συμφωνίας η οποία προχωρεί και πέραν αυτών, πέραν αυτών διότι για πρώτη φορά έχουμε δεσμευτικές υποχρεώσεις για εσωτερικές ε, σχέσεις, δηλαδή άπαξ και τεθεί σε ισχύει αυτή η συμφωνία, η Κεντρική Αμερική θα προχωρήσει προ κοινέ τεχνολογικέ προδιαγραφέ για τα αγαθά και τι υπηρεσίε. Θα υπάρξουν κοινοί κανόνε για γεωργικά προϊόντα όπω τα γαλακτοκομικά και το καταργασμένο ξύλο και τα καταργασμένα αγαθά και από τη στιγμή που θα, μπο... θα συναυθεί η συμφωνία θα μπορεί ένα ευρωπαϊκό προϊόν που έχει εξαχθεί σε μια χώρα της Κεντρικής Αμερικής να πολιθεί σε μια άλλη χωρί επιπλέον δασμούς. Άρα λοιπόν θα απορρέουν από αυτή τη συμφωνία πολύ σημαντικά ωφέλη για τις δύο πλευρές. Ιδιαίτερα σημαντικό όμως είναι ότι η οικονομική αυτή ολοκλήρωση θα αποτελέσει και βασικό πυλώνα τη πολιτική ολοκλήρωση στην περιφέρεια τη Κεντρική Αμερική. Η συμφωνία αυτή, κυρίε και κύριοι, αποτελεί κομμάτι μια γενικότερη στρατηγική για να προχωρήσουμε προ την οικονομική ανάπτυξη. Μπορεί η Κεντρική Αμερική να μην είναι ο μεγαλύτερο των εμπορικών μα εταίρων, όμως έχει, ο εταίρων όμω έχει πάρα πολύ σημαντικά και απτά ωφέλη αυτή η συμφωνία να προσφέρει και για τι δύο πλευρέ και καθώ περνούμε από μια εποχή κρίση, πρέπει να προχωρήσουμε αποφασιστικά σε κάθε μέτωπο. Προχωρούμε σε μέτρα απελευθέρωση με όλη την Λατινική Αμερική και το χώρο της Καραϊβικής. Είχαμε την συμφωνία του 99 που όμως εντωμεταξύ έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία σήμερα προσλάβει και πάνω απ' όλα πρέπει να ε, μπορέσουμε να κάνουμε πρόοδο επί τη βάση των σημαντικών ιδεών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της βιώσιμης ανάπτυξης και της περιφερειακής ολοκλήρωσης. Μπορεί κανείς να προβάλλει το επιχείρημα ότι λόγω αυτών των στοιχείων ή εν λόγω συμφωνία δεν αφορά τόσο το εμπόριο όσο την εξωτερική πολιτική. Για μένα όμως τέτοιες διακρίσεις δεν έχουν μεγάλη αξία. ιδιαίτερη αξία έχει το αποτέλεσμα που θα προκύψει από αυτή τη συμφωνία. Αποτέλεσμα οικονομικό, αποτέλεσμα πολιτικό, λόγος δηλαδή να προχωρήσουμε στο δυνατόν πιο γρήγορα, όπως ελπίζω ότι θα πράξουμε. Σας ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Πρώτος εκ των προσκεκλημένων μας από την Κεντρική Αμερική είναι ο Υφυπουργό Βιομηχανίας και Εμπορίου της Ονδούρας, κύριος Μέλβιν Ρεντόντο. Υφυπουργό Βιομηχανίας και Εμπορίου της Ονδούρας. Και προσωρινός ε, πρόεδρος που έχει μάλλον την προσωρινή προεδρία της ε, ΣΥΚΑ, του συστήματος δηλαδή ολοκλήρωσης της Κεντρικής Αμερικής. Παρακαλώ να λάβετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, Βιτάλικο Μορέιρα, Πρόεδρε της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού, κύριε Επίτροπε Ντεγκούχτ. Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι μέλη της Επιτροπής, επισκέπτες, φίλοι όλοι μας. Με μεγάλη ευχαρίστηση σας απευθύνω το λόγο ως προεδρεύων του συστήματος ε, της κεντροαμερικανικής ενσωμάτωσης για να παρουσιάσουμε τη δική μας ε, άποψη και το όραμά μας στα πλαίσια του εμπορίου, στα πλαίσια αυτής της ε, συμφωνίας της Συμφωνίας μεταξύ Νοτιομήρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρούμε ότι η συμφωνία αυτή είναι η φυσική εξέλιξη των σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κεντρικής Αμερικής διαδικασία που άρχισε την δεκαετία του 80 μέσω του διαλόγου του Σαν Χωσέ σε πολιτικά πλαίσια. Συνεχίστηκε ο διάλογος αυτός από την Συμφωνία Πολιτικού Διαλόγου και Συνεργασίας του 2003 και το Σύστημα Γενικευμένων Προτιμήσεως συν τα εμπορικά σχέδια πρόσφατα. Αυτή η συμφωνία είναι πάρα πολύ σημαντική και είναι το καταδεικνύει το στάδιο οριμότητας των σχέσεων μεταξύ των δύο περιοχών μας. Όσον αφορά την πραγματικότητα, την σημερινή, είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε κάποιες αριθμούς οι οποίοι αφορούν το διαπεριφερειακό ε, εμπόριο με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσουμε να δούμε με συγκεκριμένο τρόπο ποια είναι τα ωφέλη τα οποία θα μπορέσουν να αποκομίσουν τα δύο μέρη όταν θα τεθεί πλήρως σε ισχύ η συμφωνία αυτή. Το 2010 το διαπεριφερειακό εμπόριο ανήλθε σε περισσότερα από 11 δις δολάρια με σταθερό ποσοστό ανάπτυξης 8,34% στην ε, πενταετία 2005-2010. Και οι εμπορικές διαπεριφερειακές σχέσεις ήταν οι δεύτερες πιο σημαντικές όσον αφορά τις συναλλαγές ανά τον κόσμο. Εξάλλου, οι συναλλαγές μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή την ε, περιοχή είναι εξαιρετικά ε, καλές. Ο τρίτος εμπορικός μας εταίρος είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση με ποσοστό περισσότερο από 13% σε εξαγωγές και 6,7% σε εισαγωγές. Με αυτές τις λεπτομέρειες είναι προφανές για όλους ότι αυτή η συμφωνία είναι η πιο ε, σωστή σχέση για να μπορέσουμε να μπορέσουμε να κάνουμε τις χεμπορικές μας σχέσεις καλύτερες μεταξύ των δύο εταίρων, πράγμα το οποίο θα είναι εποφελές και για τους δύο. Πράγμα που σημαίνει ότι όχι μόνο θα μπορέσουμε να έχουμε εμείς στη διάθεσή μας ε, ένα ε, σύνολο 500 εκατομμυρίων ατόμων, αλλά και κυρίως ε, τον, ε, την Ήπειρο με, το, με τη μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη. Επίσης, θα ήθελα να σας εξηγήσω τι σημαίνει από εμπορικής πλευράς αυτή η συμφωνία. Σημαίνει δημιουργία και βελτίωση και αύξηση των δυνατοτήτων σε εμπορικό επίπεδο που σημαίνει ότι υπάρχει πρόσβαση στις αγορές και των δύο μερών, σημαίνει παροχή υπηρεσιών, ηλεκτρονικό εμπόριο, ε, σωστούς κανόνες σε τον ε, τομέα των επενδύσεων, σωστούς κανόνες και πρόσβαση στις ε, αγορές κρατικών ε, προμηθειών συγκεκριμένους κανόνες σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας κτλ. Συγκεκριμένα, ό,τι μέρο μέτρα λάβουμε θα βοηθήσουν ώστε να μπορέσει το διαπεριφερειακό εμπόριο να βελτιθεί και να υπάρξουν και άλλες δεσμεύσεις όσον αφορά την πρόσβαση στις αγορές. Πράγμα που σημαίνει ότι προφανώς η Συμφωνία Σύνδεσης στην εμπορική της διάσταση θα έχει επιπτώσεις σημαντικότατες όσον αφορά την ε, οικονομική ενσωμάτωση της Κεντρικής Αμερικής. Όλα αυτά συμπληρώνονται από την ε, σαφή δέσμευση να προωθήσουμε την ανάπτυξη του εμπορίου μεταξύ των δύο περιοχών μας με τρόπο ώστε να καταλήξουμε σε υφόρο ανάπτυξη για την οποία, πράγμα τα οποία συμπεριλαμβάνονται οι δεσμεύσεις της Ατζέντα 21 για την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη το σχέδιο εφαρμογής του Johannesburg για την ανάπτυξη και η υπουργική δήλωση του ΕΚΟΣΟΚ για την πλήρη απασχόληση και τις ε, σωστές ε, συνθήκες ε, εργασίας, καλή διακυβέρνηση, διαφάνεια, καταπολέμηση της διαφθοράς, μεταξύ άλλων, δεδομένου ότι πρόκειται για δεσμεύσεις οι οποίες έχουν αναλυφθεί για να υπάρξει αμοιβαία, να υπάρξουν αμοιβαία ωφέλη από αυτή την ε, συμφωνία. Επίσης, θα ήθελα να τονίσω ότι πρόκειται για ένα από τα χαρακτηριστικά που με τον καλύτερο τρόπο ορίζονται σε αυτή τη συμφωνία. Δεδομένου ότι είναι το πρώτο το οποίο προσυπογράφει η Κεντρική Αμερική στα πλαίσια μιας ε, διαπεριφερειακής συμφωνίας. Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα οποία προανέφερα, οι οικονομικές και εμπορικές προοπτικές ε, της Συμφωνίας Σύνδεσης δεν μπορούν να είναι παρά οι καλύτερες προϋποθέσεις για την ε, ευκαιρίες που παρουσιάζουν, διότι θεσπίζουν εμπορικούς κανόνες τελευταίας γενιάς και εγγυώνται τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητά τους. Η επέκταση επίσης της αγοράς αυτής μέσω της ενσωμάτωσης και του Παναμά στην ε, ε, ενσωμάτωση της ε, την οικονομική της Κεντρικής Αμερικής και την αηφόρο ανάπτυξη, λαμβάνοντας υπόψη της ανημετρίας, είναι από τα κλειδιά που θα μας επιτρέψουν να κάνουμε μια επιτυχή συμφωνία. Συνειδητοποιούμε το γεγονός ότι στο εσωτερικό της περιοχής Κεντρικής Αμερικής η επιτυχία αυτής της συμφωνίας περνά από τις κατάλληλες δράσεις της καλής διακυβέρνησης, από την ε, υιοθέτηση μέτρων που θα προορίσουν την ε, σταθερότητα, την ισότητα και την δικαιοσύνη όσον αφορά τον επιμερισμό των ε, κερδών αυτής της συμφωνίας θα μας βοηθήσουν να καταπολεμήσουμε την διαφθορά, την ατιμορρησία και την βία και θα μας βοηθήσουν να έχουμε καλύτερη οικονομική και κοινωνική συνοχή μεταξύ άλλων. Κύριοι μέλη και κυρίες μέλη της ΙΝΤΑ, κύριοι και κυρίες μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, φίλοι που μας ε, συνοδεύετε σήμερα, είναι σαφές ότι η Κεντρική Αμερική και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπόρεσαν να διαπραγματευτούν μία συμφωνία αμοιβαίων ωφελών, τα οποία καθορίζονται με σαφήνεια και αποδεικνύουν το ότι έχουν οριμάσει οι σχέσεις συνεργασίας και οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ μας και θα μπορέσουν να δώσουν νέες δυνατότητες ε, ανάπτυξης στους διάφορους, ε, στα διάφορα στρώματα της κοινωνίας μας και θα βοηθήσουν να αναπτυχθούν μηχανισμοί που θα βελτιώσουν, θα τελειοποιήσουν αυτή τη συμφωνία και θα μπορέσουν να την προσαρμόσουν στις αναδυόμενες νέες προκλήσεις. Αυτή η συμφωνία, μεταξύ άλλων, δίδει νέες ευκαιρίες, ευκαιρίες για να μπορέσουν να δημιουργηθούν καλύτερες θέσεις απασχόλησης που θα βοηθήσουν το, το εμπόριο και τις επενδυτικέ ροέ. Τελειώνοντα, θα ήθελα να σα ευχαριστήσω και εσέ, κύριε Μορέιρα, για την πρόσκληση που μα κάνατε να έρθουμε να σα εξηγήσουμε την δική μα άποψη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Ντεκούχτ για την εξαιρετική παρουσίασή του και όλου τους εισηγητέ που θα μιλήσουν μετά από μένα και θα μπορέσουν με τις διευκρινήσει που θα δώσουν να εμπλωτίσουν την ανάλυση αυτή τη συμφωνία. Σα ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σα δώσαμε τον λόγο καταρχά επειδή είστε και προσωρινό πρόεδρο ε, του ΣΥΚΑ, του συστήματο, είπαμε τη Κεντρική Αμερική. Ακούσαμε τι απόψει και τώρα μπορούμε να περάσουμε στου ομιλητές από τι διάφορε χώρε Κεντρική Αμερική, εξ τη. Ε, Γουατεμάλας ε, θα λάβει το λόγο ο, μάλλον η Υφυπουργός, κυρία Φλόρες, για θέματα βιομηχανίας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, εξ ονόματος της κυβέρνησης της Γουατεμάλας και του Υπουργού Οικονομικών ε, Σέρχιο Ντελατόρε θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που μας δίνεται να μιλήσουμε εδώ στην Επιτροπή σας για τη σημασία που έχει για τη χώρα μας η Συμφωνία Σύνδεσης. Η Συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ Κεντρικής Αμερικής και Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μοναδική ως προς την φύση της και σηματοδοτεί ένα ιστορικό γεγονός για το εξωτερικό εμπόριο, διότι θεσπίζει μια συμμαχία μεταξύ των δύο περιοχών που θα εγγυηθεί την ε, ύπαρξη και την, ε, το σεβασμό της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της πρόθεσης της βιώσιμης ανάπτυξης. Πρόκειται για δεσμεύσεις τις οποίες ε, έχουμε αναλάβει και συγκεκριμένα η κυβέρνηση του Προέδρου Ότο Πέρεθ Μολίνας ό,τι αφορά την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη σε ένα πλαίσιο ολοκλήρωσης ε, στο οποίο συμμετέχουμε όλοι κάτοικοι της Γουατεμάλας. Η Συμφωνία Σύνθεσης είναι ένα μέσο το οποίο θα βοηθήσει στην ενίσχυση του περιφερειακού, των περιφερειακών θεσμών. Η Επιτροπή σύνδεση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. και συμμετέχει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Κεντροαμερικανική Βουλή. Αλλά και η κοινή συμβουλευτική επιτροπή θα εγγυηθούν την πλήρη συμμετοχή και τη κοινωνία των πολιτών στην υλοποίηση και διαχείριση τη συμφωνία. Η συμφωνία αυτή επίση παγιώνει τις εμπορικές μας σχέσεις ε, και τις ε, παρέχει ασφάλεια δικαίου με έναν ε, αποτελεσματικό μηχανισμό επίλυσης διαφορών που είναι δίκαιος, που είναι προβλέψιμος και επίσης δίνει και κάποια μέτρα εμπορικής άμυνας και ασφαλιστικές δικλείδες, ώστε να μπορούν και οι επιχειρηματίες από τις δύο πλευρές να προγραμματίζουν και να πραγματοποιούν μακροχρόνιες επενδύσεις και να προωθούν τις εμπορικές ανταλλαγές. Πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε έτσι να προωθήσουμε και τι εξαγωγέ μα. Επίση η συμφωνία προστατεύει και τι γεωγραφικέ ενδείξει. Η Γουατεμάλα προσαρμόζει την εσωτερική τη νομοθεσία ό,τι αφορά τα δικαιώματα πραγματική ιδιοκτησία, ώστε να φτάσουν τα διεθνή πρότυπα προστασία. διευκολύνοντα και τη διαδικασία εγγραφή των ε, ξένων γεωγραφικών ενδείξεων. Η κυβέρνησή μας ανέλαβε καθήκοντα το Γενάρη φέτος και θέλω να σας πω ότι μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η συμφωνία αυτή. Η δημοκρατικά εκλεχθήσα κυβέρνηση του Προέδρου το Πέρεθ έλαβε πλέον τα ενία της χώρας και σημαντικές προσπάθειες πραγματοποιεί, ούτως ώστε να υπάρξει διαφάνεια και να δοθούν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Τρεις είναι οι, βασικά, τρίτα βασικά σύμφωνα στα οποία τονίζουμε, στα οποία αφιερώνουμε τις προσπάθειές μας. Πρώτα απ' όλα, ε, το σύμφωνο για μηδέν φτώχεια. Θέλουμε να, ε, μάλλον πείνα, για να μην υπάρχει πρόβλημα υποσυτισμού. Επίσης φορολογικό σύμφωνο, να έχουμε δηλαδή τους απαραίτητους σπόρους για να μπορέσουμε να εγγυηθούμε την ευημερία των κατοίκων της Γουατεμάλας. Στους δύο πρώτους μήνες της, διακυβέρνηση ε, της διακυβέρνησης της χώρας ολοκληρώσαμε την φορολογική μεταρρύθμιση. Επίσης έχουμε το Σύμφωνο Ασφάλειας και Δικαιοσύνης για την καταπολέμηση του φαινομένου της ατιμορρησίας η δέσμευση της κυβέρνησης του Προέδρου, του Προέδρου Πέρεθ Μολίνα ε, για την αλλαγή και την κοινωνική συμφιλίωση είναι πάρα πολύ σημαντική. Έχει προσυπογράψει τις ειρηνευτικές συμφωνίες ε, και από τότε που ανέλευτα τα καθήκοντά του ασκεί την ε, εντολή του για να διορθώσει κάποιες καθυστερήσεις στην υλοποίηση των συμφωνιών αυτών, για να καταπολεμήσει τις αδικίες, να αποκαταστήσει τον κοινωνικό ιστό και για να δώσει ε, τους απαραίτητους πόρους επενδύοντας ε, στο σημαντικό στοιχείο της χώρας μας που είναι οι ίδιοι οι κάτοικοι. Θέλουμε να έχουμε μια κοινωνία όπου θα κυριαρχεί η παιδεία της ειρήνης, όπου θα είναι σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα έχουμε κράτος δικαίου, σεβασμό της νομοθεσίας. Θέλουμε να υπάρχει δικαιοσύνη, θέλουμε να διώκονται όσοι διαπράττουν ε, αδικήματα κατά των εργαζομένων. Υπάρχει λοιπόν πολυτομεακή, πολυκλαδική συνεργασία. Έχουμε το ε, Υπουργείο Διακυβέρνηση ε, Εξωτερικών Σχέσεων, Εργασία, Δημόσια Διοίκηση, Φορολογικέ Υπηρεσίε που συνεργάζονται. Επίση, στον οικονομικό τομέα, η κυβέρνηση τη Γουατεμάλα έχει ξεκινήσει μία πλήρη πολιτική ε, συλλογή επενδύσεων για την ανάπτυξη της ε, χώρας και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι για να γίνει οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα η κυβέρνηση της Γουατεμάλας προ... Ε, δίνει μεγάλη σημασία στην προστασία του περιβάλλοντος, στην αξιοπρεπή εργασία και τα δικαιώματα των αυτόχθονων πληθυσμών. Όλα αυτά σας τα λέω για να σας δείξουμε ε, πόσο μεγάλη σημασία αποδίδουμε σε αυτή τη συμφωνία. Ευχαριστώ. Very much. Next, uh, on behalf of uh, Nicaragua, the Minister... Ο κύριος Ορλάντος Ολοθάνο, Υπουργός Εμπορίου της Νικαράγουα. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρο της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Βιτάλ Μορέιρα. Κύριε Επίτροπη Καρλ Ντεγούχ. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Υπουργοί, υφυπουργοί και πρέσβεις των κρατών της Κεντρικής Αμερικής. Κυρίες και κύριοι, αρχίζοντας θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μου δίνετε τη δυνατότητα να σας απευθύνω το λόγο και να σας επευθύνω χαιρετισμό εκ μέρους του Πρόεδρου του Νικαράγου, του Πρόεδρου Ντανιέλ Ορτέγα. Λέγομαι Ορλάντο Δελγαδίγιο και είμαι Υπουργό Ανάπτυξης, Συνεργασίας και Εμπορίου της Νικαράγουα. Θέλουμε να υποστηρίξουμε την ε, ενσωμάτωση της Κεντρικής Αμερικής σε θεσμικό, εμπορικό, κοινωνικό πλαίσιο, καθώς και την Συμφωνία Σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για μια ιστορική σημασία συμφωνία. Όχι μόνο διότι ε, αφορά δύο περιοχές και διότι προωθεί την δική μας περιοχή της Κεντρικής Αμερικής, αλλά διότι και εμείς και εσείς προσπαθούμε να οικοδομήσουμε τις σχέσεις αυτής εδώ και 30 χρόνια. Από την εποχή του διαλόγου του Σαν Χωζέ και της συμφωνίας του Λουξεμβούργου που υπεγράφει το 1985 και απετέλεσε την πρώτη συμφωνία μεταξύ περιοχής και περιοχής που παγιώνεται τώρα με τη Συμφωνία Σύνδεσης. Πρόκειται για μια συμφωνία στην οποία πολλά θα φέρουν και τα δύο μέρη. Αφενός τεχνολογία, κεφάλαιο και απ' την άλλη στρατηγική θέση για το διεθνές εμπόριο, δυνατότητες ε, επενδύσεων και πάρα πολλές ε, δυνατότητες που αφορούν την εκμετάλλευση της γης και την ε, παραγωγή. Πράγμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό σε περίοδο κρίσεως. Για την Ικαράγουα πρέπει να πω ότι σε στενή συνεργασία μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα μικρών μεσαίων επιχειρήσεων και εργαζομένων καθώς και με την ε, Εθνική Συμμαχία των Τριών ε, Τομέων έγινε η διαπραγμάτευση. Πρόκειται λοιπόν για μια πάρα πολύ πολύτιμη συμφωνία η οποία εμπλουτίστηκε ε, εκ των υστέρων και θα βοηθήσει την ανάπτυξη των κρατών της Κεντρικής Αμερικής. Αυτό θα το βοηθήσει και το ε, ταμείο που αφορά την αηφόρο ανάπτυξη με την ε, κοινωνική διάσταση του θέματος και με την προστασία του περιβάλλοντος, κυρίως την προστασία των υδάτικων πόρων, ώστε να μπορέσουμε να αμβλύνουμε τις διάφορες διαφορές που υπάρχουν σε περιφερειακό επίπεδο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην αφαιθεί στην τύχη του η συμφωνία αυτή. Θα πρέπει να την υποστηρίξουμε, να τη συνοδεύσουμε οι κυβερνήσεις, τα κοινοβούλια, όλοι οι επιχειρηματίες, μικροί και μεγάλοι, ακόμη και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι εργαζόμενοι, οι συνεταιρισμοί καθώς και όλες οι οργανώσεις ώστε να μπορέσει να γίνει ένα πραγματικά ενεργό μέσον για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Κεντρικής Αμερικής και για να ενισχυθούν οι καλές σχέσεις που, έχουμε με, που υπάρχουν μεταξύ ημών και ημών. Με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα εγκρίνει αυτή την ε, συμφωνία η οποία στηρίζεται σε τρεις άξονες. Τον εμπορικό, τον πολιτικό και τον τομέα της συνεργασίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Περνάμε στον επόμενο μιλητή που είναι από τον Παναμά, ο Υπουργό Εθνούς Εμπορίου, τον Διαπραγματεύσεων και το Εθνούς Εμπορίου. Είναι η κυρία συγκεκριμένη, η κυρία Σαλασάρ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε Βιτάλ Μορέιρα, Πρόεδρε τη Επιτροπής Εθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και κύριοι βουλευτές, κύριε Κάρλ Ντεχούχτ, επίτροπε αρμόδια για το εμπόριο, κύριοι υπουργοί, υφυπουργοί, κύριοι πρέσβεις και αναπληρωτές υπουργοί από την Σκεντρική Αμερική, εκπρόσωπο διαφόρων ομάδων, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Αγαπητές κυρίες και κύριοι, είναι τιμή για τον Παναμά. Είναι μια πολύ σημαντική ε, στιγμή που μπορούμε να συμμετέχουμε σε αυτή τη δημόσια ακρόαση για τις εμπορικές και οικονομικές προοπτικές της συμφωνια Σύνδεσης μεταξύ των περιοχών μας. Πρόκειται για μια εμπορική συμφωνία μοναδική στον κόσμο που δείχνει πώ δύο περιοχέ, μια μεγαλύτερη, μια μικρότερη, μπορούν να διαπραγματευθούν μια εμπορική συμφωνία, η οποία είναι άρτια, είναι ισορροπημένη και με όρους αμοιβαίως επωφελείς και για τις δύο πλευρές, διότι ε, και τα ε, συμφέροντα των δύο πλευρών έχουν ληφθεί υπόψη. Θα ήθελα να μεταλλευτώ το χρόνο που μου δίνετε για να απευθυνθώ στο κροατήριό σας και να σας επαναλάβω τη δέσμευση της κυβέρνησης του Πρόεδρου Μαρτινέλη προς την αποτελεσματική εφαρμογή αυτής της συμφωνίας. Όπως γνωρίζετε, ο Παναμάς βασίζεται, ε, στηρίζεται στην ανταλλαγή υπηρεσιών και αγαθών, στο εμπόριο. Ιστορικά η οικονομία μας και η ανάπτυξή της ε, είχε σχέση με τις εμπορικές δραστηριότητες, τις επενδύσεις. Και έτσι καταφέραμε να εκμεταλλευτούμε και τη γεωγραφική μας θέση τη τις υπηρεσίες τις οποίες παρέχουμε και έχουμε αποκτήσει παράδοση από γενιά σε γενιά τις διαρθρωτικές βέβαια εσωτερικές μεταρρυθμίσεις ε, που χρειάζεται και να γίνουν από τις ε, δημόσιες διοικήσεις. Έχουμε λοιπόν αυτή την προοπτική και θα ήθελα να σα ε, εκφράσω εξ ονόματο τη κυβέρνηση του Παναμά ότι αυτή η συμφωνία σύνδεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τους άλλους γείτονε και φίλους από την Κεντρική Αμερική φτάνει σε μια στιγμή όπου έχουμε αναπτύξει μια πολιτική εξωτερικού εμπορίου που είναι στέρεη και φιλόδοξη και έχουμε προετοιμαστεί επί σειρά ετών για αυτήν. Περιμένουμε λοιπόν και προσβλέπουμε ενθουσιασμό την ολοκλήρωση των διαδικασιών έγκριση και επικύρωση αυτή τη συμφωνία στην επίπεδο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι θα παγιωθούν οι ίδιοι στέρεοι πολιτικοί και κοινωνικοί και οικονομικοί δεσμοί που έχουν οι περιοχές μας και θα μπορέσει έτσι να επικρατήσει η ανάπτυξη, συνεργασία των δημοσίων διοικήσεων και θα ε, φανούν βέβαια όλα αυτά τα ευεργετικά αποτελέσματα και στον παραγωγικό τομέα. Θα σας δώσω κάποια στοιχεία για τις ανταλλαγές τις εμπορικές που έχουμε για να διαπιστώσετε πόσο μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης ε, σημαίνει αυτή η συμφωνία για τον Παναμά που είχε πάντοτε διεθνές, ε, ε, διεθνείς εμπορικές σχέσεις. Μια τέτοια εμβέλεια, μια τέτοια φύση συμφωνία είναι βιώσιμη μόνο όταν υπάρχει δέσμευση μετασχηματισμού, μεταρρυθμίσεων και από τις δύο πλευρές, ώστε υπεύθυνα να τηρηθούν οι δεσμεύσεις που έχουν αναλυφθεί. Στη δική μας περίπτωση διαπραγματευτήκαμε και με άλλους σημαντικούς εμπορικούς εταίρους και συγκεκριμένα την διαδικασία, η διαδικασία μάλλον ενσωμάτωσης του Παναμά στο σύστημα ε, της κεντροαμερικανικής ολοκλήρωσης, το ΣΥΚΑ. Μας ε, βοήθησε να ολοκληρώσουμε τα καθήκοντά μας και να είμαστε έτοιμοι για τη θέση σε ισχύ των συμφωνιών και βέβαια να τηρούμε τα πρότυπα και τις που έχουμε αναλάβει για την ε, ανάπτυξη και την κοινωνική ειρήνη. Θέλω να σας πω ότι από τότε που ολοκληρώθηκαν ουσιαστικά οι διαπραγματεύσεις μας, το Μάιο δηλαδή του 2010, ο Παναμάς και οι χώρες της κεντροαμερικανικής περιοχής από κοινού κάναμε κάποια βήματα, ε, ολοκληρώσαμε κάποια στάδια για να μπορέσουμε να ενσωματωθούμε στο υποσύστημα της ε, κεντρομερικανικής οικονομικής ολοκλήρωσης. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια φάση διαπραγματεύσεων ορισμένων όρων, προϋποθέσεων και προθεσμιών για να έχουμε και το πρωτόκολλο ενσωμάτωσης του Παναμά σε αυτό το υποσύστημα που σας είπα. Και ήθελα να σας πω σε αυτό το πλαίσιο ότι είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός εμπορικός εταίρος ε, οι υπόλοιπε χώρες Κεντρικής Αμερικής για τον Παναμά. Η Κεντρική Αμερική ως περιφέρεια, όπως δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία, είναι ο τρίτος κατά ε, σειρά ε, εμπορικός μας εταίρος. Και μεταξύ των δέκα βασικότερων προορισμών των εξαγωγών μας, οι τρεις είναι χώρες Κεντρικής Αμερικής. Επίσης, έχουμε διατηρήσει πολύ αρμονικές σχέσεις και συντονισμό και στις διεθνείς μας σχέσεις Οπότε καταφέραμε πρόσφατα να ολοκληρώσουμε από κοινού κάποιε διαπραγματεύσει. Μία άλλη σημαντική πτυχή που αποτελεί και ιδιαιτερότητα τη χώρα μα είναι ότι τα τελευταία τρία χρόνια έχουμε εγκρίνει σημαντικά μέτρα δημόσιων πολιτικών τα οποία μας έδωσαν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε την κρίση του 2008 και να ενισχύσουμε το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα. Μεταξύ των μέτρων που εγκρίθηκαν ε, ήταν ε, η αναδιάρθρωση των δημοσίων δαπανών της φορολογικής πολιτικής ε, και η σύναψη συμφωνιών για την αποφυγή διπλής φορολόγησης με σημαντικούς μας εταίρους, μεταξύ αυτών και πολλοί από την Ευρώπη. Ποιο είναι το μήνυμα που στέλνουμε, είναι ότι η Ευρώπη είναι ένας υπεύθυνο εταίρος μας. Το ίδιο βέβαια είναι και η όλη η περιοχή αυτή η οποία εξελίσσεται ε, σύμφωνα με τις ανάγκες και τηρώντας ε, τις δεσμεύσεις. Οι χώρες Κεντρικής Αμερικής επίσης έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο, σημαντικά επιτεύγματα. Στην περίπτωση του Παναμά, οι επενδύσεις, οι εξαγωγές τη ε, της Ευρώπης προς τις δικές μας χώρες έχουν, χώρα έχουν αυξηθεί πολύ σημαντικά την τελευταία δεκαετία. Και πιστεύουμε ότι είναι σίγουρα σημαντική για την Ευρώπη η Κεντρική Αμερική και η παγίωση των σχέσεων, αλλά και τούμπαλιν βέβαια, διότι δεν πρόκειται απλά και μόνο για εμπορικούς εταίρους. Είμαστε στρατηγικοί εταίροι ε, προ όφελο τη οικονομική μα ανάπτυξη, αλλά βέβαια και για την ευημερία πάνω απ' όλα των πολιτών μα. Αγαπητοί ε, βουλευτέ, αγαπητέ κυρίε και κύριοι, δεν θέλω σε καμία περίπτωση να δοθεί εντύπωση ότι έχουμε ολοκληρώσει το έργο μα. Φυσικά υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα που εκκρεμούν. Και φυσικά και μπορούμε να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο του μηχανισμού μα για να τηρήσουμε τι νέε δεσμεύσει και για να συμπίξουμε τι νέε μα στρατηγικέ σχέσει. Από τη δική μα πλευρά, την Κεντρική Αμερική, εμεί είμαστε έτοιμοι, είμαστε ενθουσιώδεις ε, ε, με αυτή την προοπτική να αναλάβουμε τη δέσμευση, την ίδια δέσμευση που θα αναλάβει βέβαια και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σα ευχαριστώ πολύ. Thank you Next, uh, Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής θα είναι εκπρόσωπος της Κώστα Ρίκα, ο πρέσβης Τομάς Ντουένιας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 su apoyo para convertir este acuerdo de asociación en una realidad. Muchas gracias, señor presidente. Thank you. Thank you very much indeed. And to conclude the presentations from El Salvador, Ambassador. Θα δώσω τώρα το λόγο στον Φρανθίσκο Λίμα, που είναι ο πρέσβης του Ελ στον ΠΟΕ, Πού είστε? Α, εκεί. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε Ντεχούχτα και άλλης κομισιόν που τον συνοδεύετε, κύριε Υπουργοί, Υφυπουργοί, κυρίε και κύριοι βουλευτές, ε, σύντροφοι κύριοι πρέσβεις, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, εξ ονόματος της κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Σαλβαδόρ θα ήθελα καταρχάς ε, να ε, ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους του Υπουργού Οικονομικών, ε, ο οποίος για ανηλυμένες επίσημες υποχρεώσεις δεν μπόρεσε να παραστεί στην σημαντική αυτή συνάντηση. Το τουλεχθέντος βράτω με τις ευκαιρίες που μας δίνεται για να σας παρουσιάσω τις δικές μας προοπτικές για το οικονομικό και εμπορικό σκέλος της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ Κεντρικής Αμερικής και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από αυτό το πρίσμα, η Συμφωνία Σύνδεσης ε, θεωρήθηκε πάντοτε από εμάς ως ένα μέσο που θα ενισχύσει ε, τη σχέση μεταξύ των δύο περιφερειών, θα συμβάλλει στην οικονομική και ανάπτυξη του Σαλβαδόρ μέσω νέων ευκαιριών εξαγωγών τόσο αγαθών όσο και υπηρεσιών, που θα οδηγήσει σε διαφοροποίηση των αγορών ε, και σε διεύνηση της εξαγωγικής βάσης και των ξένων άμεσων επενδύσεων. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο τρίτος εμπορικός εταίρος εκτός της ε, Υπήρου μας για το El Πολύ μεγάλη αύξηση των εισαγών είδαμε τα τελευταία χρόνια. Υπερβαίνουν τα 300 εκατομμύρια ευρώ, μάλιστα το έτος 2011. Επίσης, η αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξακολουθεί να είναι μια από τις μεγαλύτερες οικονομίες σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε το ΑΕΠ, είναι μια αγορά 500 εκατομμυρίων ανθρώπων, άρα πάρα πολύ ελκυστική αγορά για προοπτικές εξαγωγής υπηρεσιών και προϊόντων, αλλά και για επενδύσεις. Μεταξύ των βασικών εξαγωγών του Σαλβαδόρ στην Ευρωπαϊκή Ένωση τονίζουμε προϊόντα όπως ε, καφέ, ζάχαρη, μελάσα ε, από το ζαχαροκάλωμ και τα λοιπά. Ε, δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία στις ποσοστώσεις τις οποίες πραγματευόμαστε με τα προϊόντα όπως ε, ο τόνος, ε, η, κάποια προϊόντα μεταποίησης, η ζάχαρη, γιατί θέλουμε να μην ε, υπάρχουν ασυμμετρίες. Θέλουμε στην ε, συμφωνία αυτή να δούμε ένα μέσο το οποίο θα επιτρέψει αφενός να απελευθερωθεί προοδευτικά το εμπόριό μας και αφετέρου να γίνουν σεβαστές οι δεσμές μας ό,τι αφορά το περιβάλλον ε, και τα εργασιακά για να αναπτύξουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη των λαών μας. Από την άλλη πλευρά οι άμεσε ξένε επενδύσει για μικρέ χώρε όπω είναι το Σαλβαδόρ είναι ένα από τα βασικότερα εργαλεία για την πρόωθηση τη δημιουργία θέσεων απασχόληση και στον τομέα τη βιομηχανία, όσο και στον τομέα των υπηρεσιών. Από αυτή την έννοια η Συμφωνία σύνδεση προωθεί την προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων στο βαθμό ε, που παρέχει προβλεψιμότητα μακροπρόθεσμα για του επενδυτέ. Όλα αυτά επανεπιβεβαιώνουν τη, συμμαχία, τη σημασία που δίνει το Σαλβαδόρ σε αυτή τη συμφωνία σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο γιατί παγιώνει και διευρύνει τις ε, δοσμολογικές προτιμήσεις ε, μέσω του γενικευμένου συστήματος προτιμήσεων, αλλά γιατί παρέχει ασφάλεια δικαίου αυτό το νέο μέσο και στους, ε, στους επενδυτές και στους εξαγωγείς των δύο περιοχών, διότι θεσπίζονται σαφείς μόνιμοι κανόνες για τα εμπορικά θέματα η διαπραγμάτευση αυτής της συμφωνίας και η εφαρμογή της ε, θα οδηγήσει και σε μεγαλύτερη εμβάθυνση της κεντροαμερικανικής ολοκλήρωσης με βάση τη σημαντική πρόοδο που ήδη έχουμε επιτύχει σε αυτό το τομέα ως ε, περιοχή. Διαδικασίες δασμολογικές, ε, τεχνικά μέτρα, φυτογενομικά, υγειονομικά μέτρα και ούτω καθεξής. Οι διεθνείς περιφερειακές σχέσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές όπως δείχνει το ότι από τότε που θεσπίστηκε η κεντροαμερικανική ε, νέα αγορά μέχρι σήμερα, οι διαπεριφερειακές ε, ανταλλαγές έχουν αυξηθεί κατά 11,5% ετησίως και αυτό μεταφράζεται σε πάρα πολύ σαφή κέρδη για την περιοχή. Οι μικρομεσαίες και πολύ μικρές επιχειρήσεις παίρνουν το 75% ε, του μεριδίου αυτού. Με τη Συμφωνία Σύνδεσης θα, διευρυνθεί ακόμη περισσότερο η κεντροαμερικανική ολοκλήρωση, όταν ε, το, ο Παναμάς μάλιστα θα ενταχθεί στο ΣΥΚΑ, το σύστημα της κεντροαμερικανικής ολοκλήρωσης. Μέσω της Συμφωνίας Σύνδεσης επίσης, πετύχαμε να ενισχύσουμε και τους δεσμούς συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο να, ε, δώσουμε, να αναζωογονήσουμε την ανάπτυξη και να έχουμε περισσότερο ανεπτυγμένους ε, θεσμούς για την εφαρμογή της Συμφωνία Σύνδεσης ώστε όλες οι χώρες να επωφεληθούν ε, τα μάλλα από αυτή τη συμφωνία. Κυρίως δε η εξαγωγή από μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Η δημόσια κρόαση αυτή είναι πάρα πολύ σημαντικό στάδιο της διαδικασίας μέχρι την υπογραφή και επικύρωση της Συμφωνία Σύνδεσης, ώστε να έχουμε πλέον απτά αποτελέσματα και ωφέλη και για τις δύο πλευρές. Ευχαριστώ. Thank you very much. This close is the... Ευχαριστώ. Έτσι ολοκληρώνουν οι παρουσιάσει των ε, συμφωνιών από την Ευρωπαϊκή Συμφωνία, μάλλον από την Επιτροπή και του εκπροσώπου των κυβερνήσεων της, ε, των χωρών τη Ευρωπαϊκή Κεντρική. Συνεχίσουμε τώρα με τη συζήτηση. Και θα δώσω το λόγο στον κύριο Παύλο Σάλβα, εισηγητή τη Επιτροπή μα σε θέματα εμπορίου και οικονομικών σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Αμερική. Κύριε Σάλβα, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, Κύριε Υπουργοί, κύριε Υφυπουργοί, κύριοι πρέσβοι, σας ευχαριστούμε για τις ε, παρουσιάσεις σας και για το ενδιαφέρον που επιδεικνύεται για να επικυρωθεί το συντομότερο δυνατό αυτή η συμφωνία. Συμφωνώ με την σημασία την οποία έχει η συμφωνία αυτή, δεδομένου ότι πρόκειται για την πρώτη συμφωνία διαπεριφερειακή μεταξύ Κεντρικής Αμερικής και Ευρωπαϊκής Ένωσης πιστεύω ότι εκπροσωπεί ένα οικονομική και κοινωνική πρόκληση ανευπροηγουμένου η συμφωνία αυτή και κυρίως για την Κεντρική Αμερική. Πρόκειται για μια ισοσκελισμένη συμφωνία που δίνει δυνατότητες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Κεντρική Αμερική. Εξάλλου πρόκειται για μια συμφωνία που θα βελτιώσει τις επενδύσεις και θα τις καταστήσει πιο ασφαλείς. Και Βεβαίως σε θέματα υπηρεσιών, σε θέματα ανανεώσιμων πηγών ε, ενέργειας και στον τομέα της αναυτοκινητοβιομηχανίας θα είναι υποφελής η συμφωνία αυτή για την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα αποφέρει και προφανή ωφέλη για την Κεντρική Αμερική. Όχι μόνο διότι θα αυξήσει και το ΑΕΠ δεδομένου ότι είμαι σίγουρος ότι θα έχει ωφέλη ακόμη και μεσοπρόθεσμα, αλλά θα είναι και ένα πολύτιμο μέσο για να υπάρξει και η ενοποίηση της περιοχής αυτής. Βεβαίως, ακόμη έχουμε πολλά να κάνουμε και είμαι σίγουρος ότι η συμφωνία αυτή θα μπορέσει να βοηθήσει την ε, ε, περαιτέρω ενσωμάτωση όλων των κρατών της Κεντρικής Αμερικής. Ακούσαμε ε, πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, ακόμη για τις εσωτερικές αγορές κάθε χώρα της Κεντρικής Αμερικής και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι μία δυνατότητα ε, συνοχής κοινωνικής, αηφόρου ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης ποιότητας. Τελικά θα ήθελα να τονίσω τις δυνατότητες που δίδονται όσον αφορά την διαφοροποίηση των οικονομικών της Κεντρικής Αμερικής. Αυτή η συμφωνία θα πρέπει να αποτελέσει την ευκαιρία ώστε οι οικονομίες των κρατών μελών της κρατικής Κεντρικής Αμερικής να διαφοροποιηθούν. Ελπίζει και φιλοδοξεί η Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο να βασίζουν σε αγροτικά προϊόντα της εξαγωγής οι χώρες Κεντρικής Αμερικής, αλλά όπως και η Κωνσταντίνα να εξειδικευτεί σε, προηγούμενα, σε προϊόντα μεγάλης προστιθέμενης αξίας, όπως τα microchips ή άλλες υπηρεσίες. Γι' αυτό θα ήθελα να πω σε όλους τους συναδέλφους της Κεντρικής Αμερικής να καταβάλουν προσπάθειες ώστε να επικυρωθεί σύμφωνα η συμφωνία και να μπορέσουμε να υποφεληθούμε το συντομότερο δυνατό από τις ευκαιρίες που μας δίδονται. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Πάολο Φάλμπα είναι μέρος του ΕΛΚΑ. Ο επόμενος είναι ο κύριος Βιτολάσλη, εξεισηγητής για τα νομοθετήματα που διέπουν την διμερή ρήτρα διασφάλισης της συμφωνίας. Ο κύριο Λάιφτφριτ, εκπρός των σοσιαλιστών, λοιπόν. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Μια και τα ισπανικά μου είναι ανύπαρκτα και δεν θα με καταλάβει κανείς αν μιλήσω ισπανικά, θα μου επιτρέψετε να μιλήσω αγγλικά. Δεν νομίζω ότι θα δυσκολευτεί κανείς εδώ. Ως εισηγητής λοιπόν για τη ρήτρα Έχω δουλειά κάπως έχω καθήκον λίγο διαφορετικό από ε, του συναδέλφου που είναι εισηγητής για ολόκληρη τη συμφωνία. Με ένα καθήκον μου είναι να προστατεύσω όχι μόνο τα ευρωπαϊκά συμφέροντα, αλλά και να μεριμνήσω το εμπόριο όπως θα αναπτύσσετε να αναπτύσσετε σε ισότιμο θεμητό ε, τρόπο. Είναι σχετικά δύσκολο κεφάλαιο αυτό των ε, οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φερρυπίν τα συμφέροντα των υπερ ε, απομακρυσμένων, των υπερβολικά απομακρυσμένων περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παραδείγματι πρέπει να προστεθούν. Έχουμε επίσης θέματα σχετικά με τους ε, παραγωγούς μπανάνας που θα πρέπει να συζητηθούν ε, και γι' αυτό ήθελα να επισημάνω. Αλλά πάντως θέλω να πω ότι όλη η διαδικασία ήταν πολύ ενδιαφέρουσα για μένα. Ιδιαίτερα δεδομένου ότι η κοινωνία των πολιτών από την Κεντρική Αμερική μου επεσήμανε κάποια προβλήματα διαφορετικά ίσως από αυτά που θα έπρεπε να απασχολούν τον ε, εισηγητή της, ε, τον αρμόδιο διασφάλισης, αλλά εγώ πάντοτε κοιτάω τα συμφέροντα ε, όλων όσοι εργάζονται σε, και στις δύο όχθες του Ατλαντικού. και στην Κεντρική Αμερική, πάντα βέβαια μεριμνώντας και για τα δικαιώματα των εργαζομένων, των μικρότερων επιχειρήσεων που παράγουν αγαθά. Και ιδιαίτερα εταιριών που παράγουν βιολογικά προϊόντα ή που ε, αναπτύσσουν θεμητό εμπόριο. Έτσι λοιπόν η ρήτρα διασφάλισης θα πρέπει να αποβαίνει πιστεύω προς όφελος και να προστατεύει την ευρωπαϊκή βιομηχανία και τα συμφέροντα της Ευρώπης, αλλά και κάθε εργαζόμενο που μοχθεί είτε από τη μια είτε από την άλλη πλευρά της, του Ατλαντικού ε, σε κάποια επιχείρηση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω του υπουργού από την κεντρική τη Χώρα και τη Αμερική που έλαβαν τον λόγο εδώ για την ε, υποστήριξή του. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ πριν ακούσουμε άλλα μέλη της Επιτροπής, σε ακούσουμε τους ε, ειδικού μας εκπροσώπους, προσκεκλημένους. Και ξεκινώ με τον κύριο Woolcock από το London School of Economics, ο οποίος είναι ανεξάρτητος ε, εμπειρογνώμων για θέματα εξωτερικού εμπορίου. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Καθήκον μου είναι να σας ε, παρουσιάσω συνοπτικά μια μελέτη που καταρτήσαμε για την Επιτροπή σας ε, με συμμετοχή διαφόρων παραγόντων, αλλά πάντως θα αναφέρω συνοπτικά κάποια πορίσματα και ξεκινώ με σχόλιο ως προς το κατά πόσον η συμφωνία ε, είναι συμβατή, με, ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την εμπορική πολιτική. Πρώτα απ' όλα, ο στόχος της προαγωγής της περιφερειακής ολοκλήρωσης που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ικανοποιείται. Δεύτερον, είναι μια συνολική συμφωνία και σύμφωνη με την κρατούσα ερμηνεία του άρθρου 24 της ΓΑΤ 1994 και του άρθρου 5 της ΓΑΤ, της Συμφωνίας δηλαδή για τις εμπορικές συναλλαγές στο, στις υπηρεσίες. Ε, επίσης, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου εν γέννη τίνει προς ανάπτυξη νέων πιθανών αγορών. Εδώ είναι λιγότερο προφανές το κατά πόσο η ευρωπαϊκή πολιτική αυτή ικανοποιείται, γιατί η Κεντρική Αμερική καλύπτει μόνο το 0,5% των εισαγωγών και 0,3% ε, των εξαγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το έτος 2010. Μεν Πλην όμως, από ό,τι είδαμε, από ό,τι μαθαίνουμε, η Κεντρική Αμερική έχει προχωρήσει σε ταχύ αύξηση των όγκων του ιστορικού εμπορίου και δεδομένου αυτού του, αυτού του στοιχείου θα μπορούσε να στηριχθεί το επιχείρημα ότι είναι συμβατή με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετική συμφωνία. Λιγότερο προφανές είναι το να προσπαθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των Συμφωνιών Ελευθερών Συναλλαγών να καλύψει έδαφο χαμένο σε σχέση με άλλου παράγοντε του εθνού εμπορίου, όπω οι ΗΠΑ προκειμένου και τι σχέσει του με την Δομενικανή Δημοκρατία, την Κεντρική Αμερική ε, και βέβαια τον Καναδά. Και σε αυτό το τομέα θα ήθελα να πω ότι η συμφωνία τουλάχιστον καλύπτει τις συνθήκες της συμφωνίας ε, με τις ΗΠΑ και τον Καναδά. Επίσης, κέρδος ευημερίας. Το κέρδος ευημερίας δεν βλέπουμε να κατανέμεται ισομερός μεταξύ των κρατών της Κεντρικής Αμερικής, 3,5% επί του ΑΕΠ για την Κωνσταντίνα, η εκτίμηση μάλλον αισιόδοξη. από την ε, μελέτη επιπτώσεων, αλλά υπάρχουν και κάποια άλλα σημαντικά ωφέλη, τα οποία, όπως είπα όμως, δεν είναι ισομερώς κατανεμημένα μεταξύ των διαφόρων κρατών. Η Κεντρική Αμερική αναφέρεται ότι θα έχει, προβλέπεται ότι θα έχει ε, κέρδος, δηλαδή αύξηση των εξαγωγών, κατά πάσα πιθανότητα θα ενισχυθεί δηλαδή το εμπορικό πλεόνασμα της Κεντρικής Αμερικής στις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως γνωρίζετε, ίσως η Κεντρική Αμερική ήδη έχει αδασμολόγητη πρόσβαση ε, μέσω του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων ε, GSP+, εκτός από προϊόντα όπως η μπανάνα, η ζάχαρη και κάποια άλλα προϊόντα. Εν πάση περιπτώσει όμως ε, κάποια κύρια θέματα είναι ότι εξασφαλίζονται μακροπρόθεσμα τιμησιακές συνθήκες πρόσβασης, ανεξαρτήτως της όποιας ε, μεταρρύθμισης του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κέρδος εφημερίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση επί του ΑΕΠ σχετικά αμεληταίο, 2,3 δις ε, κέρδος προβλέπονται, αλλά μάλλον είναι υπεραισιόδοξη η εκτίμηση. η Ευρωπαϊκή Ένωση κερδίζει ως προς τη δυνατότητα ενισχυμένης πρόσβασης για τα κλασικά προϊόντα όπως τα μηχανήματα, ε, τα αυτοκίνητα, αλλά και ιδιαίτερα οι υπηρεσίες. Οι δε από την Κεντρική Αμερική για, τους, ε, για τα κεφάλαια 1, 2, 3 των υπηρεσιών ξεπερούν σε μεγάλο βαθμό τις δεσμεύσεις της GATS, αλλά μην ξεχνάμε ότι η GATS είναι μια συμφωνία που συνήθει από 20 χρόνια ένα-δύο σημεία για λεπτομέρειες πτυχές. Οι όροι προέλευσης, κανόνας προελέυσης ε, αναφέρονται στην ε, σώρευση που αφορά εσωτερικό εμπόριο μέσα σε μια ευρύτερη περιοχή και επομένως αυτή η διαγώνια λεγόμενη σώρευση καλύπτει διάφορες χώρες αλλά υπάρχει και δυνατότητα για επέκταση της και σε άλλες χώρες της ίδιας περιφέρειας με την οποία συνήψε συμφωνία Εμπορική Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς τα, ως τεχνικούς φραγμούς και μέτρα υγειονομικής προστασίας που μπορούν να αποτελούν σημαντικούς φραγμούς άπαξ και καταργηθούν οι τελωνιακοί δεσμοί. Είναι η συμφωνία με τους όρους της ΠΟΕ και με τα διαδικαστικά μέτρα της ΠΟΕ εν προκειμένου με τη θέσπιση ειδικευμένων επιτροπών που θα αντιμετωπίζουν ή αδίποτε ε, αναφιόμενα προβλήματα. Μέτρα ρύθμισης του εμπορίου, αντι-dumping, αντισταθμιστική δασμή και άλλα υπάγονται στην ρήτρα διασφάλισης, πολυμερής μάλλον ρήτρες διασφάλισης του άρθρου 19 της ΓΑΤ ή του άρθρου 5 της Συμφωνίας για τη Γεωργία διμερείς ρήτρες διασφάλισης επίσης προβλέπονται στο άρθρο 104 διμερός συμπληρωματικά ως προς άλλα ε, διμερεί μέτρα που είναι πάγια στις συμφωνίες ελευθερών συναλλαγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντως μπορούν να επιβληθούν και μέτρα διασφάλισης ειδικά για τις πλέον απομαξιμένες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή θα είναι ευρεία η θεώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ως προς τις, μη ε, τις πλέον απομακρυσμένες περιοχές. στον τομέα της πνευματικής διοκτησίας είναι συμβατές με τους κανόνες ε, οι διατάξεις, ενισχύουν, ε, δηλαδή αφυλάσσουν και ενισχύουν την ε, πνευματική διοκτησία, ιδιαίτερα στους τομείς που υπάγονται στην TRIPS Plus, Συμφωνία Ελευθεροπορίου στην Πνευματική Διοκτησία Plus, και ιδιαίτερα στις διατάξεις εκείνες οι οποίες καλύφθηκαν από τις διαπραγματεύσεις τις πρόσφατες διαπραγματεύσεις του 2001 με την ε, εισαγωγή, μάλλον επανεισαγωγή ε, μέτρων ευελιξίας και τη σχετική απόφαση του, Συμβουλίου, του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων του 2003 για την ερμηνεία της Συμφωνίας TRIPS, δημόσιες προμήθειες επενδύσεις, ανταγωνισμός επίσης καλύπτονται και πάλι δηλαδή έχουμε μια ευρύτατη κάλυψη. Περισσότερα, θέματα, περισσότερα σημεία στο θέμα αυτό δεν θα ε, εκθέσω, πέραν του ότι οι δεσμεύσει ως προς την αγορά. Ως προς τις αγοραστικές, ε, ως προς τις μονάδες αγοράς μάλλον ε, μπορεί να διαφοροποιείται από τη μία περιοχή στην άλλη, πέραν των κανόνων της ε, Συμφωνίας περί Δημοσίων Προμηθειών της, του ΠΟΕ. Καλύπτονται και τα θέματα των επενδύσεων. Οι χώρες της Κεντρικής Αμερικής έχουν τη δυνατότητα να αποκλείσουν κάποιους ευαίσθητους τομείς, χωρίς όμως συγκεκριμένους αποκλεισμούς από τη Συμφωνία οι επενδύσεις προστατεύονται δυνάμει των διμερών συμφωνιών, επενδύσεων. Όπως επίσης αναφέρθηκε ήδη, η συμφωνία περιλαμβάνει διατάξεις για την πολιτική του περιανταγωνισμού και την εισαγωγή μέτρων πολιτικής ανταγωνισμού και της ανάπτυξης μιας περιφερειακής αρχής για τον ανταγωνισμό εντός τριών ετών, ίσως με εξαγωγή του ευρωπαϊκού μοντέλου σε άλλες περιοχές. Ο πρόεδρο μπορείτε να μιλάτε, να, να ολοκληρώνετε σας παρακαλώ. Ναι, Πρόεδρε, κλείνω με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη βιώσιμη ανάπτυξη που, όπως αναφέρετε υπάρχει μια ε, πάγια ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα συμφωνίες, χωρίς όμως ιδιαίτερο μηχανισμό ή όργανο επαλήθευση της στήριξη αυτή. Μπορεί όμως να τον αλάβει κάποια ως άλλος φορές που θεσπίζεται για τη λειτουργία της συμφωνίας. Στην επαλήθευση μπορεί αυτή να ανατεθεί στις υφιστάμενες δομές δηλαδή και ιδιαίτερα στο τομέα της, της βιώσιμης ανάπτυξης. Περιλαμβάνονται οι κύριες προδιαγραφές του Παγκόσμιου Οργανισμού Εργασίας, και άλλες σχετικές κοινωνικές διατάξεις. Θα επισέλθω στις λεπτομέρειες, αλλά ε, υπάρχει θα έλεγα η δυνατότητα ενός μηχανισμού επαλήθευσης από εταίρους ή ενισχυμένου μηχανισμού επαλήθευσης από εταίρους, peer review. Αλλά δεν θα το εκθέσω προς τώρα γιατί δεν έχω χρόνο. Και επίσης εν γέννη θα λέγαμε ότι η α, χρησιμότητα της συμφωνίας θα αξιολογηθεί μόνο από τον τρόπο υλοποίησή τη Δεν κρίνεται τίποτα από την υπογραφή και μόνο συμφωνίας. Το πώς θα ε, υλοποιηθούν και πώς θα γίνει η παρακολούθηση της υλοποίηση των διαφορών πτυχών της συμφωνίας έχει σημασία. Μία σύσταση θα μπορούσαμε να διατυπώσουμε, δηλαδή το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή σας ιδιαίτερα, να μελετήσουν έναν τρόπο για πιο ουσιαστική παρακολούθηση της λειτουργίας της συμφωνίας. Ευχαριστώ. Περνάει ο χρόνος και έχουμε μείνει λίγο πίσω. Γι' αυτό θα είμαι λίγο πιο αυστηρός από εδώ και πέρα. Σε ό,τι αφορά το χρόνο αγόρευσης. Παρακαλώ λοιπόν τους επόμενους ομιλητές να μην ε, ξεπερνούν το χρόνο που τους έχει διατεθεί. Περνάμε λοιπόν τώρα στους εργαζομένους ε, και τον ε, Χωάν Μορένο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 δεν θα είμαι τόσο εγκομιαστικός ε, ως προς τη συμφωνία σε σχέση με τους προλαλήσαντες ε, και πραγματικά λυπούμε. Διότι εκπροσωπώ την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων, μια οργάνωση στην οποία ουσιαστικά συμμετέχουν σχεδόν όλοι οι Ευρωπαίοι συνδικαλιστές, ε, ενώ ο συνδικαλισμός όλων των ευρωπαϊκών χωρών ουσιαστικά από κάθε τάση που πάντοτε ήταν υπέρ ε, του διεθνούς εμπορίου και ήταν πεπισμένη ότι η πρόοδος της Ευρώπης ε, και η ισχύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από το άνοιγμά της προς τον κόσμο. Δηλαδή δεν είμαστε καθόλου προστατευτικοί. Θα σας εκφράσω όμως κάποιες επιφυλάξεις οι οποίες ε, κυρίως έχουν να κάνουν με κριτήρια αλληλεγγύης με τους εργαζομένους μιας περιοχής όπου Υπάρχουν πάρα πολλοί αρνητικές ε, συνθήκες. Ευθύς εξ αρχής ε, να πούμε ότι τα συνδικάτα του κεντροαμερικανικού ε, φορέα και της αντίστοιχης και της ΕΟΚΕ ουσιαστικά από κοινού παρακολουθούμε αυτή την συμφωνία. Αρχικά είχαμε μία θετική στάση και ελπίζαμε να έρθει σε αίσιο πέρα σε αυτή η συμφωνία. Θεωρούσαμε δηλαδή ότι θα μπορούσε να βοηθήσει. Δηλαδή να ενισχύσει τη διαδικασία ολοκλήρωση στην Κεντρική Αμερική αφενό και αφετέρου να βοηθήσει τις χώρες της περιοχής να περιορίσουν ή να υπερβούν τις εσωτερικέ ασυμμετρίες, αλλά κυρίως να βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας και να ε, μην έχουν περιορισμένα δικαιώματα, να αυξηθούν τα δικαιώματά τους. Τα δεδομένα, όχι μόνο τα συνδικαλιστικά, αλλά δεδομένα τα οποία επικαιρώνουν και οργανισμοί οι οποίοι δεν έχουν να κάνουν καν με το συνδικαλιστικό κίνημα, όπως και η Διαμερικανική Επιτροπή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Μα λένε ότι δυστυχώ παραμένουν πολύ σοβαρέ παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ένα φαινόμενο ατιμορρησία που το παρατηρούμε ε, σε όλη την περιοχή ουσιαστικά. Για να μιλήσω μόνο για την ε, Γουατεμάλα, 59 συνδικαλιστές έχουν δολοφονηθεί από το, 7, ε, από το 9 στο 11 και αυξάνεται ο αριθμός αυτός. Οι διεθνείς οργανισμοί πολλές φορές ε, δείχνουν προς την Κολομβία ως χώρα αναφοράς ε, για τις περιπτώσεις βίας κατά των συνδικαλιστών. Βλέπουμε να δολοφονούνται όμως στην Γουατεμάλα περισσότεροι συνδικαλιστές στη Γουατεμάλα από ό,τι στην Κολομβία. Περισσότερες γυναίκες ε, να δολοφονούνται στη Γουατεμάλα από ό,τι στο Μεξικό. Μιλώ για συνδικαλίστριες. Επίσης τα ποσοστά της εγγραφής σε συνδικάτα σε κλαδικές έχει από το 9 μειωθεί στο 2%. Λόγω αυτής του καθεστώτος ε, τρομοκρατίας και βίας που υπάρχει. Τα κεντροαμερικανικά συνδικάτα κατέβαλαν προσπάθειες για να πετύσουν εγγύησεις. Όχι μόνο να συμπεριληφθούν στη συμφωνία εγγυήσει για την τήρηση, παραδείγματο χάρη, των ε, συμφωνιών ε, του Διεθνού Γραφείου Εργασία, αλλά να υποχρεωθούν οι κυβερνήσει να υλοποιήσουν πολιτικές προώθησης ε, της αξιοπρεπούς εργασίας, πολιτικές προώθησης και προάσπισης της εργασίας, της προάσπισης ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των υπερμάχων του και του συνδικαλιστικού κινήματος εν γέννη. Νομίζω ότι εδώ έχουμε να κάνουμε ένα κοινωνικό κεφάλαιο. Δύο Ινστιτούτα, όχι εμείς, ε, αλλά δύο πολύ σημαντικοί φορείς έκαναν πολύ σημαντικές ε, προσπάθειες και από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και από πλευράς ε, Κεντρικής Αμερικής ένα έγγραφο το οποίο εκπονήθηκε για το θέμα αυτό δεν ελήφθη σοβαρά υπόψη παρότι είχε πολύ θετικά στοιχεία τα οποία δεν συμπεριελήφθησαν τελικά στα κείμενα που έχουν εγκριθεί. Παρότι θεωρούμε λοιπόν ότι υπάρχουν θετικά στοιχεία στη συμφωνία αυτή ιδίω σε ό,τι αφορά τι διάβλους συμμετοχή και τη διαδικασία που μπορεί να υπάρχει για την ενίσχυση της κεντροαμερικανική ολοκλήρωση, πιστεύουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έπρεπε να απευθύνει ισχυρή έκκληση ώστε να υλοποιηθούν και να εξασφαλιστούν μέχρι το μέλλον, ε, από εδώ και στο μέλλον βέβαια, αυτοί οι δομές που έχουν δημιουργηθεί, το φόρουμ ε, διαλόγου με, τον, ε, με τις κοινωνίες των πολιτών, διάφορες επιτροπές που επιτροπές, όχι απλά να λειτουργούν, αλλά να υπάρχουν εγγύσει ότι θα είναι αποτελεσματικά και θα έχουν και εκτελεστικό χαρακτήρα τα αιτήματά τους ε, και οι καταγγελίες τους. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θα ακούσουμε τώρα τον ε, κλάδο των επιχειρήσεων. Μάρτα Ράφεκα είναι η επόμενη ομιλήτρια εκπρόσωπος της ΓΑΜΕΣΑ. Ένας παγκόσμιος ε, παίκτη στον τομέα της ενέργειας, ε, κατασκευή ολικών ανεμογεννητριών, ολικών πάρκων. Δεν ξέρω που είναι η Μάρτα. Έχετε παρουσίαση PowerPoint. Απλά έχετε και περιορισμένο χρόνο στη θέση να το ξέρετε. Ε, ε, Χαίρετε κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, Υφυπουργοί, Πρέβης, Εκπρόσωποι. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή Εξωτερικού Εμπορίου που κάλεσε όλες αυτές τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής και τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων. Πριν αρχίσω να μιλώ για τα ωφέλη και τις ε, συμφωνίας αυτής για τους επιχειρηματίες, θα ήθελα να κάνω μία σύντομη παρουσίαση της επιχείρησής μας για να σας πω ποια είναι τα ωφέλη. Εδώ και 18 χρόνια ε, δραστηριοποιούμε στο τομέα αυτό. Είμαστε παρόντες σε 34 χώρες. Έχουμε 24.000 ΜΒ εγκαταστημένα ανά τον κόσμο και κατασκευάζουμε ε, τουρμπίνες για την ελληνική ενέργεια και αιωλικά πάρκα. Εδώ έχετε διάφορα στοιχεία, 16.000 βατ είναι οι συμβάσεις συντήρησης, 4.000 ΜΒ εγκατεστημένα για την πρόθεση των νέων ενεργειών. Και εδώ βλέπετε την ε, βιομηχανική βάση της εταιρείας μας, πώς, ε, ε, που είναι τα 34 βιομηχανικά μας κέντρα ανά τον κόσμο. Τα τελευταία χρόνια έχουμε πέντε παραγωγικά κέντρα και στη γραφική αυτή παράσταση βλέπετε πόσο σημαντική προσπάθεια διεθνοποίησης γίνεται εκ μέρους των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων τα τελευταία χρόνια. Το 2003 το 90% των μεγαβάτ που πολλούσαμε ήταν στην Ισπανία. Δέκα χρόνια μετά, 90% των ΜΒ πολλούνται εκτός Ισπανίας. Και αυτό είναι σαφές παράδειγμα της διεθνοποίησης των ε, προσπαθειών που καταβάλουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις για να επεκταθούν. 15% των πολίσεων μας το 2011 ε, γίνονται στην ε, Λατινική Αμερική με ποσοστό 19% το τέλος προηγουμένου του. Όλα λοιπόν αυτά τα μεγαβάτ που έχουμε ε, εγκαταστήσει ανά τον κόσμο αφορούν 36.000 τόνου του άνθρακος. Αν μιλήσουμε μόνο για τις δραστηριότητες της εταιρείας μας στις χώρες στις οποίες εκπροσωπούμε στην Κεντρική Αμερική, Πρέπει να πω ότι έχουμε διάφορα μεγαβάτ τα οποία έχουν εγκατασταθεί και παράγουν ενέργεια. Μπόρεσα να μιλήσω με τον ε, υφυπουργό της Ονδούρα και ε, μιλήσαμε για αυτό το οποίο θα γίνει στην Ονδούλα, το μεγαλύτερο ε, πάρκο αιωλικό που θα είναι το μεγαλύτερο πάρκο ανά τον κόσμο καλύπτει το 80% των ενεργειακών αναγκών της Ονδούρας και καλύπτει και την ε, παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε πολλές περιοχές της Ονδούρας, οι οποίες μέχρι τώρα δεν είχαν πρόσβαση σε αυτήν. Τώρα θα σας μιλήσω, αν έχω χρόνο, για αυτό το οποίο είναι σημαίνει για μας αυτή η συμφωνία. Είναι ένα βήμα προς τα μπρος για την ε, παγιοποίηση περαιτέρω καλών εμπορικών σχέσεων. Πρόκειται για μια συμφωνία η οποία έχει οριμάσει, αλλά θα πρέπει να συνεχίσουν οι προσπάθειες ώστε η παρουσία μας να γίνεται όλο και πιο σημαντική στις χώρες αυτές. Και βεβαίως θα πρέπει να συνοδευτεί από διάφορα σχέδια ε, πρωτοβουλειών που θα αναλυφθούν σε όλες τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής. Στα πλαίσια κανόνων με διαφάνεια ώστε να μπορέσει να υπάρξει εγγύηση για τον τρόπο με τον οποίο οργανώνουμε τις δραστηριότητες μας μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Θα πρέπει να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία και το διάλογο ώστε να μπορέσουμε να βρούμε από κοινού πρωτοβουλίες σε διεθνές επίπεδο ώστε να μπορέσουν επιχειρήσεις σαν την Μέσα και άλλες να προοδεύσουν στις χώρες αυτές που εκπροσωπείται ώστε να υποφεληθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι. Με αυτή τη συμφωνία έχουμε την ε, πεποίθηση ότι θα μπορέσουμε να εργαστούμε για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με τις ε, διάφορες συμφωνίες που θα ρυθμίσουν την παροχή αυτής της ενέργειας και νομίζω ότι πολλές χώρες θέλουν επίσης να κάνουν επενδύσεις σε μια τεχνολογία η οποία έχει αποδείξει ότι έχει φτάσει σε όριμο στάδιο που είναι αυτό της ιολικής ενέργειας. Έχουμε ακόμη πολλά να κάνουμε. Υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες για την ανάπτυξη αυτών των περαιτέρω καθαρών ενεργειών που βοηθούν όχι μόνο να αναπτυχθούν σε περιφερειακό, τοπικό, αλλά εθνικό επίπεδο οι χώρε αυτέ, αλλά είναι ένα βήμα προ τα μπρο ακόμη ώστε να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε του στόχου τη αηφόρου ανάπτυξη και να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τι δεσμεύσει που έχουμε αναλάβει για την μείωση των εκπομπών καυσαερίων. Τελειώνοντα, θα ήθελα να τονίσω ότι με μεγάλη ευχαρίστηση η μέσα ε, και μεγάλη περηφάνεια παρίσταται εδώ και αυτό αποδεικνύει πόσο σημαντικό είναι αυτό το οποίο γίνεται εδώ και για τη δική μας εταιρεία και για τις άλλες εταιρείες που δραστηριούνται στις χώρες αυτές και ελπίζουμε ότι το συμφωνία αυτή θα προχωρήσει παρόλο, το οποίο, παρόλο που ξέρουμε ότι έχουμε πολλά να κάνουμε ακόμη σε πολλούς τομείς. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Next speaker. Και τώρα έχουμε τον εκπρόσωπο της ε, Κοινωνίας των Πολιτών της Κρατικής Αμερικής, την εκπρόσωπο της κοινότητας των Πολιτών και της Μάντα Μαντακρούς από την Ονδούρας. Συμβούλιο Κοινωνικών Υποθέσεων της Οικονομίας από την Ονδούρα που είναι η Αμάντα. Καλησπέρα σας κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι. Κατάγομαι από ένα λαό εργατικό, με επιχειρηματικό πνεύμα, δημοκρατικό, που εμπνέεται από ανθρωπιστικά αισθήματα και παιδεία. Δυστυχώς όμως αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση όλο και μεγαλύτερης βίας, με περισσότερες ανθρωποκτονίες, ίσως τις, μεγαλύτερες, περισσότερες στον κόσμο, που ζούμε μέσα σε ένα καθεστώ ε, πολύ εύθραυστο από δημοκρατική πλευρά, όπου επικρατεί διαφθορά και καθεστώς ατιμορρησία. Για την Ονδούρα μιλάω. Είναι μια χώρα όπου έγινε ένα πραξικόπημα ε, τον Ιούνιο κλείνει τα τρία χρόνια και έχει δημιουργηθεί εκ τότε μια κοινωνικοπολιτική κρίση που δεν μπορεί ακόμη να επιληθεί. Ήρθαμε σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μιλήσουμε για τη Συμφωνία Σύνδεσης, την οποία θα αναφέρω ως ΚΑΦΤΑ ΣΥΝ, ΚΑΦΤΑ ΠΛΑΣ. Διότι αυτή η συμφωνία χρησιμοποιήθηκε ως βάση ε, για τη διαπραγμάτευση και είχε ως αποτέλεσμα να πετύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση μεγαλύτερα πλανεκτήματα για τις επιχειρήσεις. Ο στόχος μου δεν είναι να μιλήσω σήμερα για την ΚΑΦΤΑ, αλλά τα πέντε χρόνια ε, της ισχύω αυτής της συμφωνίας έδειξε ότι είχε αποτελέσματα τα οποία τελικά είναι αντίθετα με τους επιδεκόμενους αρχικά στόχους. Αυτή είναι η δική μας εμπειρία. Γι' αυτό και είναι απαραίτητο να γίνει κάποια σύγκριση με την ε, συζητούμενη σήμερα Συμφωνία Σύνδεσης. Θα περιοριστώ στη σημερινή παρουσίαση σε τρία σημαντικά σημεία για τα οποία υπάρχουν επίσημα στατιστικά στοιχεία, στα οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση. Πρώτο σημείο, ασυμμετρίες. Οι ασυμμετρίες είναι ξεκάθαρες και τις βλέπουμε σε τρία επίπεδα. Από τη μια περιοχή στην άλλη, μεταξύ των χωρών, αλλά και εσωτερικά σε κάθε χώρα. Από αυτές τις ασυμμετρίες μπορεί κανείς να ξεχωρίσει πρώτα απ' όλα η παγίωση εμπορικών σχέσεων με την Ευρώπη βάσει εξαγωγών πρώτων υλών και εισαγωγή και μεταπημένων προϊόντων. Μα πώς μπορούμε να αναπτύξουμε την περιοχή μας με φρούτα, λαχανικά και φουντούκια. Έχει αποτύχει αυτό το εξαγωγικό μοντέλο. Δεύτερον, τεχνολογικές διαφορές παραγωγής που δημιουργούν πολύ τεράστιε ε, ανισορροπίες και βάζουν σε πάρα πολύ μονεκτική θέση την Αμερική σε σχέση με την Ευρώπη. Και πώς μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί και τις γεωργικές επιδοτήσεις, που ούτε καν συζητήθηκαν στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Δεύτερο σημείο, περιβαλλοντική, περιβαλλοντικά προβλήματα και κοινωνικές επιπτώσεις. Ε, έχουμε, ε, είμαστε στην περιοχή μας ε, σε πολύ δύσκολη θέση από πλευράς περιβάλλοντος και θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερη πίεση, θα έχουμε συγκέντρωση εδαφών, θα έχουμε ε, απερίμωση των δασών, κατάχρηση και υπεκμετάλλευση του ύδατος για να αναπτυχθούν μονοκαλλιέργειες για γεωργικά καύσιμα και τελικά ε, θα έχουμε ρήπανση του αέρα και άλλε επιπτώσει πολύ αρνητικέ που άμεσα μπορεί κανεί να τι δίδει σήμερα με πλημμύρε το χειμώνα και ξηρασία το καλοκαίρι, Καταστραφή των οικοσυστημάτων και τη βιοπικιλότητα. Αυτά, μερικά από αυτά τουλάχιστον, τα έλεγε ήδη μια μελέτη κοινωνικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων που δεν λήφθηκε όμω καθόλου υπόψη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Άρα το κεφάλαιο εμπορίου ανάπτυξη βιώσιμη, δεν δίνει καμιά απάντηση για την αποφυγή αυτών των προβλημάτων, εδώ, ενώ, με ένα, ενώ δε αποκλείει και τους μηχανισμούς επίλυσης διαφορών για τα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης. Επομένω, αυτή, την έννοια η συμφωνία σύνδεση δεν είναι καύτα συν, αλλά καύτα μείον. Ένα άλλο θέμα σημαντικό, το παριθμό 3 που θέλω να αναφέρω, είναι η απασχόληση και η μετανάστευση. Έχει μειωθεί η απασχόληση και στην Ήπεθρο και στις πόλεις, λόγω κακών επενδύσεων και συγκέντρωση των πόρων. Και με την καύτα αλλά και με άλλε συνθήκες ελεύθερου εμπορίου που ισχύουν στην περιοχή βλέπουμε ότι δεν εποφελήθηκαν των ευκαιριών οι περισσότεροι, αλλά οι λίγοι. Μειώθηκε, μάλλον αυξήθηκε η ανεργία και δυστυχώς είχαμε αύξηση της ανεπίσημης εργασίας των επισφαλών θέσεων εργασίας. Γύρω στο 70% πλέον είναι οι θέσεις αυτές στην Κεντρική Αμερική και αυτές οι συνθήκες, ελεύθερου εμπορίου δεν δημιουργούν αξιοπρεπή εργασία ενώ παραβιάζουν και τα πρότυπα της, παγκόσμια, της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Τα ωφέλη αν υπήρξαν υπήρξαν μόνο και μόνο για τις οικονομικές ελίτ της περιοχής. Έλλειψη ευκαιριών λοιπόν η οποία είχε ως αποτέλεσμα αύξηση της μετανάστευσης και εσωτερικά, δηλαδή από την Ήπεθρο στην πόλη, αλλά και προς το εξωτερικό. Κυρίες και κύριοι μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εμείς λέμε όχι στην επικύρωση αυτής της συμφωνίας για να μπορέσει να αναδιατυπωθεί η συμφωνία αυτή, λαμβάνοντας υπόψη τα όσα μας έχει διδάξει η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Πρέπει να ενισχυθεί η ρύθμιση του εμπορίου και των επενδύσεων, να είναι εγγυημένη η τήρηση των εθνών προτύπων σε ό,τι αφορά τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα και επίσης να υπάρξει σεβασμός για το περιβάλλον και να γίνει δυνατόν να έχουμε μια ευρεία συζήτηση κοινωνική και στις δύο περιοχές. Εμείς εκπροσωπούμε συνεταιρισμούς, μικρούς παραγωγούς, ε, αγροτικές επιχειρήσεις και σας απευθύνουμε έκκληση γιατί έχετε συμβάλει στην ειρήνη και τη δημοκρατία στην Κεντρική Αμερική μέχρι σήμερα. Σας απευθύνουμε λοιπόν έκκληση να μην αφήσετε να το αυτό το έργο και, έργο και το καθήκον για να προωθήσετε πλέον τις δικές σας επιχειρήσεις, ε, το κέρδος σας και να εκμεταλλευτείτε τους φυσικούς μας πόρους. Γι' αυτό παρακαλούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δείξει υπευθυνότητα να δείξει το ανθρωπιστικό, το δημοκρατικό πρόσωπο υπέρ των λαών των χωρών. Σας ευχαριστώ πολύ. Είχαμε καλέσει, καλέσει συγγνώμη, και την Αλήθεια Μπάρθενα από, την ΣΕΠΑΛ, την Οικονομική Επιτροπή για την Λατινική Αμερική, η οποία όμως δεν μπόρεσε να έρθει σήμερα. Είχε όμως την καλοσύνη να μας αποστείλει ένα μήνυμα μέσω βίντεο. Καθώς όμως δεν έχουμε χρόνο, αποφάσισα να το στείλουμε σε όλους εδώ τους παριστομένους ώστε να ενημερωθείτε. Ε, επιστρέφω τώρα στα μέλη της Επιτροπής μας. Και ξεκινώ με τα μέλη της μόνιμης Επιτροπής Κεντρικής Αμερικής. Ακούσαμε τον Παύλο Σάλβα και τον κύριο Λάιφριτ. Ας ακούσουμε τώρα και τους λοιπούς συναδέλφους. Μακλάρκινγκ παρακαλώ. Πρώτη φορά είστε εδώ. Στην Επιτροπή μας. Καλώς ήρθατε. Ναι, Πρόεδρε και σας ευχαριστώ. Είμαι νέο μέλος της Επιτροπής σας. Με χαρά συμμετέχω. Χαίρομαι για την ευκαιρία που έχουμε για τον διάλογο αυτόν σήμερα. Θα ήθελα να απευθυνθώ προς όλους τους εδώ παρκημένους να τους πω ότι άκουσα με ενδιαφέρον τα λόγια σας. Μιλήσατε με πολύ πάθος, με πολύ ενδιαφέρον για τη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, για, την, για τον Επίτροπο. Μια, μια μισή ερώτηση, ύστερα από τα όσα ακούσαμε, αν θεωρεί προσωπικός ότι είναι μάλλον πολιτικό ή οικονομικό, οικονομικό έγραφε αυτή η συμφωνία και ανάλογα με την επιλογή πώς ε, αιτιολογεί αυτή την ε, επιλογή. Επίσης συγκεκριμένε ερωτήσεις για το, για, την, ε, για το εμπόριο αλκοολούχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ήθελε, αν έχει την καλοσύνη ο Επίτροπος να μας πει τι είδους εγγύησεις μπορεί να προσφέρει για την ενθάρρυνση της μεταρρύθμισης διακριτικών μέτρων που ισχύουν σε σχέση με τις χώρες κατεξιμερικής και πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υλοποιήσει την αναγνώριση της προστασίας γεωγραφικής προέλευσης που έχουμε για προϊόντα όπως το ουίσκι σκοτίας. Μια γενική ερώτηση λοιπόν και μια πιο ειδική. Ευχαριστώ πολύ. ECR σημαίνει Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές. Και πάμε τώρα στους πράσινους με τον κύριο Ζαντού. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ σε έλαβαν το λόγο. Ήταν πολύ η παρουσία παρουσιάσει. Και εύστοχα υπόθηκε όταν παρουσιάζεται μια συμφωνία, ε, ιδιαίτερα από αυτού που την έχουν υπογράψει. είναι εντύπωση ότι όλοι κερδίζουν πολλά χρήματα, κερδίζουμε μεγάλη ανάπτυξη, ε, πλεονεκτήματα για όλους. Όμως η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Δεν θα ισχυριστώ βεβαίω ότι θα χάσετε από την συμφωνία αυτή, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι το όφελο συνοδεύεται και από τίμημα. Θα ήθελα λοιπόν από πλευρά ιδιαίτερω των εκπροσώπων των κρατών τη Κεντρική Αμερική που εκπροσωπούν χώρε που βρίσκονται σε οικονομικέ δυσχέρειε, που έχουν προβλήματα και κοινωνική οικονομία και οικονομικά οι πολιτικά να μας πούν πώς σκοπεύουν να χειριστούν το θέμα του τιμήματος, του κόστους που συνεπάγεται αυτή η συμφωνία. Φερρυπίν, ποσοστό στα γαλακτοκομικά. Αυτή η ποσόστοση μάλλον είναι των γαλακτοπαραγωγών της Ευρώπης θα αποβεί παρά εκείνων της Κεντρικής Αμερικής ή στην πρόσβαση, η δυνατότητα πρόσβασης ε, ε, στις αγορές για τις μέσες Ε, Ο τωρινός πρόεδρος της Γαλλίας, φιλελεύθερος φιλελεύθερο ε, και υποψήφιος και πάλι για τις εκλογές, ο ίδιος λέει ότι θα προστατεύσει τις αγορές του, ότι θα τις κλείσει ουσιαστικά. Εσείς, Κεντρική Αμερική, τι θα κάνετε, πώς θα προστατεύσετε τις αγορές σας. Είπατε επίσης και ιδιαίτερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οφείλετε να αναφέρετε το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του περιβάλλοντος, ε, των, τα κοινωνικά. Ερωτώ λοιπόν πώς μπορείτε να αιτιολογήσετε στον πολίτη σας. Πώς θα αιτιολογήσετε λοιπόν στον πολίτη σας τις διαφορές αυτές, γιατί βεβαίως δεν μπορούμε πάντα να υπάγουμε ε, στις, στο οικονομικό συμφέρον τα μελήματα τα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, το περιβάλλον, τα κοινωνικά θέματα πρέπει και αυτά να έχουν τη θέση τους. Ένα τελευταίο σχόλιο, Παύλα, ερώτηση για τον Επιτροπό Ο Παναμάς. Ο Παναμάς θεωρείται λίγο πολύ φορολογικός παράδεισος. Τις διαπραγματεύσεις του Παναμά πώ τις χειριστήκατε. Βλέπουμε ότι μέσα στις, στη συμφωνία προβλέπεται, η, επαναβεβαιώνεται μάλλον η διαφύλαξη του τραπεζικού απορρίτου. Αυτό συνεπάγεται δηλαδή ότι είναι σε θέση να με αυτή τη συμφωνία η Ευρωπαϊκή Ένωση να ζητήσει από τον Παναμά να άρει το απόρριτο των τραπεζικών συναλλαγών. Ευχαριστώ πολύ. Σόλτ, Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πολλά πράγματα μπορούμε να συζητήσουμε ή θα οφείλαμε να συζητήσουμε σήμερα. Δεν έχουμε πολύ χρόνο όμω. Και γι' αυτό θα επικεντρωθώ σε ορισμένα και ουσιώδη στοιχεία. Η τα κοινωνικά, τα πολιτικά, τα οικονομικά δεδομένα τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στις χώρες της Κεντρικής Αμερικής. Πρέπει ασφαλώς να αποτελέσουν την λιδία λίθο για την αξιολόγηση της επιτυχούς υλοποίησης μιας συμφωνίας όπως η παρούσα. Γι' αυτό απευθύνω πρώτα στον Επίτροπο μια ερώτηση, διότι και εμείς βεβαίως θα πρέπει να ενημερώσουμε και να, προ... να παρουσιάσουμε την συμφωνία αυτή στον πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να του εξηγήσουμε γιατί πρέπει να την συνάψουμε. Πώς θα εξηγήσω λοιπόν σε έναν Έλληνα, Ισπανό, Πορτογάλο πολίτη μέσα σε αυτή τη δίνη της μεγάλης ευρωπαϊκής κρίσης τα πλεονεκτήματα αυτής της συμφωνίας όταν ε, η Σύνοδος Κορυφής του G20 έχει προ... αποφασίσει περισσότερη διαφάνεια για τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Και ως εκ τούτου, εγώ βρισκόμαι σε μια δύσκολη θέση, διότι αυτή η συμφωνία εισάγει μάλλον την αντίθετη τάση από αυτά τα οποία είχε προβλέψει η G20 ή αντίστοιχα διαδικασίες και νομοθετήματα που ε, προχωρούν μέσα από τις διαδικασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έτσι λοιπόν, Ε, αυτό δεν προβλέπεται παραδείγματι στο άρθρο 95 παράγραφο 3. Η, δε, για δε εκπροσώπους των κρατών της Κεντρικής Αμερικής έχω κάποιες ερωτήσεις επίσης. Στην ε, συμφωνία ε, προβλέπονται ειδικέ διατάξεις ε, για το αραχιδέλαιο, για το φινικέλαιο, για τα αλκοολούχα και τη ζάχαρη. Έχετε συνειδήσει τι είδους συνέπειες μπορεί να φέρει ως προς την παραγωγή τροφίμων, γεωργική παραγωγή τροφίμων, ως προς ε, την, ε, τις συνθήκες, τις περιβαλλοντικές και τέλος προς τους ενδογενείς πληθυσμούς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κύριε Επίτροπε, θα επενδύσει για να ενισχύσει τις εξαγωγή, το εξαγωγικό δυναμικό της Κεντρικής Αμερικής. Υπάρχουν κάποιες μελέτες ε, στον τομέα αυτόν ή αφήνεται την ανάπτυξη των εξωτερικών, του εξωτερικού αυτού εμπορίου στη μοίρα της, στα χέρια μας περιπτώσει των, των κρατών της Κεντρικής Αμερικής. Για δε τη Γουατεμάλα έγινε μια σύνοδος κορυφής, όπου ο πρόεδρος Γουατεμάλας πρότεινε την νομιμοποίηση του εμπορίου ναρκωτικών με την Λατινική Αμερική και σε αυτό εμπλέκεται και το Μεξικό. Έχετε καμιά συνείδηση των συνεπειών καταστροφικών συνεπειών που θα έχει αυτή η νομοποίηση του εμπορίου ε, ναρκωτικών. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάποια πρόθεση να φροντίσει ώστε παιδιά που θα έχουν τελειώσει το σχολείο και που κινδυνεύουν από τα καρτέλ των ναρκωτικών να βρουν μία διέξοδο, γιατί δεν υπάρχει ούτε θέση εργασίας, ούτε κοινωνική πλαισίωση το ΣΥΠΗΝ. Άρα πάλι βρίσκονται εκτεθειμένα στα καρτέλ των ναρκωτικών τα νεαρά αυτά παιδιά. Η δεν νομοποίηση των ναρκωτικών είναι ο σωστός δρόμος, είναι μια προσέγγιση θεμητή. Ή, εν πάση περιπτώσει, διμερός, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς θα το αντιμετωπίσει το ζήτημα αυτό. Δεν έχει αυτό επίπτωση και στη συμφωνία, ε, την εμπορική συμφωνία με την Κεντρική Αμερική. Αυτά προς το παρόν στις προς Μάλιστα, ο Επίτροπος ε, δεν ξέρω αν αντελήφθη την πρώτη σας ερώτηση, κύριε Σόλτς. Κύριε Σόλτς, δεν κατάλαβα τι είπατε. Για πρώτη ερώτηση Είπατε ότι θα μου κάνετε μια ερώτηση, αλλά μάλλον δεν την κατάλαβα. Θέλετε να επαναλάβετε. Το G20 έχει στήσει περισσότερη διαφάνεια και ενίσχυση των οργανισμών επιτήρησης και ρυθμιστικών φορέων. Το 159 παράγραφος 3, 195 παράγραφος 3, ε, προτείνει ακριβώς το αντίθετο από τις κατευθύνσεις που έχει δώσει η G20. Δεν θα επιτρέπει δηλαδή έλεγχο ροής κεφαλαίων. Ή τα κεφάλαια θα, θα παρακολουθούνται δυνάμει των νόμων της χώρας υποδοχής. Δεν αποτελεί αυτό αντίφαση με τη συμφωνία του G20. Και αντίστοιχα με κατευθύνσεις που εμείς Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με άλλες χώρες του G20 λαμβάνουμε ε, στα θέματα των διεθνών συναλλαγών. Καλώς λέει ο πρόεδρος. Η κυρία Μπίρντερ από, την, από τους φιλελευθέρους. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ξέρω ότι δεν έχουμε χρόνο και πρέπει να ακούσουμε και τις απαντήσεις βεβαίως. Θα είμαστε δυνατόν πιο σύντομοι και ότι είναι πολλά τα σημεία που θα ήθελα να διατυπώσω. Ο Όλμαρ έκανε μια πολύ εύστοχη παρατήρηση, εάν είναι οικονομική δηλαδή, ή έλμα μάλλον, αν είναι ε, οικονομική ή πολιτική συμφωνία περισσότερο, γιατί προσπαθούμε ποτέ να βοηθήσουμε και την ε, ολοκλήρωση των κρατών αυτών, άρα έχει μάλλον πολιτικό χαρακτήρα, αλλά βλέπω ότι προσεγγίσουμε από την οικονομική σκοπιά. Ε, επίσης με χαρά άκουσα ότι ο Επίτροπος ε, βλέπει και καλή προστασία του περιβάλλοντος μέσα από τη συμφωνία αυτή να προκύπτει. Σήμερα είχα το μεσημέρι συνάντηση με περιβαλλοντολόγους από την πατρίδα μου, από το Ηνωμένο Βασίλειο και στην εκδήλωση αυτή ένα 12χρονο κορίτσι σηκώθηκε, πήρε το λόγο και μας εξέφρασε τις ανησυχίες που έχει για τον κόσμο που θα μεταδώσει, που θα παραδώσει στα δικά της παιδιά και ήταν μόνο 12 ετών. Μας μίλησε για τον πλανήτη, μας μίλησε για την αναζήτηση τροφίμων στην ε, κοντινή περιοχή, να μην ταξιδεύουν τα φρούτα από την μια, από την μια άκρη του κόσμου στην άλλη, να μην ε, καταναλώνουμε δηλαδή κατά τρόπο μη βιώσιμο μία αηφόρο. Το χρειαζόμαστε το εμπόριο, ναι, και εγώ το θέλω. Αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να δώσουμε απάντηση στα, α, στις ανησυχίες των δεκάχρονων παιδιών, όχι μόνο εδώ στην Ευρώπη, αλλά και της Κεντρικής Αμερικής και να εξηγήσουμε τι κάνουμε στον πλανήτη μας. Έχουμε βεβαίω ρήτρε βιώσιμη ανάπτυξη. Ε, μιλάμε πάντα για βιώσιμη ανάπτυξη, αηφόρο ανάπτυξη και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά τι σημαίνει τελικά όλο αυτό, γιατί και σε προηγούμενη ακρόαση είχαμε το ερωτηματικό του τι σημαίνει αηφόρο ανά ανάπτυξη στην Ευρώπη και τι μπορεί να σημαίνει φερειπέ στη Γουατεμάλα. Γι' αυτό λοιπόν ακριβώ αυτό θα πρέπει να συζητήσουμε σε μια ιδιαίτερη ακρόαση, τι σημαίνει αηφόρο ανάπτυξη. Γιατί διαρκώ επαναλαμβάνουμε τη φράση αυτή, αλλά πρέπει και να αντιληφθούμε τι συγκεκριμένα ε, περιλαμβάνει. Και επίση με χαρά βλέπω ότι υπάρχουν δεσμευτικέ ρήτρε για τη συμμετοχή τη κοινωνία των πολιτών, ρευτόρια πράγματα. Αλλά έχουμε εδώ ω βουλευτέ στην Ευρώπη την αντίληψη ότι η, κοινωνία, η, τη βεβαιότητα αυτή η κοινωνία των πολιτών είναι πράγματι μια ελεύθερη κοινωνία των πολιτών. Για, με τον Καναδά, Φερρυπίν, ξέρουμε ότι υπήρχαν κάποιες συγκεκριμένες ρήτρε που ε, σε σχέση με τον Παναμά ε, περιόριζε πολύ τις, ε, τις δυνατότητες συμμετοχής κοινωνίας των πολιτών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι γνώμη έχει γι' αυτό και πώς μπορούμε να το καλύψουμε. Επίσης, Στην Ευρώπη έχουμε πολλές φορές διεπενδυτικά μέτρα επιθετικά που νομίζω ότι θα πρέπει να ρυθμίσουμε οι επιχειρήσεις μας δηλαδή που αναλαμβάνουν δράση σε τρίτες χώρες δεν μπορεί να, να μετέρχονται τέτοια μέσα. Η κοινωνική ε, ευθύνη των επιχειρήσεων είναι μια αρχή πάρα πολύ σημαντική, αλλά πέραν αυτού πρέπει να προστατεύσουμε και ε, τι επιχειρήσει εκείνε ή του φορεί εκείνου μικρή κλίμακα, του παράγοντε μικρή κλίμακα, από του οποίου έγινε λόγο και νωρίτερα, ε, έναντι των ε, μεθοδεύσεων που αναπτύσσονται από ορισμένους επιχειρήσεις να αναπτύσσουν τις δραστηριότητες τους σε περιοχές του κόσμου όχι τόσο προηγμένες ως προς τις μεθόδους εξαγωγής, παραγωγής και ούτω καθεξής. Εκεί ούτω καθεξής. Αυτή είναι η κοινωνική ευθύνη που πρέπει να πετύσουν από τις επιχειρήσεις μας, όχι για μας εδώ στην Ευρώπη, ούτε ε, στην Κεντρική Αμερική, αλλά για τα 12 χρόνια εδώ τη Ευρώπη και τη Κεντρική Αμερική. Ευχαριστώ και τώρα σε ακούσουμε τον κύριο Σολαφράνκα, που χωρί να είναι τη Επιτροπής μας είναι πάντα ευπρόσδεκτο και ο οποίο είναι εισηγητή τη Επιτροπή των Εξωτερικών Υποθέσεων για την ίδια αυτή ε, συμφωνία. Κύριε Σολαφράνκα, έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρο. Ω εισηγητή ε, τη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων θα ήθελα να σας πω ότι πρόκειται για μια συμφωνία σύνδεσης Πρώτα απ' όλα, σημαίνει ότι θα παίξουν στην πρώτη εθνική οι χώρες της Κεντρικής Αμερικής την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως το Μεξικό και η Χιλή. Είναι συνεκτική η ε, συμφωνεί αυτή με όλα τα ψηφίσματα που εγκρίναμε και με την απόφαση των 27 και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και κυρίως μας επιτρέψει να περάσουμε στην όριμη ηλικία σχέσεων που έχουν περάσει από εκχωρήσεις μονομερείς εκκριτικές, ενώ εδώ τίθενται οι βάσει βάσεις για και τα θεμέλια για ισότιμες σχέσεις. Είναι λοιπόν σημαντικό και θα το πω ότι λαμβάνει υπόψη η, τις αυτή η συμφωνία, διότι προβλέπει την χρονοδιάγραμμα βάσει των οποίων με κάποιες εξαιρέσεις θα εισέλθουν όλα τα προϊόντα της Κεντρικής Αμερικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το να πούμε ότι δεν προβλέπονται οι ασυμμετρίες, κύριε Πρόεδρε, για την άποψή μου, σημαίνει ότι το πρωτεύον το συγχαίουμε με το δευτερεύον και ε, δεν βλέπουμε ποια είναι τα σημαντικά στοιχεία αυτής της συμφωνίας. Πρώτα απ' όλα, ό,τι έχει γίνει, έχει γίνει βασιζόμενο στι αρχές που διέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, όταν θα γίνουν ανταγωνιστικές και θα μας παρουσιάσουν νέα προϊόντα οι χώρε της Κεντρικής Αμερικής, δεν θα μπορέσουμε να κλείσουμε τις θύρε. Όσον αφορά τη δημοκρατική ρήτρα, νομίζω ότι αποτελεί βασικό στοιχείο όλων των συμφωνιών και οι εκπρόσωποι των χωρών αυτών που ε, διαπραγματεύτηκαν την συμφωνία με τους 27 ξέρουν ότι είναι αυτοί οι οποίοι εμφανίζονται και στις υπόλοιπες ε, συμφωνίες. Η ρήτρα η δημοκρατική δεν θα πρέπει κύριε Πρόεδρε να ερμηνεύεται με παρτεναλικό παρτερναλιστικό τρόπο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οτιδήποτε γίνει και ό,τι συναυθεί γίνεται βάσει της αμοιευότητας και είναι υποχρεωτικό για τα δύο μέρη. Εγώ θα ήθελα να κάνω την ίδια ερώτηση που έκανα και στον ε, ε κύριο Ντεγκούχτου και θα φύγω σε λίγο διότι έχω μεγάλη συνάντηση στην Επιτροπή μου. Πρόκειται για την καθυστέρηση που υπάρχει εδώ για την επικύρωση. Πέρασαν δύο χρόνια και αυτό είναι κάτι το οποίο πλήττει την αξιοπιστία τη Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουμε είναι από κοινού να σκεφτούμε, κύριε Επίτροπε, πώ η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να μειώσει τέτοιου είδου προθεσμίε ώστε ε, να προχωρήσουμε χωρίς βεβαίως να το κάνουμε αυτό εις βάρος του εξαιρετικού τρόπου με τον οποίο εργαζόμαστε. Εγώ αυτή είναι η πρόταση που θα κάνω στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, κύριε Πρόεδρε. Ξέρετε, επίση πρέπει να σα πω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να αλλάξει ούτε ένα κόμμα σε σχέση με αυτά που συμφώνησαν 27 με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά βεβαίω στο δικό μα το ψήφισμα ε, θα πούμε ότι πρόκειται για συμφωνία η οποία προάγει τα αμοιβαία συμφέροντα και ημών και ημών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Thank you very much. Before I give the floor to Pablo Thalba to close. Πρέπει να δώσω το λόγο στον κύριο Θάλμπα για να κλείσουμε τη συζήτηση αυτή. Θα δώσω το λόγο στον Επίτροπο Ντεγκούχτ για να απαντήσει σε κάποιες ερωτήσεις που του έθεσαν τα μέλη απευθείας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ναι, έχετε δίκιο. Έχω την εντύπωση ακούγοντα του ε, βουλευτέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι πριν να διαπραγματευτούμε μια συμφωνία ε, εμπορίου με μια τρίτη χώρα, απαιτείται να μεταρρυθμίσουμε την ίδια τη χώρα. Και μόνο μετά μπορούμε να συνάψουμε εμπορικέ σχέσει μαζί της. Αυτό ε, προκύπτει, φαίνεται να προκύπτει από τις ε, παρεμβάσει ορισμένων εξημών. Φυσικά αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Αυτό που κάνουμε τις συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών είναι ότι ορισμένες αρχές εδρεωμένες μέσα στη συνθήκη πρέπει να γίνονται σεβαστές. Έχουμε κεφάλαιο σχετικά με την αηφορία. Έχουμε και άλλες δυνατότητες. και δυνατότητες να αντιδράσουμε όταν τα πράγματα πάνε ε, προς τη λάθος κατεύθυνση. Αλλά δεν μπορείτε να απαιτείτε να ε, μεταρρυθμίσουμε ολόκληρο τον κόσμο κατά το δικό μας πρότυπο πριν να ξεκινήσουμε η αδίποτε ε, οικονομική συνεργασία με τις άλλες χώρες. Αυτή την εντύπωση τουλάχιστον μου δίνουν οι παρεμβάσεις που ακούω όταν έρχομαι εδώ. Εν πάση περιπτώσει όμως δεν μπορεί αυτό να ε, συνεπάγεται ότι δεν είναι η, μια τέτοια χώρα παράγων που προάγει το εμπόριο. Από την άλλη δεν μπορούμε να πάμε και σαν πειρατές που θα ε, απομυζήσουν όλα τα πλούτη μιας άλλης περιοχής. Εμείς ε, σεβόμαστε πάντα την ε, αλυσίδα της ε, παραγωγής, της προμήθειας, αλλά από την άλλη πρέπει πάντα να διατηρείται μια λεπτή ισορροπία όχι όμως υπό την έννοια που προβάλλουν ορισμένοι σήμερα για κάποιες ειδικές ε, για κάποια ειδικά θέματα, φέρνει του κυρίου Ζαντού, στο θέμα των ε, φόρων. Πρόκειται για μια συμφωνία σύνδεσης που δεν καλύπτεται στο εμπορικό κομμάτι. αλλά μάλλον στις οικονομικές πτυχές και συμφωνίας. Και πέραν τη συμφωνία συνδέσεως πρέπει να επισημάνω για τον Παναμά ειδικέτερα ότι είναι σε διαδικασία υπογραφή συμφωνίας για την αντιμετώπιση της διπλής ε, φορολόγηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντιμετωπίζεται λοιπόν το ζήτημα που επισημαίνεται, αλλά όχι μέσα σε αυτή τη συμφωνία. Ένα άλλο ζήτημα για τα ωφέλη που αποκομίζει από τη Συμφωνία Σύνδεση Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσπάθησα να το εξηγήσω στην παρουσίασή μου. Δεν νομίζω να μου επιτρέψει ο πρόεδρο να επαναλάβω τα ίδια λόγια. Ιδιαίτερα όμω για το ουίσκι που φαίνεται να ενδιαφέρει ιδιαίτερα την κυρία Μακλάρκιν. Ο Παναμάς είναι κύριος αγωγέας ουίσκι από την περιοχή. 70% του ουίσκι προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, φαντάζομαι το μεγαλύτερο κομμάτι από τη Σκωτία, και θα ε, απελευθερωθεί το εμπόριο αυτό, άπαξ και τεθεί σε ισχύ η συμφωνία. Και οι άλλες αντίστοιχα χώρες Κεντρικής Αμερικής θα απελευθερώσουν τις δικές τους αγορές έξι χρόνια αργότερα, όπως προβλέπεται στη συμφωνία. Πριν να τεθεί σε προσωρινή εφαρμογή συμφωνία, αλλάζει όχι μόνο η νομοθεσία σχετικά με τη κανόνες προελεύσεως, αλλά και η υλοποίησή της. Προσωρινή υλοποίηση, όπως και να έχει, δηλαδή από την κύρωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μιας συμφωνίας μπορεί να αρχίσει η εφαρμογή. Αυτό προβλέπεται. Στη σχέση μας με τους ε, εταίρους από την Κεντρική Αμερική. Πρόβλημα λοιπόν με το χρόνο δεν βλέπω. Εν τω μεταξύ όμως βλέπω ότι ο κύριος Σαλαφράγκα έχει αποχωρήσει. Φαίνεται ότι ήταν στενά τα χρονικά περιθώρια. Μα, το κύριο πρόβλημα πάντω είναι η μετάφραση πάντα σε αυτές τι περιπτώσεις. Είναι ογκώδει συμφωνίε, χιλιάδε σελίδε πολλέ φορέ και πρέπει να μεταφραστούν στι 23 επίσημε γλώσσε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πράγμα το οποίο πριν από την κύρωση νομίζω δεν έχει κανένα νόημα. Πρέπει ούτω ή άλλω κάποια στιγμή να μεταφραστούν σε όλε τι γλώσσε οι συμφωνίε, φερειπίν διότι θα πρέπει να υλοποιηθούν από τις τελωνιακές αρχές. Αλλά τότε επιλεκτικά γίνεται μετάφραση μόνο των ε, σχετικών κεφαλαίων. Ιδάλλως, η συνολική μετάφραση ολόκληρων των κειμένων ε, θα σήμαινε ε, τουλάχιστον ενός έτους καθυστέρηση. Οπότε θα είχε κανένα νόημα. Φυσικά αυτό μπορεί να το αλλάξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμείς δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Το έχουμε πει στο συμβούλιο, σας το λέμε και σε εσά κάθε φορά που αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα αυτού του χρόνου, ότι πιστεύουμε πως θα πρέπει να δοθεί μια διαφορετική λύση. για το εμπόριο και την ε, βιώσιμη ανάπτυξη, το σχετικό κεφάλαιο θεσπίζει διαφανείς και πλήρης ε, εκτεταμένους μηχανισμούς διαιτησίας που μπορεί μονομερός να θέσει λειτουργία το ένα συμβαλλόμενο μέρος και που άπαξ και σε λειτουργία ακολουθούν συγκεκριμένε προθεσμίες και χρονοδιάγραμμα και άρα μπορεί όντω να τεθεί σε λειτουργία στους μηχανισμούς όπως προβλέπετε και στη συμφωνία με την Κολομβία. Θα ήθελα εν τέλει πρόεδρε να κάνω μια παρατήρηση Εγώ είμαι υπέρ αυτής της συμφωνίας, κύριε Πρόεδρε, κυρίως διότι αποτελεί ένα πρώτο υπόδειγμα συμφωνίας εμπορικών συναλλαγών μεταξύ μιας όριμης οικονομίας αφενός και αφετέρου ορισμένων λιγότερο όριμων οικονομιών, κάποιων μόλις, ε, μόλις αρχίζουν να οργανώνονται και άλλες είναι αναπτυσσόμενες ή λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Άρα βεβαίως και χρειάζονται οι όροι του ισότιμου εμπορίου, στο οποίο ασφαλώς θα διδραματίσει το ρόλο του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από την άλλη, αν κοιτάξουμε τα αποτελέσματα που μας προσφέρει το εμπόριο και τα συγκρίνουμε με τα άλλα αποτελέσματα της ε, α, λυπής της προσπάθειας, τότε ασφαλώς μπορούμε να πούμε ότι είναι σημαντικά και αυτά. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο θα ήθελα να σας δώσω, ελπίζοντας ότι θα κυρώσετε τη συμφωνία σύνδεσης του ταχύτερο δυνατό. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι είναι πολύ σωστό και δίκαιο να δώσω το λόγο και στην άλλη πλευρά, του εκπροσώπου των χωρών της Κεντρικής Αμερικής, για να απαντήσουν στα σχόλια που έκαναν οι διάφοροι ενδιαφερόμενοι για τη συμφωνία. Ο κύριος ε, από την Ονδούρα Μέλμιν Ρεδόντο, υπουργό εδώ, που είναι και προσωρινός πρόεδρος ε, του ΣΥΚΑ, θα πάρει το λόγο για να εκπροσωπήσει ουσιαστικά όλη την περιοχή. Κύριε Φιπουρή, έχετε το λόγο για λίγα λεπτά. Να μπορέσετε να απαντήσετε στα σχόλια των ε, διαφόρων ε, εμπλεκομένων φορέων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Φυσικά και σημειώσαμε όλες τις παρατηρήσεις, τις συστάσεις και τις απόψεις που ακούσαμε σήμερα το απόγευμα στην ακρόαση αυτή. Αναμφίβολα θεωρούμε ότι φαίνεται ξεκάθαρα από όλε αυτέ τι δηλώσει ότι είναι ανάγκη να συζητήσουμε σε μεγαλύτερο βάθος ορισμένα από τα θέματα, αλλά φαίνεται επίση ότι υπάρχει και η βούληση να οριοθετηθεί η συμφωνία αυτή ότι είναι μια συμφωνία οικονομική, πολιτική, συμφωνία συνεργασίας που θα ανοίξει τις πόρτες ε, για έναν ε, πιο πλούσιο χώρο συζητήσεων. Οι απόψεις που εξέφρασαν σήμερα οι φίλοι μας από την κοινωνία των πολιτών, αυτό που δείχνουν ακριβώς είναι ότι έχουμε φτάσει σε ένα στάδιο οριμότητας, όπου πλέον είναι δυνατή η ελεύθερη έκφραση και η ελεύθερη κριτική και επισήμανση των προβλημάτων τα οποία θα πρέπει να επιληθούν. Όλα αυτά τα σημειώνουμε όπως και την ανάγκη να έχουμε πολύ ξεκάθαρους μηχανισμούς για την υλοποίηση της Συμφωνίας Σύνδεσης στην Κεντρική Αμερική ώστε να διορθωθούν ή να απαλληφθούν αυτά τα προβλήματα που μας επισημάνατε και από την ευρωπαϊκή πλευρά και από την πλευρά της Κεντρικής Αμερικής. Νομίζω ότι είναι συνετό και σκόπιμο να αναφέρουμε ότι ο δρόμος που έχουμε διανύσει μέχρι τώρα είναι θετικός. Είναι μεγάλες προκλήσεις. Αυτό το δείχνουν ε, και τα σχόλια που ακούσαμε σήμερα. Η οικονομική ανάπτυξη δεν μπορεί να υπάρχει αν δεν συνοδεύεται από κοινωνική ανάπτυξη και η κοινωνική βιωσιμότητα χωρίς οικονομική ανάπτυξη είναι επίσης αδύνατη. Η Συμφωνία Σύνδεσης ε, είναι μια πολύτιμη συνεισφορά σε αυτή την ολοκληρωμένη ανάπτυξη, με σταθερότητα και με δημοκρατία. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε κάτι το οποίο αναφέραμε προηγουμένως, δηλαδή ότι η συμφωνία δεν πρέπει να θεωρηθεί ως ένα εργαλείο το οποίο θα επιλύσει όλα τα προβλήματα που ακούσαμε σήμερα. Είναι όμως ένα μέσο που πράγματι με τη δημιουργία νέων χώρων, πολύ καλό και καθορισμένων που χαιρετίστηκαν άλλωστε από όλους τους συμμετέχοντες, αυτό θα συνεισφέρει στο να, να βελτιώσουμε και να τελειοποιήσουμε τη συμφωνία, να θέσουμε όλα τα προβλήματα και να τα αντιμετωπίσουμε. Αυτό το οποίο ανοίγει ουσιαστικά η συμφωνία είναι ένα παράθυρο ελπίδας, μια ευκαιρία για να δούμε και εμείς και να μάθουμε ε, από τους Ευρωπαίους ε, εταίρους πώς λύθηκαν ή πώς λύνονται τα προβλήματα και πώς μπορεί, και πιστεύω ότι είναι ένας κοινό ε, τόπος συζήτησης για να βρούμε λύσεις που θα οδηγήσουν σε ένα καλύτερο μέλλον και για τις δύο περιοχές. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω όλους τους εισηγητές, όλους όσους έλαβαν το λόγο για τις παρεμβάσεις τους γιατί έθεσαν το δάκτυλο επί των τύπων των ύλων επί προβλημάτων τα οποία θα πρέπει στο επόμενο στάδιο τη ολοκλήρωση των σχέσεων Ευρωπαϊκή Ένωση και Κεντρική Αμερική να φύγουν. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ για να ολοκληρώσουμε αυτή την ακρόαση. Θα δώσω το λόγο για μια ακόμη φορά στον δικό μα εισηγητή, τον Παύλο Θάλμπα, που δεν είναι απλά μόνιμος εισηγητή για τι σχέσει μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Κεντρική Αμερική, αλλά και ειδικότερα εισηγητή για τη συμφωνία αυτή συμφωνία σύνδεσης που περιλαμβάνει ένα ευρύτατο φάσμα Συμφωνία Εμπορικών Συναλλαγών που όπως είπε και ο Επίτροπος είναι κεντρικός πυλώνας της συμφωνίας. Παύλο Θάλμπα, έχει το λόγο για να κλείσει τη συζήτηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Ντεγκού, κύριε Επίτροπε, και εγώ συμμερίζομαι αυτά που είπατε για την σημασία που έχει αυτή η συμφωνία σε όλους τους τομείς, αλλά και το μέλημα που εξέφρασε ο κύριος ε, ε, Σαλαφράγκα. Τι γίνεται από την υπογραφή μέχρι τη στιγμή που φτάνει σε εμά η συμφωνία. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει το πρόβλημα το γλωσσικό που είναι δύσκολο και κατανοώ επίσης το ότι αυτό δεν είναι κάτι που έχει αντίκτυπο αρνητικό, αλλά στην περίπτωση του Περού και της Κολομβίας έχει σημαντικές επιπτώσεις και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων επίσης ανέφερε κάποια θέματα, γιατί θα ήθελα να γίνουν τα πράγματα μεγαλύτερη ταχύτητα. Τώρα όσον αφορά την συμφωνία αυτή, πιστεύω ότι η μελέτη της ε, London School of Economics μας είπε είναι, ποια θα είναι τα ωφέλη. Και η Business Europe σύσσωμα υποστηρίζει αυτή τη συμφωνία που θα είναι επωφελής οπωσδήποτε για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη και βεβαίως θα δημιουργήσει και εδώ σε εμά θέσεις απασχόλησης. Σημερίζομαι την ανάλυση του Επιτρόπου, ο οποίος λέγει ότι η στρατηγική Trade for Growth θα αποφέρει ωφέλη όχι μόνο στους εμπορικού μας εταίρους, αλλά κυρίως και στην ευρωπαϊκή οικονομία. Τώρα, όσον αφορά τα θέματα τα οποία συζητήσαμε εδώ σήμερα το απόγευμα, θα ήθελα να ταινίσω κάποια από αυτά. Το ΣΕΧΕΧΕΠ πρέπει να είναι ένα ε, ένας από τους λόγους για τους οποίους θα πρέπει να υπογραφεί το συντομότερο δυνατό η συμφωνία αυτή διότι αυτό ανταποκρίνεται στις προσδοκίες όλων μας, όχι μόνο και του δικού μας Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Ευρωπαϊκών Κοινοβουλίων, αλλά και τις ε, ε, προσδοκίες όλων των κοινοβουλίων των κρατών της Κεντρικής Αμερικής. Για να απαντήσω στον κύριο Χουάν Μορένο και αυτά τα οποία είπε για την καταστρατήγηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Βεβαίως η κατάσταση δεν είναι τέλεια σε καμία περιοχή του κόσμου. Εξάλλου αυτά τα προβλήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να τα δούμε μέσα στην προοπτική τους. Και νομίζω ότι ούτω ή άλλω Υπάρχει βελτίωση του τομέα αυτό στι περισσότερε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και στην συμφωνία υπάρχει και μια ρήτρα που αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, πράγμα που θα αποτελέσει κίνητρο για τη βελτίωση τη κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλη την περιοχή. Είμαι σίγουρο ότι η συμφωνία αυτή θα βοηθήσει την ε, βελτίωση τη κατάσταση όλων των εργαζομένων των κρατών τη Κεντρική Αμερική. Σύμφωνα με μελέτε, αναφέρεται ότι τα ευρωπαϊκέ επιχειρήσει που ε, δραστηριοποιούνται στην Λατινική Αμερική προσφέρουν καλύτερες εργασιακές συνθήκες από τις τοπικές επιχειρήσεις. Άρα θα διευκολύνει η συμφωνία αυτή την εγκατάσταση πολλών ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στις χώρες Κεντρικής Αμερικής και θα βοηθήσει την βελτίωση των κοινωνικών και εργασιακών ε, συνθήκων για τους εργαζόμενους της Λατινικής Αμερικής. Σε σχέση με αυτό το οποίο η κυρία Ρεβέκας για την επιχείρηση μέσα συμφωνώ ότι ο τομέας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχει πολλές δυνατότητες ανάπτυξης. Και εδώ η ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ κρατών είναι σημαντική για να μπορέσει να αναπτυχθεί περαιτέρω η χρήση αυτών των ενεργειών. Άρα η... αυτό είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει περισσότερο την ε, περιοχή της Κεντρικής Αμερικής. Και ο τομέας αυτός θα βοηθήσει την περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής ώστε να υπάρξει και πράσινη ενέργεια σε μεγαλύτερο ποσοστό στις χώρες αυτές, σε σχέση με την κυρία Κρούθ, που έλεγε ότι αυτό το πρότυπο θα αποτελέσει ένα πρότυπο φρούτων, λαχανικών και καρυδιών μόνον, νομίζω ότι η συμφωνία αυτή δίνει την δυνατότητα να υπάρχει διαφοροποίηση των διαφόρων προϊόντων που θα συμπεριληφθούν σε αυτή τη συμφωνία και που καλύπτει τα προϊόντα τα οποία παράγουν οι χώρες αυτές και θα βοηθήσει και περαιτέρω εξαγωγές προϊόντων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε αυτή τη συμφωνία. Αναφέρθηκε επίσης ο σημαντικός τομέας της ηλεκτρονικής, τον microchip. Και πιστεύω ότι εδώ μπορεί να υπάρξει μεγάλη ευκαιρία για ανάπτυξη οικονομίας. Τελικά. Θα ήθελα να επαναλάβω ότι είμαι πεπισμένο ότι αυτή η συμφωνία αποτελεί δυνατότητα ενίσχυση τη κοινωνική συνοχή στην περιοχή αυτή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους όσους συμμετείχαν στην ακρόαση αυτή. Ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου τώρα να ευχαριστήσω όλος ιδιαίτερος τους προσκεκλημένους μας, όχι μόνο τους ανεξάρτητους ομιλητές, αλλά ιδιαίτερος τους ομιλητές τη τις χώρες Κεντρικής Αμερικής. Πρέπει να σας πω ότι είμαστε πάρα πολύ περήφανοι τη δυνατότητα που έχουμε να κάνουμε τέτοιου είδους συζητήσεις. Να ανοίξουμε το βήμα σε εκπροσώπους εμπορικούς. Και βεβαίως είμαστε οι καλύτεροι σε θέματα ανοιχτού πνεύματος και διαφάνειας. Ό,τι γίνεται στο Κοινοβούλιο γίνεται μέσα αυτό το πνεύμα. Σας ευχαριστώ πολύ που μας φωτίσατε για τα θέματα που σας απασχολούν. Τελείωσε η συζήτηση τώρα όσον αφορά την εμπορική συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την κεντρική, ε, χώρες Κεντρικής Αμερικής και προχωρούμε στην κανονική μας ημερήσια διάταξη. Please, uh, those who are in the room, uh, Uh, Παρακαλώ να αποχωρήσετε στο δυνατόν πιο γρήγορα και αθόρυβα. Έχουμε πολύ ακόμα δουλειά σήμερα εδώ. Please, uh, distinguished guests, uh, you were, you were invited to speak, not to stay. Μπορείτε να μιλάτε λάβετε το λόγο μάλλον στο επόμενο κομμάτι της συνεδρίασης, αλλά όχι όρθιοι μέσα στην αίθουσα. Ah. Yes, yes. Yes. Thank you. Please do not take advantage of my soft and weak voice. Παρακαλώ, μην εκμεταλλεύεστε την καλοσύνη μου και την κλικιά φωνή μου. Είστε έτοιμοι για το κεφάλαιο 31 της Μεσής Διάταξης. Κεντρική Αμερική, εμπορικές συμφωνίες πάλι, αλλά με κανονισμό. Ρήτρα διασφάλισης. Εσωτερικό θέμα δηλαδή, νομοθετική διαδικασία για μας. Η συγκητής μας είναι ο Γιώργ Λάιχτφριντ, στον οποίο και δίνω το λόγο. Έχεις το λόγο, Γιώργη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέμα στο δυνατόν πιο σύντομο. Συνήθω, οι συνάδελφοι όταν ξεκινάνε έτσι μακρηγορούν μάλλον. Σας διαβεβαιώ ότι δεν θα σας κρατήσω. Έχω πει στους συναδέλφου ό,τι είχα να του πω στην προηγούμενη συνάντηση και του. Πράγματι δεν μένει, δεν μένει τίποτα πια να πω. Ε, σε τι θα επικεντρωθώ λοιπόν. Θα ήθελα να πω ότι πρέπει να αναζητήσουμε προστασία κυρίως για τους παραγωγούς μας στις ε, πλέον απομακρυσμένες περιοχές όπως προσπάθησα να υποδείξω διακριτικά και σε σχέση με τις ε, προτάσεις της Επιτροπής Γεωργίας προσπαθώ να ενισχύσω τη θέση του Κοινοβουλίου και να υποχρώσω ταυτόχρονα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την έκθεσή μου να μας ενημερώνει πιο τακτικά για τα τεκτενόμενα και να παρακολουθεί πιο εντατικά τις προτάσεις. Αυτό είναι λοιπόν το νόημα των προτάσεων που νομίζω ότι είναι και σύμφωνο με το πνεύμα της συμφωνίας. Προσπαθούμε να διαφυλάξουμε και τα ε, συμφέροντα των επιχειρηματιών, των επιχειρήσεων αλλά και των εργαζομένων που δεν πάνε πάντα χέρι-χέρι. Μόνο. Και προσπαθούμε βέβαια και να προστατεύσουμε τα συμφέροντα όλων των εμπλεκομένων στη συμφωνία. Προσπαθώ να συμπεριλάβω κάποιες πτυχές, ε, μικρότερες επιχειρήσεις, επιχειρήσεις, γεωργοί που ασχολούνται ιδιαίτερα με τα βιολογικά προϊόντα, με το θεμητό εμπόριο και προσπαθώ ιδιαίτερα να αναφερθώ στο θέμα της κατανάλωσης ύδατος. Υπάρχει, αν πατώ με ψήφισμα ή πιο δεσμευτικό κείμενο των Ηνωμένων Εθνών και θα προσπαθήσω να το ενσωματώσω στην ε, ρήτρα διασφάλιση, διότι είναι, πιστεύω, θέμα σημαντικό για την Κεντρική Αμερική. Για δε το τυπικό κομμάτι της εκθέσεως, χρονοδιάγραμμα για τις τροπολογίες 16 Απριλίου, εξέταση 25 ή 26, έγκριση στην Επιτροπή 29 ή 3 Μαΐου, ολομέλεια τον Ιούλιο. Αυτό σκοπεύουμε να κάνουμε και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Είμαι πολύ περίεργος λοιπόν εδώ και με περιέργεια περιμένω ακούσω τις προτάσεις των αγαπητών συναδέλφων. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργ. Υπάρχει κάποιος ο οποίος θα ήθελε να σχολιάσει. Εκπρόσωπο τη Κομισιόν, παρακαλώ, έχει το λόγο. Ο κύριο ε, Μούλε θα πάρει πρώτο το λόγο, κύριε Στέρντι. Ωραία. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, πράγματι θέλουμε να ε, μιλήσουμε δύο. Ο ένας θα μιλήσει για τις μπανάνες και τον πόρο και εγώ προσωπικά θα σας αναφέρω κάποια πιο γενικά σχόλια για αυτό τον κανονισμό και την έκθεση του κυρίου, κυρίου Λάιχτφριτ. Πρώτα απ' όλα θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον κύριο Λάιχτφριτ για την έκθεσή του, για το έργο το οποίο έχει επιτελέσει σχέση με το θέμα αυτό και θέλουμε επίσης να τονίσουμε την αρχή η οποία διέπει ουσιαστικά αυτήν την έκθεση, δηλαδή θα πρέπει ουσιαστικά ε, να ακολουθήσουμε αυτό το πλαίσιο. Πέντε κατηγορίες μπορούμε να διακρίνουμε σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες. Πρώτα απ' όλα για την επιτήρηση, την παρακολούθηση, την περισσότερη ενημέρωση από την Κομισιόν. Ήταν η πρώτη κατηγορία. κάποιε άλλες τροπολογίες αφορούν πιο κοινωνικά ζητήματα, δηλαδή δικαιώματα των εργαζομένων, ε, συνδίκες εργασίας κτλ. Ενώ υπάρχουν και κάποιες τροπολογίες ε, οι οποίες αναφέρονται στο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων. Μια άλλη κατηγορία τροπολογιών αφορά το μηχανισμό σταθεροποίησης για τις μπανάνες. Ο κύριος Λάχτφριτ, στην έκθεσή του επιδιώκει με το κορεάτικο μοντέλο την μεγαλύτερη δυνατή ομοιότητα. Όταν συζητήσαμε τον κανονισμό διασφάλισης ε, για την Κορέα υπήρξαν κάποια κοινωνικά ζητήματα και περιβαλλοντικά θέματα βέβαια, τα οποία ανέκυψαν. Οι τροπολογίες οι οποίες σχετίζονται με το κοινωνικό περιβαλλοντικά, εργασιακά ζητήματα. Με τη δήλωση Επιτροπής νομίζω ότι λαμβάνονται υπόψη. Μια αντίστοιχη λύση είδαμε σε ό,τι αφορά και το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ενεργοποίηση των ερευνών. Επίσης υπήρξε συνένεση ότι καμία τροπολογία δεν μπορεί να έρχεται σε αντίθεση με τις συμφωνίες στο πλαίσιο της Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου. Αν υπάρχουν διαφορές σε σχέση με τροπολογίες για το μηχανισμό σταθεροποίησης της μπανάνες, ο συνάδελφος κ. Γκλάχη θα σας πει τα σχετικά. Κάποιες τροπολογίες εφόσον εγκριθούν θα κάνουν πιο δύσκολο την αναζήτηση μέτρων διασφάλισης και σε σχέση με το κρατικό μοντέλο. Εμείς λοιπόν θα πρέπει να σταθμίσουμε τις επιπτώσεις που θα έχει μια τέτοια τροποποίηση. Μια τροποποίηση που, όπως είπα, δυσκολεύει περισσότερα τα πράγματα. Είναι, για παράδειγμα, τροπολογία 14 που ζητά από τη βιομηχανία που θέλει να μείνει ανοιχτή μια έρευνα, να παρέχει και πληροφορίες για τις συνθήκες εργασίας. Αυτό δεν ε, εντάσσεται κατά ανάγκη στο κρατικό μοντέλο. Άλλες τροπολογίες τώρα, αν εγκριθούν, θα επιβάλλουν μεγάλο διοικητικό άχθος, όχι μόνο και στην Κομισιόν, αλλά και στους οικονομικούς παράγοντες. Αυτό αφορά όλες ιδιαίτερες τροπολογίες που αφορούν κάποιες απαιτήσει αναφοράς και παρακολούθησης. Ορισμένα από τα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να αναφέρονται, να παρακολουθούνται, είναι στη δικασία της Κομισιόν, αλλά θα πρέπει σίγουρα και να επαληθεύονται. Οι πόροι μας λιγοστεύουν όλο και περισσότερο. Είναι μια επίπτωση λοιπόν που θα πρέπει να τη λάβει υπόψη η Επιτροπή σας. Δεν θα μακρηγορήσω αναφέροντας λεπτομέρειες, αλλά βέβαια είμαστε έτοιμοι να τις συζητήσουμε τις λεπτομέρειες αυτές. Ο κύριος Γκλάιφ τώρα, ο συνάδελφός μου, θα σας ε, σχολιάσει το θέμα του εμπορίου μπανάνας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Τα σχόλιά μου αφαιρούν ε, την ε, συμφωνία με το Περού και την Κολομβία. Θα πρέπει να υπενθυμίσω ότι ο μηχανισμός παντροπής μπανάνας είναι μια ειδικού είδους διασφάλιση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν υπάρχει αποσταθεροποίηση της αγοράς εξαιτίας μεγάλου αριθμού εισαγωγών, μεγάλου ποσοτήτων εισαγωγών. Πρόκειται για μηχανισμό ο οποίος είναι ευέλικτος, μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή γρήγορα, πολύ πιο γρήγορα από την διμερείς διασφαλίσεις και πρόκειται και υπάρχει και μηχανισμός προειδοποίησης και διάρκεια της περίοδου της μεταβοήτης. Σας εξήγησε ο συνάδελφος στην αρχή, από της συμφωνούμε, αυτό ο εφαρμοστικός κανόνας δεν μπορεί να είναι αντίθετο με τα κείμενα και τις δεσμεύσει που έχουμε αναλάβει στα πλαίσια των Συμφωνιών ελεύθερη Αγοράς. Διότι μια τέτοιου είδους διαφορά, και εδώ φοβούμαι ότι μια τέτοιου είδους διαφορά δημιουργείται από κάποιες τροπολογίες οι οποίες καθιστούν υποχρεωτική η αυτόματη τον ε, μηχανισμό σταθεροποίηση της μπανάνας. Αυτό είναι κάτι που δεν προβλέπεται στα FTAs και είναι σε αντίθεση με τις συμφωνίες που έχουμε συνάψει με τους εταίρους μας. Και κάτι τέτοιο δεν πρέπει να συμβεί. Επίση, κάποιε τροπολογίε με δημιουργούν δεύτερο πρόβλημα. Θα πρέπει να δεσμευθούμε στις, με τις παρούσες ε, συμφωνίες που έχουμε κάνει στα πλαίσια των συμφωνιών στη Γενέβη και με τη ΣΥΠΑ τα θέματα τα δεσμολογικά επίθεσης θα πρέπει να τα σεβαστούμε και υπάρχει και η αυτόματη διασφάλιση που προσφέρουν κάποιες ε, ε τροπολογίες οι οποίες αφορούν κάποια αυτόματες ποσοστώσεις. Κάνω λοιπόν έκκληση σε εσά. Θα πρέπει να μην προτείνουμε τροπολογίες οι οποίες δεν συνάδουν με τις συμφωνίες που έχουμε ε, ε, υπογράψει όσον αφορά τις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών, κυρίως αυτές που αφορούν τις ποσοστώσεις στον τομέα των μπανανών. Η... Ξέρουμε ότι είναι ευαίσθητο προϊόν η μπανάνα, το έχουμε πλήρως λάβει υπόψη, αλλά δεν μπορεί να υπάρξει πύλης ε, απελευθέρωση. Προβλέπονται το 2020 κάποιοι μηχανισμοί για να μπορέσουμε να έχουμε μια κατάσταση σταθερότητας μέχρι τότε. Και τελευταία παρατήρηση κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν κάποιες άλλες τροπολογίες που υποδεικνύουν κάποιο νομισματικό αντιστάθμισμα για τους παραγωγούς, όπως προβλέπεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, στα πλαίσια των δεσμεσεών μας στο FTA. Θα πρέπει επίσης να υπενθυμίσω και εδώ ότι το αντιστάθμισμα για τους Ευρωπαίους μπανανοπαραγωγούς συμπεριλαμβάνονται στην ε, ε, κοινή οργάνωση αγοράς μπανάνων στα πλαίσια της συμφωνίας το 2006. Και αυτό είναι κάτι το οποίο λαμβάνεται υπόψη σε όλες τις προσεχείς συμφωνίες, άρα δεν μπορεί κανείς να σκεφτεί ότι θα δικαιολογήσει περαιτέρω την καταβολή κάποιων ποσών στους Ευρωπαίους μπανανοπαραγωγούς πέραν αυτών που προβλέπονται σε αυτή τη συμφωνία που προανέφερα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ερωτήσω το εξής. Στο άρθρο 10 των διασφαλίσεων συμπεριλαμβάνει η Επιτροπή στο κείμενο το ότι αν έχουμε να κάνουμε με μεγάλη επιδείνωση κατάστασης αλλάζουν τα πράγματα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο προβλέπει και σε κάποιες ε, τροπολογίες ο εισηγητής. Ποιος είναι ο ορισμός αυτής της μεγάλης επιδείνωσης, σοβαρής επιδείνωσης αν θέλετε να κάνετε. Αυτές ε, ε, μιλάτε για σοβαρούς τραυματισμούς, serious injury. Αυτό είναι κάτι που αφορά μια έννοια πολύ σαφή. Με... Και με την ευρεία και με τη στενή έννοια του όρου. Μπορεί κανείς να καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Πρόκειται Λοιπόν, από τη μία λέμε injury, τραυματισμός, από την άλλη serious deterioration σοβαρή επιδείνωση. Πρόκειται για όρους με διαφορετική έννοια. Το serious deterioration δεν είναι τόσο αυστηρό όταν πρόκειται για μία ζημία όπως ο τραυματισμός. Θέλουμε λοιπόν να δώσουμε μια κάποια ευελιξία σε αυτούς τους όρους. Ο εισηγητής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλύτερος ορισμός. Ναι, θα συμφωνήσω με τον εκπρόσωπο της Επιτροπής. Ασφαλώς και έχει δίκιο σε αυτό. Ευχαριστώ και για τις υποδείξεις. Θα προκύψουν φυσικά κάποιες τροπολογίες όταν δούμε πιο ξεκάθαρη εικόνα για το τι χρειάζεται να κάνουμε και τι όχι. Από αυτά που έθιξε η Επιτροπή πιο συγκεκριμένα, καταρχάς οι συνθήκες απασχόλησης βεβαίως, το να εξετάσουμε τις συνθήκες απασχόλησης είναι σημαντικό πιστεύω και είναι σημαντικό και για τους ανθρώπους που πρέπει να εργαστούν στον κλάδο αυτόν. και για να αντιλαμβάνονται τι τους προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι προσθεμένη αξία φέρνει η προσθεμένη αξία. Για δε την μπανάνα συγκεκριμένα. Αντιλαμβάνομαι ότι η Επιτροπή ίσως να μην είναι πολύ ικανοποιημένη με κάποιες από τις τροπολογίες. Να τα συζητήσουμε αν θέλετε. Αλλά δεν μου αρέσει η έκφραση. Δεν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Εάν εμείς το αποφασίσουμε, κυρία Επιτροπή, θα συμβεί. Γι' αυτό λοιπόν καλό θα ήταν να δούμε, να συζητήσουμε τι επιπτώσεις μπορεί να έχει αν το αποφασίσουμε. Αλλά ως νομοθέτης την αρμοδιότητα για την απόφαση, εάν πρόκειται να συμβεί ή όχι, την έχουμε εμείς. Ευχαριστώ πολύ Γιώργ. Προθεσμία 16 Απριλίου, 12 το μεσημέρι. Και πάμε στο σημείο 32, Συμφωνία Εμπορίου, Σταθεροποίηση. Αντίτρα διασφάλιση μηχανισμού σταθεροποίηση τη πράγμα στο πλαίσιο τη Συμφωνία Ελευθερών Συναγών μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση, Κολομβία και Περού με τον Μπέρντ Λάγκε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Είναι, όπως ε, καταλαβαίνετε, πολύ σημαντικό αυτό το νομοθετικό ε, κείμενο, όπως άλλωστε και οι ε, ρήτρες διασφάλισης για την κεντρική Αμερική. Έχουμε την ίδια γραμμή με τον Γιώργ Λάιχτφριτ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταθέσει μια δέσμη μέτρων νομοθετικών αντίστοιχο με αυτό των προτάσεων για την Νότια Κορέα και αντίστοιχο με κάποιες από τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Άλλωστε και ο κύριος άλλο και εγώ είχαμε συμμετάσχει ε, στη σχετική διαπραγμάτευση, είχε υιοθετήσει. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να επισημάνω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν έχει αξιοποιήσει επαρκώς το πεδίο χειρισμών που της προσφέρεται. Υπάρχουν και άλλοι τομείς, φερρυπίν. Ιάννα, δεδομένης ή ενόψη μία μιας συμφωνίας διαφιλονικούμενης, πρέπει να πούμε, στην κοινωνία των πολιτών, είναι απαραίτητο να ενισχυθεί ο διάλογος με την κοινωνία των πολιτών. Και προτείνω ως εκ τούτου κατά την επιτήρηση των συνεπειών της συμφωνίας, των παρακολούσεων συμφωνιών της συμφωνίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να έχουμε οργανωμένο διάλογο με την κοινωνία των πολιτών. Και εδώ συνδέεται και ένα άλλο Δεύτερο σημείο, σε ποιο βαθμό η Επιτροπή μπορεί να δώσει υποδείξεις ή συστάσεις για τις έρευνες που θα διεξάγονται. Στη συμφωνία με την Νότια Κορέα είχαμε το, την έννοια του interested parties. Για κάθε ενδιαφερόμενο επιχείρηση συνδικαλιστική οργάνωση κτλ. που θα μπορούσαν να ζητήσουν μια σχετική έρευνα. Και εδώ νομίζω μπορούμε ξεκάθαρα να πούμε, για να είναι σαφέ, ότι και η κοινωνία των πολιτών έχει ένα συμφέρον να παρακολουθήσει μια τέτοια εξέλιξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ως εκ τούτου μπορεί να ζητήσει την εξαγωγή έρευνα. Και επίσης εδώ συνδέεται ένα τρίτο σημείο αν μπορεί να λάβει δράση το Κοινοβούλιο. Το συζητήσαμε και πάλι με την ευκαιρία της Νότιας Κορέας και πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο και πάλι θα μείνει σε επαγρύπνηση και θα πει ότι παραμένει ως νομοθέτης στην επιτήρηση αυτών των θεμάτων. Τα κριτήρια τώρα, τέταρτο σημείο. Τα συζήτησαμε και τον κύριο Λάιχτφριτ τα ζητήματα δηλαδή κοινωνικών ε, συνθήκων εργασιακών, συνθήκων που είναι πολύ σημαντικά για την, για την αξιολόγηση και τη λήψη αποφάσεων, δύναμη του άρθρου 4. Πέμπτο σημείο που σε σχέση με την ε, Νότια Κορέα το έχουμε λησμονήσει, είναι η ετήσια έκθεση. Και εδώ περιμένουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί είναι καλό να γνωρίζουμε τι τελικά προκύπτει, τι υλοποιείται μέσα από τη συμφωνία, τι κάνει η Επιτροπή, πώς ελέγχει αν τηρήθηκαν ε, οι συνθήκες, οι προϋποθέσεις της ε, ε, συμφωνίας με την Νότια Κορέα, γιατί την πρώτη έκθεση θα την καταθέσει για την Νότια Κορέα τον Ιούλιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άρα θα δώσει και μια ε, σειρά από προτάσεις για περαιτέρω δράση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ίσως απλώς να λησμόνησε λοιπόν να συμπεριλάβει την πρόβλεψη για έκθεση Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξού και εγώ προτείνω την τροπολογία υπαριθμών 18. Και τελευταίο σημείο για την μπανάνα, γιατί το είχαμε συζητήσει. Οι τροπολογίες μου νομίζω δεν έχουν ε, προβλέψει αυτοματισμούς. Άρα δεν βλέπω εδώ πρόβλημα συμβατότητας. Απλώς θα ήθελα ο έλεγχος, η παρακολούθηση, ο μηχανισμός επιτήρησης να εισαχθούν μέσα στο σύστημα, έχοντας όμως και μια ερώτηση. την οποία βλέπουμε στην τροπολογία 24, μια και θα περάσει δύο χρόνια. Ερώτηση που έχει να κάνει με τις ποσοστώσεις για την εισαγωγή των μέτρων στο τομέα της μπανάνας. Εάν δεν αλλάζουν τα αριθμητικά στοιχεία, δεν θα πρέπει να αλλάξουν ε, οι προτάσεις σχέση με αυτά που ισχύουν πριν από δύο χρόνια. Δεν πρέπει να καταργηθούν. Εξού και προτείνω την ανθρωπολογία 24, για να ε, προσαρμοστώ μάλλον στην νομοθεσία και όχι στις ρυθμίσεις που βασίζονται στις ποσοστώσεις. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει κανείς να κάνει σχόλιο. Σκιώδης, ο κύριος Σάλμπα, η κυρία Χέλμετ. Όχι, ο Σάλμπα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σε ευχαριστούμε, συνάδελφε, για την δουλειά που έκανες πάει προς τη σωστή κατεύθυνση. Τώρα όσον αφορά το μηχανισμό της μπανάνα και οι δύο εκθέσεις νομίζω ότι περιέχουν τις ε, ε, προτάσεις που έκανε που υπάρχουν στην έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και αναφέρουν τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν καθώς και αυτά τα οποία προβλέπει ε, το σχετικό άρθρο για την ε, αλλαγή καθιστώτηση τις μπανάνες. Αυτά το προβλέπουν κάποιες τροπολογίες. Ο, ο κύριος Λάγκε προτείνει κάποια ε, αλλαγή όσον αφορά τον μηχανισμό της επιτήρηση την μπανάνα. Νομίζω ότι είναι κάπως αντιβατική, αλλά εν πάση περιπτώσει. Όσον αφορά τα πιο φιλεγόμενα μέρη, αφορούν τις ε, μπανάνες που αφορούν την ε, ρήτρα διασφάλισης. Η ρήτρα διασφάλισης δεν νομίζω ότι σωστά βρίσκεται εδώ πέρα. Θα πρέπει μάλλον να αναφερθεί, όπως αναφέρθηκε στον τρίτο, μηχανισμός διετησίας. Υπάρχουν επίσης, τώρα Κώστη, εγώ κάνω μία αξιολόγηση και των δύο συμφωνιών. Δεν ξέρω ε, αν επιτρέπεται, δεδομένου ότι τα συζητούμε από κοινού. Γι' αυτό αναφέρομαι στις δύο αυτούς τους μηχανισμούς Διασφάλειας. Υπάρχει η τροπολογία 5, Κολομβία, Περού, που αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα κοινωνικά και τα εργασιακά, καθώς και τα περιβαλλοντικά θέματα. Νομίζω ότι εδώ δεν είναι ο κατάλληλος ε, τόπος να συζητήσουμε αυτά τα θέματα, δεδομένου ότι, όπως είπαμε προηγουμένως, προβλέπεται και ειδική, ρήματα, ειδική ρήτρα συγγνώμη, για το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το θέμα αυτό θα πρέπει να το ξανασυζητήσουμε. Επίσης, υπάρχουν κάποιες άλλες τροπολογίες που ζητούν στην ετήσια έκθεση της Επιτροπή να μας δώσει κάποιες πληροφορίες όσον αφορά τα βιολογικά προϊόντα, την κατανάλωση και τις ε, σε εμπορικές ροές του δικαίου εμπορίου. Δύσκολα μπορεί κανεί να το αιτιολογήσει, αλλά εν πάση περιπτώσει είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο, όπως πάντα. Όσον αφορά τη διεύρυνση, του, την επέκταση του όρου ενδιαφερόμενα μέρη, υπάρχει ο ορισμός της Επιτροπής, ο ορισμός είναι επαρκής. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται τώρα να κάνουμε απαρίθμηση ε, όλων αυτών των ορισμών στη ρήτρα. Όσον αφορά τα ναι, επιτήρηση. Γίνεται λόγος για τους εμπορικούς μας εταίρους, για τους εργάτες και η ρήτρα διασφάλισης δεν ασχολείται με τέτοιου είδους θέματα. Νομίζω ότι το θέμα αυτό θα πρέπει να αναφέρεται στις διατάξεις όσον αφορά την ίδια τη συμφωνία. Ε, μέσα στις απαιτήσει για την επιτήρηση γίνεται λόγος και για τις συνθήκες εργασίας. Νομίζω ότι αυτό είναι αντιπαραγωγικό και δυσκολεύει την κατάσταση για αυτόν ο οποίος θέλει να υποβάλει αίτημα και ακόμη και για τις ίδιες υπηρεσίες της Επιτροπής είναι δύσκολο διότι είναι θα είναι υποχρεωμένος να αναλύσουν το θέμα αυτό και να το αιτιολογήσουν ε, στην έκθεσή τους. Έτσι δυσκολεύει ακόμη περισσότερο η όλη διαδικασία διερεύνησης και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν δίδει ευελιξία στην Επιτροπή τη στιγμή την οποία θέλει να κάνει κάποιες έρευνες για κάποια θέματα. Νομίζω ότι το θέμα αυτό μας οδηγεί ίσως σε αντίθετη κατεύθυνση. Ενώ εμείς θέλουμε οι διαδικασίες να είναι ταχείες και ευέλικτες και αν δημιουργηθεί πρόβλημα να μπορεί να τεθεί όλος ο μηχανισμός με όλες αυτές τις ρήτρε σε ε, λειτουργία με τρόπο σωστό. Επίσης εδώ αναφέρεται ότι θα πρέπει να παρουσιάζονται διάφορε προφορίες για την απασχόληση. Ε, ενδεχομένως θα μπορούσε κανείς να προσθέσει για το θέμα αυτό και μία νέα παράγραφος νεοτολογική σκέψη. Χωρίς να παρακολουθήσω περισσότερο, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εισηγητές για την εργασία που επιτέλεσαν. Είμαστε ούτως ή άλλως ανοιχτοί σε διάλογο, για αν υπάρχουν διαφορές μέσω διαλόγου μπορούμε να τις ξεπεράσουμε, να τις επιλύσουμε. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Σούλτς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τους συζητητές για τον τρόπο με τον οποίο συνεργαστήκαμε, με θετικό τρόπο. Και θα ήθελα να κάνω μία παρατήρηση σε σχέση και με τις δύο συμφωνίες, Κεντρικής Αμερικής και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχω την εντύπωση ότι ίσως θα έπρεπε εδώ να συμπεριλάβουμε συγκεκριμένες και ακριβείς ε, προτάσεις για τον ε, επιτήρηση και την τήρηση κυρίως των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μετά από την ακρόαση που είχαμε τώρα επί δύο ώρες. Διότι ενδεχομένως κάτι θα πρέπει να κάνουμε για να έχουμε πολύ θετική συνεισφορά εμείς από τη μεριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να καθησυχάσουμε τους φόβους κάποιον και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Αυτό ίσως θα μας βοηθήσει να ε, προσθέσουμε και ένα νέο στοιχείο επιτυχίας για όλους αυτών των συμφωνιών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα, όπως και με την προηγούμενη έκθεση, μπορείτε να μας εξηγήσετε τις ποσοστώσεις. Πριν είχαμε τα πάντα πριν όπλων, μετά είχαμε τη ζάχαρη, τώρα έχουμε την μπανάνα. Έχουμε ανοίξει πόλεμο. Μήπως είναι μη δασμολογική φραγμή. Μήπως κινδυνεύουμε να πούμε σε μια κατάσταση κατά την οποία θα μας παραπέμψει ε, σε δίκη ο ΠΟΕ ή δεν πειράζει επειδή είναι διμερή συμφωνία. Πρόεδρε, ευχαριστώ για την ερώτηση. Πολύ απλά να σας το εξηγήσω. Έχουμε δεσμευτική πολυμερή δεσμεύση από τον ΠΟΕ να ε, εγκαταλείψουμε τις ποσοστώσεις για την μπανάνα και να προχωρήσουμε σε καθεστώς μόνο δασμολογικό. Οι ε, τροπολογίες που θα καταστήσουν υποχρεωτική και αυτόματη την εισαγωγή διασφαλιστικής δικλίδας και αύξηση του ε, δασμού για την μπανάνα άπαξ και φτάσουμε σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο είναι μη δεσμολογικός φραγμός και άρα παράνομη για την ΠΟΕ και ω εκ τούτου είτε διμερό σχέση με τι ε, απευθεία δεσμεύσει από του εταίρου μα σε επίπεδο ΠΟΕ, θα συνεπάγεται πολύ σημαντικά νομικά προβλήματα και δυσκολίε. Χωρίς μικρόφωνο, κύριο Στόρτζη. Κύριος Ντέιβιτς. παρακαλώ. Νταβίτ, μάλλον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα όπως λέγεται να κάνω κάτι κι εγώ για τη δική μου χώρα κατά κάποιον τρόπο για το θέμα της μπανάνας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την συνάδελφο Λάγκε για την εργασία που έκανε στον τομέα αυτό, που αποδεικνύει ότι όχι μόνο ξέρει την κατάσταση, αλλά όλα αυτά τα θέματα με τα, τα οποία πραγματεύεται τα παρακολουθεί με μεγάλο πάθος. Όπως ελέγχθη προηγουμένως και από τον συνάδελφο, πιστεύω ότι κάποιες από τις παραγράφους της έκθεσής του, τις οποίες εξέτασα, δεν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στις ρήτρες διασφάλισης, αλλά στην, ε, στον κορμόν θέλετε της ίδιας της εμπορικής ε, συμφωνίας. Αυτό το monitoring, αυτό το, το άλλο θέμα της προστασίας των πέντε δικαιωμάτων νομίζω ότι εάν υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να γίνει, αυτό θα είναι. Επίσης, όπως είπε και ο κύριος Σούλτς, πιστεύω και εγώ ότι για τα ανθρώπινα δικαιώματα, επειδή υπάρχει ειδικό κεφάλαιο, εκεί θα πρέπει να αναφέρονται ειδικά. Το υπενθύμησε και ο συνάδελφος ε, ε, Σούλτς και είναι κάτι το οποίο και εγώ στη δική μου την έκθεση θα το συμπεριλάβω. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, πρέπει να πω ότι αισθάνομαι <laughs> απογοήτευση που δεν είπε τίποτα η Επιτροπή. Θα πρέπει να το συζητήσουμε δήμερος για την αηφορία καταρχάς αγαπητοί συνάδελφοι. Σε αυτή τη ασφαλιστική έκθεση, έκθεση δηλαδή για τη ρήτρα διασφάλισης, αυτό μας ενδιαφέρει περισσότερο και μόνο είναι εάν μέσα από το κεφάλαιο περί αφορίας μπορούμε να έχουμε συνέπειες έξω από το εμπόριο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή προσπαθούμε να κρίνουμε το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στην Κολομβία ή όπου αλλού, αλλά εάν μπορεί να έχει συνέπειες ως προς τις εμπορικές σχέσεις και εάν μπορούμε σε αυτές να εφαρμόσουμε τη σφαλιστική δικλίδα. Αυτά. Στα λοιπά, η έκθεση του κύριου Νταβίτ. Μπορούμε βεβαίως να τη συζητήσουμε, αλλά θα πρέπει και να δούμε εάν Φερρυπίν θα εισρεύσει μαζική παραγωγή άνθρακα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα έχει και χαρακτήρα dumping. Ε, ως εκ τούτου προτείνουμε συμπληρωματικά κριτήρια, τα οποία μας μπορούμε και διμερώς να συζητήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Μπέρντ. Προθεσμία 6 Απριλίου 2012. Εμπορική συμφωνία με Κολομβία και Περού με 33 της διάταξης. Ο Μάριο Ντάβιντε. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι εδώ που λέει η πρώτη ανταλλαγή απόψεων, ε, δεν ξέρω αν θα θυμάστε όμως κύριε Πρόεδρε, ότι προβλεπόταν να έχουμε μια αναφορά από τη London School of Economics για αυτό το θέμα. Δεν είχε γίνει την προηγούμενη φορά και είχαμε πει ότι θα προσπαθούσαμε να φροντίσουμε να γίνει αυτή τη φορά για να έχουμε κάποια σχόλια του LSE για το σημαντικό αυτό θέμα. Έχουμε τη μελέτη, τη λάβαμε, είναι πλήρη. θέλουμε να ευχαριστήσουμε το LSE. Εγώ προσωπικά Έχω στην προηγούμενη ανταλλαγή απόψεων καλύψει τα περισσότερα από αυτά τα οποία ήθελα να πω. Όλοι γνωρίζουμε ότι είναι ένα άκρος πολιτικό ζήτημα κυρίως και ότι τα περισσότερα κεφάλαια σε ό,τι αφορά το εμπόριο δεν δημιουργούν και τόσα προβλήματα όσο κατά το παρελθόν ή με άλλες συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών. Έχουμε βέβαια τα ζητήματα με τα κοινωνικά δικαιώματα, ανθρώπινα δικαιώματα, εργασιακά δικαιώματα, βιώσιμη ανάπτυξη και ούτω καθεξής. Έχω σκοπό σε όλα αυτά να αναφερθώ. Ένα άλλο σημείο που πρέπει να το επισημάνουμε και πριν ε, τη δική μου έκθεση, γιατί εσύ ξέρεις πολύ καλύτερα από όλους μας εδώ στην αίθουσα, ε, θα κατατεθεί μια προφορική ερώτηση στην Ολομέλεια και πρέπει να φροντίσουμε τα επόμενα χρόνια να εξασφαλιστεί η παρακολούθηση και να έχουμε πει και δηλώσει τι θέλουμε να παρακολουθεί η Κομισιόν, άπαξ και άρχισε να ισχύει η συμφωνία αυτή αλλάζει η κατάσταση. Στις χώρες έχουμε ένα ειδικό πρόγραμμα προστασίας, 120 εκατομμύρια δολάρια είναι το ποσό. Με μεγάλη επιτυχία λειτουργεί, αν και μπορούμε να εκφράσουμε τη λύπη μας για κάποια προβλήματα. Αλλά κανένας ε, στο πρόγραμμα δεν δολοφονήθηκε από τότε που άσχησε να ισχύει ό,τι και αν ήταν αυτός, δήμαρχος, ακτιβιστής, δημοσιογράφος κτλ. Και αυτό είναι επιτυχία. Ο κύριος Σόλς και άλλοι είχαν οργανώσει μια ακρόαση όπου ακούστηκαν διάφορα στοιχεία, αναγνωρίστηκε η πρόοδος. Από τότε που έχει αναλάβει τα ενία της χώρας ο πρόεδρος Σάντος ε, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Θα σας παρακαλώ να διαβάσετε και την έκθεση του Human Rights Watch, την οποία θα αναφέρω και στην ε, έκθεσή μου και ένα έγγραφο από το Κογκρέας των ΗΠΑ. Ξέρετε ότι η Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών μεταξύ Κολομβίας στην προκειμένη περίπτωση και ΗΠΑ θα τεθεί σε ισχύ τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους. Και αυτό θα συμπέσει λίγο πολύ με την ψηφοφορία που θα έχουμε εμείς στην Ολομέλη για το θέμα αυτό. Αλλά δύο σημεία για να τελειώνω. Το πρώτο είναι να δοθεί έμφαση και θα δώσουμε έμφαση στην ε, έκθεσή μας σε ένα νέο νόμο που θέλουμε να ενισχυθεί. And, ε, to inform the house of... Restitution law και στην τελευταία συνεδρία των ε, πρέσβεων ε, του Κορεπέρ δηλαδή, ε, από τον αρμόδιο για το εμπόριο αντιπροσώπων, ε, δόθηκε το πράσινο φως για υπογραφή από τα κράτη-μέλη. 14 με 28 Μαΐου θα γίνει αυτό. Στο Κορεπέρ διάφορα συμβούλια. Η υπογραφή από την Κομισιόν και τους, και τους δύο νέους εταίρους μας θα λάβει χώρα τον Ιούνιο, δηλαδή λίγο αργότερα από ό,τι αρχικά προβλεπόταν. Ίσως λοιπόν θα χρειαστεί να προτείνουμε και ένα διαφορετικό χρονοδιάγραμμα για την έκθεση αυτή. Και αυτό ακόμη και αν πιστεύουμε ότι θα μπορούσαμε παρόλα αυτά να ψηφίσουμε το Σεπτέμβριο στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ και συγγνώμη να μακρηγόρησα. Σας ευχαριστώ κύριε Ντάβιτ. Και προτείνω να ακούσουμε τη μελέτη του London School of Economics. και στα θέματα τα οικονομικά, αλλά και στις ε, αηφορίες τα ζητήματα. Την έχετε, αγαπητοί συνάδελφοι, όλη τη μελέτη. Ο κύριος Βούλκοκ. Κύριε Γούλκοκ, παρακαλώ να λάβετε το λόγο για να σας ακούσουμε. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Πάλι εδώ έχουμε μία συνολική ε, μελέτη, μια γενική μελέτη, στην οποία σας παρουσιάζω. Προσπαθούμε να επικεντρωθούμε στις ε, γενικές γραμμές, κυρίες γραμμές, γιατί δεν έχει κλείσει αυτή η έκθεση. Ε, πρώτα απ' όλα πρέπει να επισημάνω ότι δεν πρόκειται για μια συμφωνία κατά περιφέρεια, παρότι ήταν αρχικά ο στόχος αυτός της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Ε, το ότι δεν κατέστη δυνατό μάλλον οφείλεται σε διχοτομή, σε διχασμούς στο εσωτερικό της κοινότητας των Άνδεων και ιδιαίτερα μεταξύ Κολομβίας και Περού που τους οδήγησε χωριστά από την Βολιβία και το Εκουαδόρο να ε, συνάψουν σχέσεις εμπορικές με τους εταίρους. Η Βολιβία και το Εκουαδόρ είχαν την συμμαχία της Βολιβίας όπως ονομάζεται. Αν και από ό,τι φαίνεται τώρα ε, εξετάζει το ενδεχόμενο η Βολιβία και το Εκουαδόρ να ξανανοίξουν διαπραγματεύσεις. Δεν μπορεί λοιπόν να αναμένει κανείς να επιδεινωθεί η διχοτόμηση στην ε, κοινότητα των άντων, γιατί ήδη υπήρχε αυτή, άρα δεν επιδεινώνεται λόγω της συμφωνίας. Ε, οι οικονομικές συνέπειες δεν χρειάζεται να εκθέσω εξωδικότερα τις βλέπετε στην έκθεσή μας. Προσφέρει πάντως και ενισχύει την πρόσβαση για τις εξαγωγές Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα στην Κολομβία, όπου η δασμολογική προστασία ήταν υψηλότερη από αυτή της περίπτωσης του Περού σημαντικές αναμενόμενες, σημαντικά αναμενόμενα εφέλιο, προς την ενίσχυση του εμπορίου λόγω των δεσμεύσεων που αναλαμβάνουν η, Βολιβία και το, η Κολομβία και το Περού και που υπερβαίνουν τις άλλες του ΠΟΕ. Επίσης, είναι, σύμφωνη, σύμφωνη, είναι συμβατή με την ερμηνεία των κανόνων του ΠΟΕ και σε σχέση με τη Συμφωνία Κεντρικής Αμερικής για όσους ήταν πριν παρόντες. Η αγορά είναι σχετικά μικρή. 42η ως προς τις εξαγωγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, το Περού και 44η η Κολομβία. Αλλά στο σύνολο των εμπορικών συναλλαγών με την περιοχή. Φαντάζομαι ότι η ερμηνεία που θα δίνοντα μια συμφωνία είναι ότι είναι σύμφωνη με τις ε, ε, με τη φιλοδοξία για πρόσβαση στις αγορές αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δραστηριοποιείται σε περιοχή όπου ήδη υπάρχουν ανταγωνιστές ΗΠΑ, Καναδάς, αλλά και Κίνα, η οποία έχει συνάψει διμερή συμφωνία με το Περού. Και ενδιαφέρον θα είναι να δούμε και τις συμφωνίες της Κίνας η Συμφωνία της Κίνας είναι μια γενική συμφωνία, καλύπτει αγαθά υπηρεσίες ε, δικαιώματα ιδιοκτησία, ε, ιδιοκτησίας και γεωγραφικής προέλευσης, πρόσβαση, ε, επένδυση, προστασία επενδύσεων και ρήτρα μάλλον ευνομένου κράτου και ω εκ τούτου, εάν συνάψει αντίστοιχε συμφωνίε με άλλε χώρε Κεντρική Αμερική, τη Λατινική Αμερική η Κίνα, μάλλον αυτό θα έχει σημαντική συνεπίση στις πρόσβαση τη αγορέ ως προς την ισορροπία, δηλαδή ωφέλη για την Κολομβία και το Περού. Όπως είναι γνωστό, ήταν ήδη μηδενικέ οι δασμοί υπό το σύστημα κεντρικευμένων προτιμήσεων Plus, αλλά όπως και με την Κεντρική Αμερική θα προχωρήσουμε σε πρόσθετη απελευθέρωση στην μπανάνα και στο μίσο όπως η παραδείγματι το σταφύλι, το επιτραπέζιο σταφύλι, σταφύλι δηλαδή για, ε, ως φρούτο. Αλλά δεν αποκλείονται και άλλες αλλαγές στο σύστημα των σε σχέση μάλλον με το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων για το μέλλον. Οι δασμοί απελευθερώνονται σταδιακά και ο, κανένας δασμός δεν απελευθερώνεται με τη θέση σε σχέση της συμφωνίας. Προβλέπει όμως τη δυνατότητα και συνέχιση της απαγόρευσης ε, για τις τιμές στο χώρο των άνδεων ε, η συμφωνία σε ευαίσθητους τομείς όπως οι υπηρεσίες υγείας, κοινωνικές υπηρεσίες, ε, υπηρεσίες δημόσιου ωφέλους όπως διανομή νερού, δίκτυα νερού κτλ. Επιτρέπει παρεκκλήσεις. Υπάρχει επίσης μια επιφύλαξη όπως σε κάθε εμπορική συμφωνία ε, για την διαφύλαξη της ακαιρεότητας των χρηματοπιστωτικών αγορών των εμπλεκομένων κρατών. Προβλέπεται απελευθέρωση των κινήσεων κεφαλαίων αλλά με ρήτρα διαφύλαξης στο άρθρο 180 για ειδικέ συνθήκες και εν τέλει οριζόντιες παρεκκλήσεις, εξαιρέσεις μάλλον για την δυνατότητα οι χώρες αυτές να διατηρήσουν ή να εισαγάγουν μέτρα για λόγους προστασίας κοινωνικά μειονέκτουσων ομάδων, μειονεκτικών ομάδων ή εθνοτικών ομάδων. Καλύπτεται θέματα πραγματική διοκτησία λοιπόν, δημόσιων προμηθειών, ανταγωνισμού, κανόνες προελεύσεως όπως και με τη Συμφωνία της Κεντρικής Αμερικής. Προβλέπεται σωρευτική ε, διαγώνια σώρευση για όλη την περιφέρεια πνευματική ιδιοκτησία, θέμα διαφιλονικούμενο και που συστήθηκε πολύ αρχή των διαπραγματεύσεων, δεν προβλέπεται επέκταση, παράταση μάλλον της διάρκειας ζωής ε, διπλώματος ευρεσιτεχνίας, πέντε χρόνια για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, περισσότερο δηλαδή από ό,τι είχε προβλέψει η Ευρωπαϊκή Ένωση ιστορικό τη και πρόσβαση σε ουσιώδη φάρμακα δυνάμει και των θηλώσεων στόχα. στα ζητήματα των ανθρωπινών δικαιωμάτων και της ε, φοροανάπτυξης όπως και στην Κεντρική Αμερική. Έχουμε την ε, πάγια ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα με θετική υποχρέωση, δηλαδή δεν αποτελεί απλώς ε, μία ρήτρα που λέει ότι θα πρέπει το εμπλεκόμενο κράτος, η εμπλεκόμενη κυβέρνηση να εφαρμόσει κτλ. Πρέπει και να διασφαλίσει την εφαρμογή των δεσμεύσεων στο πλαίσιο της συμφωνίας μέσα στην δικαιοδοσία του, την επικράτειά του. Επίσης, ε, δεν υπάρχει, όπως στην περίπτωση και της ε, Κεντρικής Αμερικής, ειδικό όργανο παρακολούθηση. Την παρακολούθηση πρέπει να αναλάβει κάποιος άλλος δηλαδή. Η Επιτροπή Εμπορίου είναι αρμόδια σε σχέση με την ε, συμφωνία αυτή. Οι αρχές των δικαιωμάτων έχουν επίσης εφαρμογή και άρα μπορεί οποιοδήποτε μέτρο σε περίπτωση παραβίαση, μέρος σε περίπτωση παραβίασης να αναλάβει τα αρμόζοντα μέτρα, εξαρτάται βέβαια υπό ποιου όρου και ποια μέτρα θα ληφθούν. Μπορεί η συμφωνή γνώμη λοιπόν στην ε, συμφωνία αυτή να αποτελέσει ε, συγχωροχάρτη για παραβίαση ανθρώπινων δικαιώματα. Υπάρχει το ερώτημα αυτό φυσικά, αλλά από την άλλη υπάρχει και η απάντηση ότι μπορεί μια τέτοια συμφωνία να αποτελεί ουσιαστική πίεση για τη βελτίωση, την διατήρηση και ενίσχυση τη υφιστάμενη και ορατή πρόοδου στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Υπόθηκε όμω ήδη στην συζήτηση ότι το κύριο ζήτημα εδώ είναι πάνω απ' όλα η παρακολούθηση της διαδικασίας. Στις διατάξεις περί αηφόρου ανάπτυξης έχουμε σε ένα βαθμό σύμπτωση με τρίτρα ανθρωπινών δικαιωμάτων, όπως και στις βασικές συνθήκες του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, συμβάσεις του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Επίσης, παρακολούθηση από την Υποεπιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εμπορίου, που θα μπορούσε εν μέρη να αξιοποιηθεί για να ενισχυθούν οι πτυχές εκείνων των, εκείνες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν να κάνουν με τις ε, διαπραγματεύσεις για συμφωνίες ελεύθερου συμφωνίες συνθήσεις κτλ. Ε, Κλείνοντα, θα ήθελα να επισημάνω, σε σχέση με τις χώρες αυτές τη Λατινική Αμερικής, ότι η έγκριση του κειμένου είναι μόνο μια αρχή. Η υλοποίηση είναι το κύριο σημείο εδώ. Πρέπει δηλαδή πάνω απ' όλα να επαγνήσουμε για ουσιαστική υλοποίηση και ως προς τις πτυχές του εμπορίου και των επενδύσεων, αλλά και ως προς τις ανθρώπινες, τα δικαιώματα και τη ρήτρα για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Μας δώσατε μια εικόνα των συνεπειών αυτής της συμφωνίας και τα καλά της σημεία και τα πιο αδύναμα. Ας ακούσουμε τώρα τους συναδέλφους, ο κύριος David Martin, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα πολύ σύντομο σχόλιο προς τον εισηγητή. Να πω πρώτα απ' όλα ότι συμφωνώ με τα περισσότερα από όσα είπες και πολύ σωστά λες ότι υπάρχει τουλάχιστον στο χαρτί μια πολύ έντονη ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όπως μας έδειξε και παρόλα αυτά το London School of Economics, δεν υπάρχει όμως ε, ο μηχανισμός παρακολούθησης ε, της ρήτρα στη συμφωνία αυτή. Ίσως στο πλαίσιο της διαδικασίας σύμφωνης γνώμης θα πρέπει να καταρτήσουμε και ένα ψήφισμα που να λέμε ότι θα πρέπει πρώτα να έχουμε την κοινότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πριν την εφαρμογή και να είναι προηγούμενο να δημιουργούνται τέτοιες κοινότητες, ε, ακόμη και αν αυτό δεν το λέει η συμφωνία. Και ένα παράδειγμα είναι και η συμφωνία με το Μαρόκο. Ε, βέβαια και έγινε μετά την υπογραφή της συμφωνίας, αλλά νομίζω πρέπει να επιμείνουμε να γίνονται ταυτόχρονα αυτά τα δύο. Γιατί χρειαζόμαστε μια κοινότητα παρακολούθησης. Γιατί αν το αφήσουμε στα συνήθεια όργανα δεν υπάρχει καμία ε, συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην παρακολούθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δηλαδή ουσιαστικά οι εμπλεκόμενοι θα αποφασίζουν κατά πόσον παραβιάστηκαν ή δεν παραβιάστηκαν τα ανθρώπινα δικαιώματα και αυτό δεν είναι καλοδεχούμενο. Τώρα, αν δεν υπάρχει εφαρμογή, ε, τι να το κάνουμε. Ε, ξέρουμε από το GSP SIN, το, σύστημα, το γενικευμένο σύστημα των ε, προτιμήσεων, πρέπει να εφαρμόζονται οι διατάξεις. Για τα υπόλοιπα, σε ό,τι αφορά παραδείγματος το ελεύθερο εμπόριο, είμαι υπέρ. Ε, για το σκέλος που αφορά την Κολομβία, αν δεν πιστώ ότι θα υπάρξει βελτίωση ε, στην κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εγώ δεν θα τη στηρίξω. Ευχαριστώ. Κύριε this, this... Ευχαριστώ. Η εκθέση αυτή μας έχει κάνει όλους να χτυποκαρδίσουμε και να στενοχωρηθούμε. Υπήρξε πάρα πολύ μεγάλη άσκηση πιέσεων από ομάδες λόμπι και κυρίως από την κοινότητα των πολιτών. Από την Κολομβία, από περιβαλλοντικές ομάδες. Ακούστηκαν ε, ψηλόφωνα ή χαμηλές ή μικρές φωνές, αν θέλετε, ιδίως από την Κολομβία. Δεν ξέρω αν είμαι οι χαμηλές, οι μικρές φωνές αν θέλετε, ιδίως από την Κολομβία. Δεν ξέρω αν είμαι μόνη που το πιστεύω, αλλά νομίζω ότι ήταν πιο ισχυρές οι φωνές αυτές από αυτούς που ήταν υπέρ. Τουλάχιστον δεν ήρθε κανείς να χτυπήσει δική μου πόρτα από τους άλλους. Πρέπει να ξέρουμε ότι μπορούμε αυτό το κείμενο το εφαρμόσουμε. Πολύ σωστά είπε ο συνάδελφος David Μάρτιν. Αλλιώς τι να το κάνουμε να είναι καλό το κείμενο. Δεν έχει κάποιο νόημα. Αναφέραμε τη Συμφωνία Καναδά-Κολομβίας όπου γίνεται λόγος για την ελευθεροτυπία. Αν δεν υπάρχει ελευθεροτυπία, τότε τα ανθρώπινα δικαιώματα, επιβολή της νομοθεσίας, δεν γίνεται με τον σωστό τρόπο. Και δεν πρέπει να το δεχθούμε. Αυτό που με ανησυχεί πραγματικά είναι ότι ακόμη και αν έχουμε και την παρακολούθηση Χρειάζονται 27 χέρια να σκοθούν στο Συμβούλιο. Ένας μόνο από το Συμβούλιο που έχει μία εξορρυκτική βιομηχανία, έχει υπογράψει ένα συμβόλαιο κάπ κτλ. Ε, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να υψωθούν και τα 27 ε, χέρια για να σπάσει ε, το, η συμφωνία αυτή. Ανησυχώ ιδιαίτερος λοιπόν. Με πολύ χαρά άκουσα ότι υπάρχει αυτός ο μηχανισμός. Ότι μπορούμε με κάποιο τρόπο να προσθέσουμε ένα ψήφισμα σε αυτή τη ε, διαδικασία. Ίσως αυτό να είναι η απάντηση. Αλλά ανησυχώ. Έχω τεράστιες ανησυχίες. Ευχαριστώ πολύ. Ο Γιάν Ζαχράντιλ έχει το λόγο. Το πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την έκθεση αυτή. Νομίζω ότι ένα πολύ ενδιαφέρον μέρος έκθεση αυτής αρχίζει στη σελίδα 12, εκεί που γίνεται συγκριτική ανάλυση με άλλε συμφωνίε, όπως αυτή την οποία έχουμε με τη ΣΥΠΑ και τον Καναδά, με την Κίνα επίση. Εάν δει κανεί επιμέρου ε, κάποια χωριστά κομμάτια, μπορεί να βρει ότι, ότι αυτή η συμφωνία με το Περού και την Κολομβία σε σχέση με τις άλλες έχει ένα θετικό πρόσημο. Και σε κάποια σημεία, αν δείτε τα πιο σημαντικά κομμάτια της σε σχέση με τις άλλες ε, συμφωνίες που έχουν υπογραφεί, δίδεται η εντύπωση ότι έχει πολύ καλές ε, ε, δυνατότητες και μπορεί κανείς να συνενέσει σε αυτή την συμφωνία. Διότι όπως λέγω, αν εξετάσει τις άλλες, κάποιες από αυτές δεν είναι της ίδιας ποιότητας και οι στόχοι δεν είναι παρεμφερείς. Άρα ίσως αξίζει ε, να κάνουμε, να σταθούμε λίγο περισσότερο σε αυτού του είδους της συγκρίσεις. Ευχαριστώ, δεν ζητήκανε άλλο στο λόγο. Να δούμε. Πώ μπορούμε να προλάβουμε, μια και έχουμε ακόμα ένα σημαντικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Ε, αλλά ας δώσω και το λόγο στον εισηγητή. Thank you very much, uh, Chair. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το πρώτο σχόλιο που έγινε είναι ότι κάποιοι ε, λυπούνται διότι δεν πρόκειται για μια πρωτότυπη συμφωνία. Εγώ δεν συμφωνώ. Χαίρομαι διότι θα μόνο σε αυτό το στάδιο με τον Πέρο και την Κολομβία. Διότι βλέποντας τι συνέβη δηλαδή την ψηφοφορία με, το, με τη Βολιβία και το τι έγινε σε επίπεδο ΙΕ, δεν θέλω με αυτούς να συνάψουμε καμία συμφωνία. Τώρα, David, με ξέρεις εδώ και 20 χρόνια. Ξέρεις δεν είμαι μαζοχιστής. Και όταν ανέλαβα την έκθεση αυτή, πίστευα όντω ότι χρειαζόμαστε τέτοιου παρακολούθηση και το υποστηρίζω αυτό που λέγεται. Το πρόβλημά μου με το σχέδιο έκθεση που κυκλοφόρησε κυρίω στην ομάδα σου είναι ότι είχε κατατεθεί η προφορική ερώτηση. Εγώ συνυπέγραψα, αλλά στο ψήφισμα δεν αντικατοπτριζόταν το πνεύμα αυτό. Αλλά όσον αφορά την παρακολούθηση, όντω. και κυρίω τα θέματα που ανέφερε Και χαίρομαι που το έθεσε το θέμα αυτό, το σημείωσα και θα το εξετάσω. Έτσι έχουν τα πράγματα. Doubts at this stage. Όσον αφορά τις αμφιβολίες που εκφράστηκαν από τη συνάδελφο όλους όντως μας πλημμυρίζουν τα αιτήματα από την κοινωνία των πολιτών και από κάποιους που καταγγέλουν ότι όντως υπάρχουν πραγματικά προβλήματα. Κυρίως στην Κολομβία, αλλά και στο Περού. Δεν είναι αποκλειστικότητα της Κολομβίας το σύνολο των προβλημάτων που αναφέρονται. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να σας πω ότι πιστεύω ότι οι αντίστοιχες αρχές των δύο χωρών αυτών που προέρχονται από δύο διαφορετικά εντελώς μέρη του πολιτικού ε, φάσματος. Ε, ενεργούν καλή την πίστη. Και αν πρέπει εμείς να κάνουμε την παρακολούθηση, την εποπτεία από τη δική μας μεριά, στα πλαίσια του ΣΕΣ, φαντάζομαι ότι Και στις δύο αυτές ε, δημοκρατικές ε, χώρες αυτό σημαίνει μεταξύ άλλων ότι όντως πρόκειται για δημοκρατία, γιατί μπορεί όποιος δεν συμφωνεί να εκφράσει την αντίθεσή του και να διαμαρτυρηθεί. Άρα δεν νομίζω είναι και τόσο κακές. Στις 27 Απριλίου λοιπόν θα έχουμε το σχέδιο εκθέσεως. Παρακαλώ κύριε Βουλκοκ, το θέμα της ε, Γουλκοκ. Σύγκριση συμφωνίας με τη συμφωνία των Πολιτειών. Πολύ σύντομα όμως. Νομίζω ότι είχε να κάνει περισσότερο με διαφορές μεταξύ της προσέγγισης των Πολιτειών στις ε, συνθήκες εργασίας και το κοινωνικό περιβάλλον και τη συνέπεια αυτών στο εμπόριο. Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση πιο πολύ τίνει προς τις, την προαγωγή συμπεφωνημένων ε, συνθήκων εργασίας. Αυτή είναι η διαφορά. Η Κίνα βέβαια στις, στις συμφωνίες της δεν συμπεριλαμβάνει τίποτα για προδιαγραφές περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Καλώς ευχαριστώ. 27 Απριλίου θα ξαναδούμε το θέμα και τώρα στο επόμενο θέμα. Υπαριθμόν 34. Σίγμα δέλτα σίγμα αλφα. ΑΚΑΑ. Πολύ σημαντικό και ο κύριος Βιταλ θα λάβει το λόγο. Είμαι εξ officio εγώ εισηγητής του θέματος αυτού. Και ως... Παρακαλώ προσέξτε τι λέω. Ως επιβάλλουν οι κανόνες, περιμένω τη γνωμοδότηση της Επιτροπής για να συντάξω την έκθεσή μου. Αυτή τη φορά όμως δεν μπορούσα να το κάνω αυτό, διότι υπάρχει το χρονοδιάγραμμα και ήμουν υποχρεωμένος να παρουσιάσω ένα σχέδιο έκθεσης για την συνεδρίαση μας αυτή. Εγώ, λοιπόν, έφερα σε πέρα στις υποχρεώσεις που είχα, χωρίς να γνωρίζω στο τέλος Ποια θα είναι η άποψη που θα υπερισχύσει στην Επιτροπή μας. Σας υπενθυμίζω ότι είχαμε αποφασίσει να κάνουμε μια έκθεση, μια άσκηση ειδική, για να δούμε δηλαδή αν υπάρχει συνέπεια μεταξύ των εμπορικών μέτρων και του τι κάνουμε στα πλαίσια της εξωτερικής μας πολιτικής και δράσης με το Ισραήλ. Ακούσαμε τον Επίτροπο Ντεκούχ και ζητήσαμε και την γνωμοδότηση της ΑΦΕΤ. Στη συνεδρίαση με τον Επίτροπο δεν μπορέσαμε να καταλήξουμε σε οριστικά αποτελέσματα. Τον ακούσαμε και η αντίδραση Επιτροπής μας ήταν ε, πρέπει να πω αμφιλεγόμενη. Δηλαδή άλλοι ήταν υπέρ, άλλοι ήταν κατά. Πολλοί συνένεσαν, συμφώνησαν και πολλοί άλλοι ήταν υπέρ της αντίθετης άποψης. Άρα δεν μπορούσα να καταλάβω τελικά πώς διαμορφώθηκε η οριστική θέση Επιτροπής. Το ίδιο συνέβη και με τη γνωμοδότηση της ΑΦΕΤ. Δηλαδή ακόμη δεν έχουμε οριστική θέση γνωμοδότηση εκ μέρους της ΑΦΕΤ. Χρειάστηκε όμως εγώ να συντάξω το σχέδιο εκθεσής μου. Άρα αυτή την φορά δεν μπορούσα να πετριμένω τι θα κάνει η Επιτροπή μου και η δική μου η άποψη, η κρίση είναι αυτή που συμπεριλαμβάνεται στην έκθεσή μου. Εάν καταλήξει η Επιτροπή σε διαφορετικές απόψεις, εγώ θα αλλάξω την έκθεσή μου και όπως πάντα ό,τι κάνω θα το κάνω με στόχο να αντικατοπτρίστε η άποψη της Επιτροπής μας. Χθες αποφάσισαν οι συντονιστές να αλλάξουν το χρονοδιάγραμμα, γιατί πρόκειται για ευαίσθητο θέμα και η απόφασή μας για το φάκενο αυτό είναι να περιμένουμε τη γνωμοδότηση της ΑΦΕΤ. Τι σημαίνει αυτό. Ότι η ψήφιση της έκθεσής μου αναβάλλεται για αργότερα, μέχρι να έχουμε τη γνωμοδότηση της ΑΦΕΤ και αν χρειάζεται να αλλάξω και το περιεχόμενο του σχεδίου έκθεσής μου. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να ανοίξουμε συζήτηση για το σχέδιο έκθεσής μου, επειδή τα πράγματα έχουν έτσι. Αλλά αν νομίζετε ότι πρέπει να κάνουμε κάτι διαφορετικό, εσείς θα αποφασίσετε. ας αποφασίσει ο Προεδρεύων. Χρειάζεται να κάνουμε συζήτηση τώρα, μετά από την απόφαση που πήραν χθε οι συντονιστές. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, δύο συνάδελφοι στον το λόγο, δεν ξέρω. Χρειάζεται πολύ σύντομα, κύριε Σάκε και μετά η κυρία Λάτφορντ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κάποια τεχνικά ερωτήματα έχω για την πρόταση που μας έχετε υποβάλει. Όλοι αντιλαμβανόμαστε την κατάσταση στην οποία μας έχει οδηγήσει αυτή η απόφαση. Και θα ήθελα να τονίσω για μια ακόμη φορά ότι ως φιλελεύθερη πιστεύω ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι οικουμενικά και καταδικάζω στεναρά την παραγνώριση των δικαιωμάτων και τη ευημερία των Παλαιστινίων από του Ισραηλινούς και κυρίω ότι καταπατούν με του επικισμούς ε, και τις διεθνείς συμφωνίες, το διεθνέ δίκαιο. Η χώρα μου, η Ολλανδία, συνεχώ σπάει ε, την κοινή θέση για το ε, σε σχέση με το Ισραήλ και για αυτά τα θέματα. Τέλος πάντων, πολύ λυπηρό. Είναι πολιτικά αυτά τα ζητήματα και έχουν να κάνουν με τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο. Έχω μάλλον έχω ασχοληθεί με αυτό το θέμα, ε, το ΆΚΑ όπως το λέγαμε παλιότερα, ε, τη συμμόρφωση για την αποδοχή των προϊόντων ε, από τεχνικής πλευράς μέχρι τώρα, αλλά όχι πια. Δεν μιλάμε για μια τεχνική αναβάθμιση. Νομίζω ότι ουσιαστικά πρόκειται για πρωτόκολλο προς τη Συμφωνία Σύνδεσης. Λέτε βέβαια εσείς ότι ουσιαστικά πρόκειται για de facto ε, διεύρυνση, επέκταση των σχέσεων και θα δημιουργήσει ε, δυνατότητες πρόσβασης Ισραηλινών φαρμακευτικών και άλλων εταιριών ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει λοιπόν να δούμε, μπορούμε χωρίς ενδιάμεση έκθεση να αναστείλουμε τη σύμφωνη γνώμη. Τα, οι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που υπάρχουν σε εμπορικέ συμφωνίε συζητήσαμε την Κεντρική Αμερική διαμακρών σήμερα, αλλά τέτοιες ρήτρε έχουμε και σε συμφωνίες σύνδεσης, στη συμφωνία σύνδεσης με το Ισραήλ. Δεν είναι στα πρωτόκολλα, αλλά στη συνήθεια τη συμφωνία, το σώμα της συμφωνίας σύνδεσης. Εφαρμόζονται σωστά οι ρήτρε αυτές. Μήπως αυτό το μονοπάτι πρέπει να βαδίσουμε αν θέλουμε να ε, δώσουμε έμφαση σε αυτόν τον όρο. Στο σημείο F Συγματάφ δηλαδή, λέει, λαμβάνοντα υπόψη ότι για του ίδιου λόγου από το 2008 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αρνείται να δώσει την έγκρισή του για το πρωτόκολλο που αφορά τη συμμετοχή του Ισραήλ σε κοινοτικά προγράμματα. Από το 2009 όμω, νομίζω, όταν τέθηκε σε ισχύ στην δεκτή Σαββόνα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει έναν διαφορετικό ρόλο στην πλαίωση τη διαδικασία συμφωνή γνώμη. Πώ συνδέονται και συγκρίνονται αυτά τα δύο μεταξύ του, οι δύο έννοιε. Έγκριση, συμφωνή γνώμη δηλαδή. Τέλο, νομίζω ότι ο ρόλο μα είναι να αποφύγουμε την πόλωση, την περαιτέρω πόλωση και πρέπει να είμαστε επικοδομητικοί. Υπ' αυτήν την έννοια, νομίζω ότι πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη μα ω Κοινοβούλιο και θα έλεγα αντί να καθυστερήσουμε και να συνδέσουμε αυτό το θέμα σε μια συμφωνία ειρηνευτική, η οποία δεν αναφέρεται καν ως όρος, για την εμπορικές μας σχέσεις με το Ισραήλ. Νομίζω ότι αντιθέτως θα πρέπει ολοταχώς να δούμε τα θέματα ε, του ανθρω... των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου να τα θέσουμε στους Ισραηλινούς, αλλά να έχουμε στη θέση μας και τα κατάλληλα εργαλεία για να το πράξουμε. Και δεν είμαι βέβαιη ότι το πρωτόκολλο αυτό είναι και ένα τόσο καλό εργαλείο προς αυτή την κατεύθυνση. Ίσως όμως αν απαντήσεις σε τεχνικά μου ερωτήματα θα καταλάβω λίγο και τι ε, γίνεται με την καταλληλότητα αυτού του εργαλείου. Καλώ, ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συναδέλφοι, αλλά δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Καθένα λοιπόν ένα λεπτό για να μπορέσει και ο κύριο Μωρέρα να συμπληρώσει κάτι, κυρία Λάτσφορτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που μου δίνετε το λόγο, γιατί δεν είμαι μέλο τη Επιτροπή. Τακτικό. Ε, Όπω είπε και η κυρία Σάκε, πρέπει το Κοινοβούλιο να αναλάβει τι ευθύνε του είναι όντω, κατά την άλλη σημαντικό να ψηφίσουμε στην Ολομέλεια. Έχουμε καθυστερήσει αρκετά. Δύο χρόνια έχουμε καθυστερήσει. Και νομίζω ότι μόνο παρελκυστική πολιτική μπορεί να χαρακτηριστεί το να χρειαστούν άλλα δύο χρόνια για να εγκριθεί η συμφωνία. Δεν είναι δημοκρατικό λοιπόν και στην Κολομβία Περού είδαμε ότι υπάρχουν διαφορετικέ απόψει. Εν πάση α το πάμε το θέμα στην Ολομέλεια και να εκφράσει ο καθένα τι απόψει του με το ναι και με το όχι για να εγκρίνει εμεί. Κύριε Μωρέιρα, μιλήσατε για την ε, ε, αυτεπάγγελτη ανάληψη της έκθεσης από σας. Θα ήθελα να σε επισημάνω όμως, ότι δεν μπορεί να είναι μια θέση ισορροπημένη η καθυστέρηση της έγκρισης της εκθέσεως κατά δύο χρόνια. Χωρίς μικρόφωνο κύριε Λάτφουρτ. Πρέπει να σας διακόψω λέει ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ κύριε Ζαχράντιλ. Πρόεδρε πολύ σύντομα η ομάδα μας διαφωνεί με αδίποτε αναστολή, καθυστέρηση, γιατί πιστεύουμε όντως ότι είναι πολύ τεχνικής φύσης, εμπορικής φύσης η συμφωνία και δεν υπάρχει λόγος να επιμολυνθεί με υπερβολικές πολιτικές ε, σκέψεις. Παρακαλώ λοιπόν να μας ε, υποδείξετε μια ξεκαθαρή εικόνα για χρονοδιάγραμμα και γιατί ε, εάν είπαμε ότι μπορούμε να το δούμε μόνο μετά από την ε, γνωμοδότηση της ΑΦΕΤ, πρέπει να ρωτήσω κι εγώ τι συγκεκριμένα μπορούμε να περιμένουμε. David Martin. Πρόεδρε, δείξατε σολομόντια σοφία την κρίση σας προηγουμένως και πιστεύω ότι και εδώ θα το πράξετε. Είναι νομίζω ξεκάθαρο ότι το Ισραήλ παραβιάζει την ε, νομοθεσία Καλό θα ήταν λοιπόν να αποφύγουμε την απόρριψη, γιατί υπάρχει και αυτή η πιθανότητα, και άρα πρέπει να δώσουμε περιθώριο για συζήτηση. Γι' αυτό λέμε περισσότερο χρόνο. Στο υπαριθμό ένα όμως παράγραφο, εκεί που λέμε, ε, που, λέμε που γίνεται λόγος για ε, περίπτωση επιτυχούς ολοκλήρου της ρευτικής διαδικασία, καλύτερα θα ήταν να μην είμαστε τόσο ε, ρητοί και να αποφύγουμε την συλλογική κύρωση της Γάζας που επιβάλλεται από το Ισραήλ. Κύριο Σόλτς τελευταίος. όχι, όχι, εσείς εκεί. Um, uh, πάρα πολύ γρήγορα. Εγώ έχω εργαστεί εκ μέρου τη Βρετανική κυβέρνηση για την συμφωνία ειρήνευση με τη Βόρεια Ιρλανδία και τα έχω δει εκ των έσω. Το να ασκείται τέτοια πίεση δεν βοηθάει. Ίσως ε, κάποιες χώρες να κάνουν λάθη σε κάποια σημεία και πραγματικά και εγώ επικριτικά βλέπω κάποιες πρακτικές του Ισραήλ, αλλά αυτή η πίεση δεν βοηθάει τη διαδικασία. Αντίθετα, θα τους οδηγήσει να περιχαρακωθούν ακόμη περισσότερο, το είδαμε και στη Βόρεια Ιρλανδία. Και βγήκαν από τα χαρακώματα ε, πολύ αργά για να επικρατήσει τελικά η ειρηνευτική διαδικασία. Λοιπόν, ε, μην έχουμε το αντίθετο αποτέλεσμα. Ας προσπαθήσουμε να πετύχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε και όχι να καθυστερούμε. Και τώρα πια ο κύριο Σόλτ, τελευταίο. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θα μακρηγορήσω ούτε εγώ. Έχουμε ασχοληθεί και άλλη φορά με το θέμα. Και θα ήθελα να συμφωνήσω ρητά με τον εισηγητή ότι πρέπει να περιμένουμε τη γνωμοδότηση Επιτροπής των Εξωτερικών έχουμε άλλωστε συνεννοηθεί εδώ ότι πρόκειται για ένα θέμα με πολύ ξεκάθαρη πολιτική βαρύτητα. Τώρα, αν πρόκειται για, ε, πολιτι... για εμπορικές σχέσεις, για αναβάθμιση σχέσεων, ό,τι και να είναι, είναι δευτερεύον το θέμα σε σχέση με την πολιτική σημασία της συμφωνίας. Και γι' αυτό πρέπει και να ξεκαθαρίσουμε σε ποιο βαθμό και πώς θα αναλάβουμε δράση. Γι' αυτό λοιπόν θα ήταν καλό νομίζω να ε, περιμένουμε πρώτα την πολιτική εκτίμηση, την Επιτροπή των Εξωτερικών. Α, ναι, και ο κύριο Τέιλορ. Πρόεδρε, δεν συμφωνώ ότι είναι τεχνικό το ζήτημα. Ε, είναι ξεκάθαρα πολιτικό, το είπαμε, άλλωστε κάθε ένας από τους συναδέλφους πάνω στο θέμα της, ε, μετάφρα... της πολιτικής σημασίας του θέματος τοποθετήθηκε. Πιστεύω ότι θα πρέπει να προχωρήσει. Από την άλλη δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τις παραβιάσεις ε, του διεθνούς δικαίου. Πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι ε, επισημαίνουν ότι θα πρέπει να τιμωρηθεί το Ισραήλ για την ε, συμπεριφορά του κτλ. Και δεν μπορούμε να αφήσουμε κάθε περιθώριο δράσης στο Ισραήλ. Όταν αυτό συνεχίζει να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο δεν μπορούμε να αναβαθμίζουμε τις εμπορικές σχέσεις. Δεν μπορούμε να θάβουμε το κεφάλι μας στην άμμο και να ισχυριζόμαστε ότι δεν θα φέρει καμιά αλλαγή ή όποια θέση εγκρίνουμε ή απορρίψουμε. Ναι, κύριε. Πρόεδρε, ως και του ΕΛΚ θα ήθελα να πω δύο λόγια. Συμφωνώ πολύ με, τον, με τη συντονίστρια και τους άλλους συνάδελφους που έλαβαν τον λόγο προηγουμένα. Πρέπει να περιμένουμε τη γνωμοδότηση της ΑΦΕΤ. Η δε προθεσμία της ΑΦΕΤ είναι ξεκάθαρη. Ξέρουμε πότε θα ψηφίσει η ΑΦΕΤ τη γνωμοδότηση της τέλη Απριλίου και άρα νομίζω ότι είναι σαφέστατο το χρονοδιάγραμμα για την Επιτροπή μας. Και μπορούμε να προχωρήσουμε.